Μπορούμε να ξεκινήσουμε παρακαλώ γιατί δεν έχουμε και λίγα. Στην ημερήσια διάταξη η Μαρίτα δυστυχώς δεν μπόρεσε να παραστεί γιατί είναι σε μια άλλη συνεδρίαση στο εξωτερικό. Προτείνω να ξεκινήσουμε με την ημερήσια διάταξη. Μήνυμα από του διερμηνεί. Οι διερμηνεί σα ενημερώνουν ότι συνεχίζονται για τρίτη εβδομάδα κινητοποιήσει μα για τι συνθήκε εργασία, καθότι η δίκηση δεν έχει έρθει σε καμία επαφή μαζί μα για την επίλυση τη εργασιακή διένεξη. Επίση, έχουν επιταχθεί οι μεγάλε καμπίνε σε αυτή τη συνεδρίαση. Σα ενημερώνουμε ωστόσο ότι η συγκεκριμένη συνεδρίαση δεν θα επηρεαστεί από τι εν λόγω κινητοποιήσει. Σχέδιο μερίσια διάταξη. Πρέπει να πω ότι πολλέ ομάδε ήθελαν να φύγει να σημερινή για διάταξη για τι ψηφοφορίε. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε ξεκάθαροι, καλό είναι πριν ξεκινήσουν οι ψηφοφορίε ε, να δούμε πώ θα προχωρήσουν. Donc voilà pour euh, l'ordre du jour. Je sais pas s'il y a d'autres remarques. Non. Donc on peut. Euh... Έχουμε όλες τις ε, γλώσσες εκτός από βουλγαρικά, μαλτέζικα, κροατικά. Γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα ε, κίνημα, υπάρχουν κινητοποιήσεις από τους διερμηνείς ε, και στην προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής απασχόλησε εκφράσαμε την υποστήριξή μας ε, και το ενδιαφέρον μας στις κινητοποιήσεις και στη διένεξη και το μεσημέρι τόσο ή άλλως θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψε με τους διερμηνείς. Θέλω όμως να τους ευχαριστήσω από τώρα για το έργο τους. Σε ό,τι αφορά τις διοργανικές διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη, Είχαμε έναν τριμερή διάλογο για την αθεώρηση της οδηγίας για τα καρκινογόνα και μεταλλαξιογόνα χθε το βράδυ. Επικυρώσαμε τα σημεία τα οποία είχαν ρυθμιστεί σε επίπεδο τεχνικής ομάδας όμως ε, σε ό,τι αφορά ε, τα καυσαέρια από τους κινητήρες δίζελ ε, ήταν το θέμα που μας απασχόλησε σχεδόν σε όλη τη διάρκεια αυτού του τριμερούς διαλόγου. Ήταν σαφής η εντόλη του Κοινοβουλίου για να σας επενθυμίσω σε ό,τι αφορά το καθορισμό ενός ανώτατου ορίου και το παράρτημα 1-3, που δεν θέλω να επισέλθω τώρα εδώ σε λεπτομέρειες. Δεν καταφέραμε να προχωρήσουμε πέραν αυτού κατάσταση ε, παραμένει η ίδια, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, ε, οι συνομιλίες ε, και είμαστε και σε διαβλέψεις με την Βουλγαρική Προεδρία. Αυτά σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση οδηγίας για τα καρκινογόνα. Δεν ξέρω αν είναι εδώ ο εισηγητής για τα guidelines. Παρακαλώ, αν θέλετε να πάρετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις ε, εισηγητές. Ήταν ε, πολύ παραγωγικές οι εργασίες μας, εντατικές. Το ε, θέμα είναι οι guidelines κατευθύνες γραμμής για την απασχόληση. Η Βουλγαρική Προεδρία πραγματικά πήρε πρωτοβουλία στο Συμβούλιο για την εκθεσή μας και καταφέραμε από κοινού να κάνουμε ένα βήμα προς μια στενότερη συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την ε, εκπόνηση του τελικού εγγράφου. Στο μεταξύ, εγώ αλλά και η Γραμματεία ήρθαμε σε επαφή με SPC, MCO, Βουλγαρική Προεδρία και με το, την ομάδα εργασίας και την Κομισιόν θελήσαμε να υποστηρίξουν τις απόψεις μας και να ληφθούν υπόψη για την τελική απόφαση του Συμβουλίου. Βέβαια, μόνο διαβούλευση προβλέπεται. Βέβαια, υπήρξε άνοιγμα, γνήσιο άνοιγμα πλευρά ε, Συμβουλίου, των ε, υπεύθυνων για την προπαρασκευαστική εργασία και από την Κομισιόν. Στο τελικό κείμενο που ε, έλαβαν τα μέλη του Συμβουλίου από το Κρεπέρα αναφέρονται κάποια πράγματα που πιστεύω ότι θα δημιουργήσουν μια καλή πρακτική και ένα καλό προηγούμενο για το μέλλον. Την Πέμπτη αναμένεται να εγκριθούν αυτές οι κατευθυντές γραμμές 21 ε, Ιουνίου. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τι πετύχαμε. Ορισμένες προτάσεις μας ε, είναι στο τελικό κείμενο, όχι όλες ε, με την ισχυρή δίπλα που θα θέλαμε, όμως πάντα το βήμα που έγινε προς τα μπρος είναι σημαντικό. θα ήθελα να σας δώσω κάποιες πληροφορίες ε, στο τελικό κείμενο, τα πιο βασικά. Σημαντική τροπολογία για την ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Το τελικό κείμενο λέει ότι τα τρία θεσμικά όργανα, ιδίω ό,τι φάσει κατευθύνες γραμμές γραμμέ για τι πολιτικέ απασχόλησει των κρατών μελών, διατηρούν τη δέσμευσή του. Μιλάει πάρα πολύ γρήγορα ο μιλητής και δεν μπορεί να μεταφραστεί. Θα πρέπει να συνεχιστούν προσπάθειες που έχει ξεκινήσει η Βουλγαρική Προεδρία. Δεύτερον, η πρότασή μας ήταν στο 5-1. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητα. Ελήφθη υπόψη. Έξι. Για την εκπαίδευση προτάσει μα έχουν συμπεριληφθεί στο τελικό κείμενο. Η αρχή τη διαβίου μάθησης, ίσες ευκαιρίε για όλη την εκπαίδευση και η προσχολική εκπαίδευση και εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση κτλ. κτλ για τι ευκαιρίες στην αγορά εργασία. Επόμενο, 6, 5. Η διατύπωση για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φίλων. Πιο ισχυρή διατύπωση. Όχι όσο θα τη θέλαμε. Αλλά είναι ένα βήμα προ τα εμπρό και η σημασία τη ισορροπημένη προσοχή πνευματική ζωή που είναι στο κείμενο. Τέλο, το σημαντικότερο για μένα και το πιο δύσκολο. Συντάξεις. Το συστήσαμε διαμαρκρόν το θέμα με τους προσώπους Συμβουλίου και Επιτροπής και το αποτέλεσμα είναι ότι έγινε δεκτή πρότασή μας για τη συντάξη, στο τελικό κείμενο, ότι πρέπει δηλαδή να προσφέρω παρκές εισόδημα. Σε ό,τι αφορά το όριο συνταξιοδότηση, δεν συμπεριελήφθη η πρότασή μας και έχει αντικατασταθεί. Θα σας πω πως είναι στο τελικό ε, κείμενο. Πιθανή αύξηση του ορίου συνταξιοδότηση θα πρέπει να πλησιωθεί με στρατηγικές ε, για τον ε, ενεργό Σε Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για να σα ενημερώσω ότι θα έχουμε και κάποιου επισκέπτε, ε, περίπου 15 επισκέπτε που έχουν ε, προσκληθεί από την κυρία Μελάν. Επίση, ε, το απόγευμα θα έχουμε κάποιου προσκεκλημένου από τον κύριο Ντιντιέ τη Ένωση των Τυφλών και Αμβλιόπων από την Προβάνς και θα έχουμε και 20 επισκέπτες που έχουν κληθεί από την κυρία Μωρίν Σαρτιέ ε, στο τέλος της πρωινής συνεδρίασης. Αυτά ως ανακοινώσει ε, και σας προτείνω να περάσουμε στο σημείο 3 της ημερησής διάταξης ε, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολούμενους και για 5 λεπτά θα δώσω το λόγο στην κυρία Κάρλα Περέιρα που είναι τμήματάρχης ε, στην ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Απασχόλησης και Εξυγχρονισμού για την ε, Κοινωνική Προστασία. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επιτροπή για την ευκαιρία που με δίνετε να αναφερθώ σύντομα στις συστάσεις για την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία. Αυτή είναι η πρόταση της Κομισιόν που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του πακέτου ε, της κοινωνικής δικαιοσύνης το Μάρτιο του 2018. Ελπίζουμε ότι αποτελεί μια απάντηση σε κάποιες από τις ανησυχίες της Επιτροπής αυτής και του Κοινοβουλίου που αναφέρθηκαν στην έκθεση που προετοιμάσατε για τον ε, Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, όπου ως ε, θεσμικό όργανο υπογραμμίσατε τη σημασία του να επεκταθεί η κοινωνική προστασία και σύντομα νέες μορφές εργασίας. Η σύσταση αυτή λοιπόν είναι η πρόταση της Κομισιόν για να απαντήσει στις ανησυχίες αυτές μπορείτε να δείτε ότι η αδελφή πρωτοβουλία για την ε, οδηγία ε, που θα συζητήσετε αργότερα σήμερα τους διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή. Προκύπτει ω αποτέλεσμα μια διαδικασίας που υλοποιήσαμε πέρσι. Είχαμε διαβούλευση με τους κοινωνικού εταίρους σε δύο επίπεδα και είχαμε μια ανοιχτή δημόσια διαβούλευση πέρσι. Επομένως, αυτή η σύσταση ελπίζουμε ότι αντικατοπτρίζει και τις ανησυχίες των ενδιαφερομένων μερών που συζήτησαν μαζί μας. Ο στόχος της ε, σύστασης, η στόχη της σύστασης μάλλον, είναι δύο, για να τους συνοψίσω. Καταρχήν, καταρχήν να επεκταθεί η κοινωνική προστασία και σε όσους βρίσκονται στην αγορά εργασίας, αλλά λόγω των ε, σημερινών συμβάσεών τους δεν έχουν πρόσβαση σε κοινωνική προστασία, δηλαδή σε παροχές συνταξιοδοτικές, ε, σε άδεια ε, μητρότητας, πατρότητας, σε ταμείο ανεργίας κτλ. Και επίση ε, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι είναι βιώσιμα τα συστήματά μα κοινωνική προστασίας. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται ε, υπό αυτές τις νέες μορφές απασχόλησης και αν έχουμε όλο ένα και περισσότερους ανθρώπους που δεν συνεισφέρουν στα συστήματα κοινωνικής προστασίας ε, προφανώς διακυβεύεται η χρηματοδότηση του όλου συστήματος. Η σύσταση βασίζεται στο άρθρο 153 της Συνθήκης ε, και 352 έχοντας ε, κατά νου και τις απαιτήσει επικουρικότητας ε, που θέτει η συνθήκη, πιστεύουμε ότι η σύσταση ουσιαστικά αφήνει στα κράτη-μέλη να λάβουν τις ουσιαστικές αποφάσεις για το σχεδιασμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Επομένως, στη σύσταση δεν κάνουμε προτάσεις παραδείγματο χάρη για τη χρηματοδότηση των συστημάτων ή για το πώ τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τα σχεδιάσουν. Για το ποιο είδη, ποια είδη καθεστώτων θα πρέπει να θεσπίσουν τα κράτη-μέλη και ποιο είναι το επίπεδο προστασίας που θα πρέπει να παρέχεται. Τα στοιχεία αυτά που φυσικά είναι σημαντικά στον τομέα αυτό αφήνονται να καθοριστούν από τα κράτη-μέλη καθώς είναι αρμόδια στον τομέα αυτό. Η σύσταση καλύπτει ως προς το ουσιαστικό πεδίο εφαρμογή ε, έξι κλάδους κοινωνικής προστασίας, ε, τις ε, παροχές για την μητρότητα και την πατρότητα, την ασθένεια, τις συντάξεις, τις παροχές σε σχέση με τα εργατικά ατυχήματα και τις παροχές αναπηρίας και σε προσωπικό πεδίο εφαρμογής καλύπτουμε όλους τους εργαζομένους και τους αυτοπασχολούμενους. Ε, υπάρχουν τέσσερα κυρία στοιχεία στη σύσταση. Καλεί τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν υποχρεωτική κάλυψη κοινωνικής προστασίας για τους εργαζόμενους ε, σε όλους τους τομείς που σας ανέφερα μόλις και καλεί τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν υποχρεωτική κάλυψη για τους αυτοπασχολούμενους σε όλους αυτούς τους τομείς με εξαίρεση της, ε, τα επιδόματα ανεργίας, όπου προτείνουμε μια εκούσια προσέγγιση. Επίσης, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα που αποκτά κάποιος ε, στο πλαίσιο της κοινωνικής προστασίας μπορούν να μεταφερθούν από την ε, μία δουλειά στην άλλη. Έτσι λοιπόν έχουμε και κάποια στοιχεία που αφορούν ε, τη δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων κοινωνικής προστασίας και ότι οι κανόνες που σήμερα διέπουν τα δικαιώματα και τις εισφορές ε, στο σύστημα κοινωνικής προστασίας σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούν εμπόδια σε νέες μορφές απασχόλησης. Και τέλος, έχουμε και ένα σημείο που αφορά τη διαφάνεια για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες διαθέσιμες στους πολίτες σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους αλλά και τα δικαιώματά τους ε, στον τομέα της κοινωνικής προστασίας. Θα μπορούσα να πω και άλλα, αλλά θα σταματήσω εδώ γιατί νομίζω κάλυψα τα πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Τώρα για το ΕΛΚ. Ο κύριος Μπέκερ. Ε, να του δώσουμε το λόγο αφού καθίσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την εκπρόσωπο της Κομισιόν για αυτό το θέμα. Το ΕΛΚ θέλει να προτείνει δύο πρόσθετε ερωτήματα. Το ένα θα πρέπει να λέει έχοντας κατά νου ότι η πρόταση θα θίξει ιδίω τι μικρές ε, και μεσαίες επιχειρήσεις, πώς θα διασφαλίσει η Κομισιόν ότι η σύσταση δεν θέτει δυσανάλογο άχθος σε αυτές, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στη ΜΜΕ. Δηλαδή, η αξιολόγηση αντικτύπου της Κομισιόν λέει ότι οι ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις κυρίως εθίγονται από αυτή τη νέα πρόταση. Γι' αυτό θέλουμε να έχουμε αυτή την ερώτηση. Και το δεύτερο, η πρόταση λαμβάνει υπόψη διάφορα εθνικά συστήματα κοινωνικής προστασίας και την ε, οικονομική τους βιωσιμότητα. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να τεθεί στην προφορική ερώτηση για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Και υπάρχει και άλλη μια πτυχή αναφορά στον ε, πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Ε, είναι πιο πλήρης και καλύπτει όλα τα στοιχεία που θέλουμε να καλύψουμε στην προφορική ερώτηση. Θα πρέπει λοιπόν να διαγράψουμε την παραπομπή στο ψήφισμα, γιατί δεν ε, χρειάζεται αυτή η αναφορά στο ψήφισμα αν ε, αναφερόμαστε στον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Γκουτιέρες Πριέτο, παρακαλώ, για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και την ε, εκπρόσωπο της Κομπισιόν για την ε, παρέμβασή της. Θα πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τελικά συζητάμε για το πώς θα κάνουμε διανομή του πλούτου ή πώς θα συνεχίσουμε να διατηρήσουμε το ουσιαστικό στοιχείο που μας διαφοροποιεί από οποιοδήποτε άλλο μέρος ε, στον κόσμο, το κοινωνικό μας μοντέλο, δηλαδή η κατανομή του πλούτου, της ανάπτυξης που παράγει η οικονομία μας και επίσης πώς θα μειώσουμε τις ανισότητες διατηρώντας μια συνεκτική κοινωνία. Είδαμε πως τα έτη της οικονομικής κρίσης, το χάσμα μεταξύ των φτωχών και των πλούσιων πολυπλασιάστηκε στι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό οφείλεται κυρίω σε δύο λόγου. Καταρχήν, επειδή η απασχόληση έχει χάσει πολλά σε ποιότητα και έχουν, έχει υπάρξει και μεγάλη μείωση των μισθών ω συνταγή εξόδου από την κρίση. Αυτό το είχαμε ως κοινό παρανομαστή σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το δεύτερο είναι ότι η ανακατανομή μέσω της κοινωνικής προστασίας ε, επίσης πάγωσε. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε ένα νέο μέλλον που θα είναι ικανό να διατηρεί το σύνδεση των πολιτών ε, με τις δημοκρατικές κοινωνίες, με τα δημόσια συστήματα, ακριβώ μέσω κάποιων πολιτικών που αναδιανέμουν τον πλούτο. Η σύσταση της Κομισιόν που αποτελεί επίσης συνέπεια ε, της πολιτικής ε, δέσμευσης ε, που τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν κάναμε πέρσι στο Γκέτεμπουργκ προκειμένου να εγγυθούμε ίσες ευκαιρίες στο σύνολο των κοινωνιών μέσω του κοινωνικού πυλώνα, δεν μπορεί να αποτελεί απλώς μια διακήρυξη προθέσεων θα πρέπει να τα υλοποιήσουμε αυτά στην πράξη και γι' αυτό οι συστάσεις δεν είναι το καλύτερο εργαλείο δεν είναι το πιο δεσμευτικό νομικό εργαλείο, ούτε το πιο ισχυρό πολιτικά για να μπορέσουμε να τα θέσουμε όλα αυτά στην πράξη. Δεν είναι η πρώτη σύσταση που γίνεται προς αυτήν την κατεύθυνση. Ήδη το 1992 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια σύσταση σε όλα τα κράτη-μέλη και 26 χρόνια μετά συνεχίζουμε χωρίς να μπορούμε να εφαρμόσουμε το κοινωνικό μοντέλο έτσι όπως το είχαμε σχεδιάσει εδώ σε επίπεδο ευρωπαϊκών οργάνων. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να περάσουμε από τις συστάσεις, τις αποφάσεις, στις οδηγίες για να δημιουργήσουμε ένα ελάχιστο κοινό παρανομαστή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την ποιότητα των θέσεων απασχόλησης, την κοινωνική προστασία που θέλουμε να δώσουμε στις κοινωνίες μας και για να στείλουμε και ένα μήνυμα ελπίδας στους πολίτες που έχουν υποφέρει πολύ τα τελευταία δέκα χρόνια οικονομικής κρίσης και έχουμε την πολιτική υποχρέωση αλλά και η ηθική υποχρέωση να μπορέσουμε να του εγγυηθούμε ένα μέλλον με πιο ίσε ευκαιρίε. Έτσι λοιπόν, εμεί υποστηρίζουμε το κείμενο τη Κομισιόν, ε, δεν ε, κατανοούμε την πρόθεση του ΕΛΚ να επιχειρήσει μέσω νέων ερωτήσεων ε, να μειώσει το πολιτικό βάρος αυτής της ερώτησης και αυτής της σύστασης. Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο σε όλα τα βήματα που κάνουμε να υπάρχει ισχυρή δέσμευση απέναντι σε μια πιο δίκαιη κοινωνία με περισσότερες ε, ευκαιρίες, με ισότητα ευκαιριών. Ευχαριστούμε. Κυρία Μάκιντάιρ. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τη Σκιώδη. Και η ομάδα μας θα ήθελε να διασφαλιστούν δύο σημαντικές πτυχές στο ερώτημα, στην ερώτηση προς την Κομισιόν. Η πρόταση για σύσταση όσον αφορά τους αυτοπασχολούμενους και τους άλλους εργαζομένους σημαίνει ότι οι χώρες που είναι σε καλύτερη θέση για να λάβουν αποφάσεις για την προστασία των αυτοπασχολουμένων και τους ε, εργάτες νέες μορφές εργασίας θα πρέπει να τοποθετηθούν. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά συστήματα στην Ένωση που αντανακλούν διαφορετικές παραδόσεις και προτιμήσεις. Παρ' όλα αυτά, Αξίζει να ασχοληθούμε με την διαφοροποίηση που βοηθάει τις ε, επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Και αυτή η διαφοροποίηση διασφαλίζει και την ελκυστικότητα των διαφορομορφων μορφών εργασίας. Θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε από την Κομισιόν για τις επιλογές που έχουν οι χώρες μέλη στην ευκαιρία τους θα δούμε λοιπόν, θα θέλουμε να δούμε το πώς η Κομισιόν αντανακλά ακριβώς αυτή την ετερογένεια αυτών των μορφών απασχόλησης στις χώρες της Ένωσης και κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να γίνει με θετικό τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Καλβέ Αμπών λείπει. Μήπως κάποιος τον αντικαθιστά. Η Γκουε. Όχι. Και αυτοί λείπουν. Πράσινη. Η κυρία Τζιν Λάμπερτ και αυτή λείπει. FTD η Λόρα όχι ούτε και αυτή ο κ. Μαρτέν για το ΙΕΝΕΦ ο κ. Μελά ε, ζητά συγγνώμη επειδή έχει κολλήσει στο, στην κίνηση από το αεροδρόμιο ωραία λέει ο πρόεδρος κλείσαμε με το γύρο τοποθετήσεων τον Ιούλιο θα ψηφίσουμε 12 Ιουλίου και μετά στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο του 18. Αυτά για αυτό το σημείο. On και έχουμε ακόμα δύο-τρία λεπτά, μήπως η Κομισιόν θέλει να δώσει κάποιες σύντομες απαντήσεις γιατί σε λίγο θα ψηφίσουμε σε λίγα λεπτά και μισή. Παρακαλώ κυρία μου. Ναι, καταρχάς να, ευχαριστώ, να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για το ενδιαφέρον για τη σύσταση. Πρόεδρος Διακόπτη, σας παρακαλώ πολύ, κάνετε ησυχία να ακούσουμε την Κομισιόν και την απάντησή της. Παρακαλώ, παρακαλώ κυρία μου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και πάλι λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για το ενδιαφέρον που δείξατε για αυτή τη σύσταση. Και να πω βέβαια ότι οι συζητήσεις μας συνεχίζονται στο Συμβούλιο και η συμβολή του Κοινοβουλίου έχει μεγάλη σημασία για μας. Ως Κομισιόν, με χαρά βέβαια θα απαντήσουμε τις ερωτήσεις του Κοινοβουλίου στη συνέχεια και βλέπουμε ότι η ποικιλομορφία των συστημάτων στις χώρες μέλη αποτελεί μια αξία για την Ένωση και ελπίζουμε η σύσταση να στηρίξει αυτή την ποικιλομορφία. Αλλά βέβαια θα πρέπει να στηρίξουμε και να υποστηρίξουμε τις ίδιες ευκαιρίες και την ίδια προστασία για όλους στην Ένωση. Αυτό λοιπόν αφορά τους πολίτες της Ένωσης και ελπίζουμε να αναγνωρίσετε τους τρόπους με τους οποίους χρηματοδοτούνται τα συστήματα και διοργανώνονται. Αυτό παραμένει ανοιχτό και έγκυται στις χώρες μέλη να διερευνήσουν τις δυνατότητε αυτές αφού εφαρμόσουν τη σύσταση. Αυτά από μένα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα περιμένουμε ακόμα Δύο-τρία λεπτά για να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Ωραία, για τη διαδικασία. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη ψηφοφορία για το τριμερή διάλογο του σχεδίου προπολογισμού 2019. Παρακαλώ, κάντε ησυχία, λέει ο πρόεδρο. Πρώτη λοιπόν ψηφοφορία, ξαναλέει ο Πρόεδρο για την εντολή σχετικά με το τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προπολογισμού 2019 ζητήθηκε να αφαιρεθούν το 5 και 6 από την ημερήσια. Ε, θα ήθελα να μου πείτε αν είστε υπέρ ή κατά της αφαίρεσης των σημείων 5 και 6 της ημερήσιας διάταξης. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά και μετά ανάλογα με το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που έγινε άμεσα θα περάσουμε στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες σε σχέση με τα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Αυτά για τα διαδικαστικά. Περιμένω να καθίσετε όλοι σας. να βάλετε και το, την κάρτα σας στο μηχανηματάκι. Ωραία. Προτείνω να ξεκινήσουμε. Μιλάμε πάντοτε για το σχέδιο προπολογισμού 2019 και την εντολή για τον τριμερή διάλογο. Ναι, κύριε Ερμέρ. Μια ερώτηση διευκρινιστική σε σχέση με αυτά που είπατε. Τώρα τι ψηφίζουμε συγκεκριμένα τι, είναι αυτό το οποίο ψηφίζουμε, ποια γνωμοδότηση, τι ψηφίζουμε τέλος πάντων αυτό, τι ακριβώς ψηφίζουμε. Γιατί είναι σημαντικό. Κάντε μια ερώτηση. Ακριβώ να μα πείτε περί σε πρόκειτο. Ναι, καταρχά για το κείμενο του προπολογισμού, ξεκάθαρα αυτό. Δεύτερη ψηφοφορία σε σχέση με το αίτημα κάποιων ομάδων να αφαιρεθούν από την ημερήσια διάταξη τα σημεία 5 και 6. Θα ψηφίσουμε αν είμαστε υπέρ τη αφαιρεση ή κατά τη αφαίρεσης, δηλαδή τη παραμονή αυτών των σημείων. Να μας πείτε λοιπόν αν θέλετε να παραμείνουν τα σημεία 5 και 6 στην ημερήσια και να προχωρήσουμε αντίστοιχα ή να τα αφαιρέσουμε. Γι' αυτά λοιπόν θα ψηφίσουμε. Είναι ξεκάθαρο. Όχι, δεν είναι ξεκάθαρο, λέει κάποιο, ε, ποιε είναι οι επιπτώσει, γιατί έχουν και την Ολομέλεια. Ναι, κοιτάξτε, αν υπερψηφίσουμε χωρί να πάμε στην Ολομέλεια, αν ψηφίσουμε να αφαιρεθεί, δεν θα πάει στην Ολομέλεια. Αν ψηφίσουμε να παραμείνει, θα πάει στην Ολομέλεια. Απλό είναι. Αλλά ούτω ή άλλω πρέπει να ψηφίσουμε, έτσι. Κύριε Λαβριό, Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι σημαντικό να ακούσετε όλοι, όλοι οι παρόντες. Εντάξει για την ε, πρώτη ψηφοφορία, προπολογισμό εντάξει, δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχουν προβλήματα. Για το δεύτερο σημείο έχουμε θέμα διαδικαστικό. Γιατί μιλάμε για τον τύπο και όχι την ουσία. Για ένα θέμα όμω τύπου διαδικαστικό, από εκεί μπορούν να απορρεύσουν πολύ σημαντικά ζητήματα ουσίας. Γιατί αν τα αφαιρέσουμε από την ημερήσια, ανεξάρτητα την άποψη που έχουμε για το κείμενο, δεν θα έχουν το σύνολο των βουλευτών την ευκαιρία και το δικαίωμά του το αναπόσπαστο, να τροποποιήσουν το κείμενο. Ανεξάρτητα από την εθνικότητα του κάθε βουλευτή εδώ, ανεξάρτητα από την πολιτική τοποθέτηση ή την πολιτική οικογένεια του κάθε βουλευτή, υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε. Δηλαδή την ίδια την υπόσταση του Ευρωβουλευτή. Δηλαδή τη δυνατότητα να τροποποιήσει στην Επιτροπή ή στην Ολομέλεια το κείμενο, αν υπάρχουν βέβαια οι προποθέσει. Διαφορετικά δεν έχουμε πια υπόσταση βουλευτή. Να αφαιρέσουμε λοιπόν αυτά τα δύο σημεία από την ημερήσια δεν σημαίνει ότι είμαστε υπέρ κατά του κειμένου. Δεν έχει σημασία εξάλλου. Και καταλήγω, Πρόεδρε, αλλά νομίζω είναι σημαντικό να το διευκρινίσουμε αυτό για αυτά τα ζητήματα. Θα έλεγα λοιπόν, αυτοί που θέλουν να αποτρέψουν τους βουλευτές να τροποποιήσουν τα κείμενα δεν έχουν λόγο να το κάνουν γιατί έχουν πλειοψηφία. Τη στιγμή που αυτοί που θέλουν να τροποποιήσουν ίσως να είναι μειοψηφία γιατί λοιπόν μας τα απαγορεύουν και αφήνουμε τον Λομέλη να αποφασίσει. Το είχαμε συζητήσει και ο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα, πρόεδρο. Σα είπα ποιο είναι το διακύβευμα. Δεν θέλω να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, γιατί αν αρχίσουμε συζήτηση στι 10 δεν θα έχουμε ψηφίσει καν. Και έχουμε πάρα πολλά σημεία στην ημερήσια διάταξη, οπότε προτείνω, λέει ο Πρόεδρος, να προχωρήσουμε είναι ξεκάθαρη και η διαδικασία και η ψηφοφορία. Οπότε θα ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία για τον προπολογισμό, σχέδιο προπολογισμού 19. Τροπολογία 1. Ναι, λέει ο πρόεδρο. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Έχουμε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται τροπολογία 3 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται τροπολογία 4 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συγγνώμη, α. Συμβαστική α. 11, τροπολογία 11, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική β, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική γάμα. Συμβαστική γάμα. Υπέρ. Κατά.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 αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 25 άρχεται η ψηφοφορία περάς εγκρίνεται 25-19 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27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 Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για το σύνολο. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας της ψηφορίας. Εγκρίνεται 37, 7 και 3 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Maintenant, vote de procédure. Και τώρα ψηφίζουμε από τις διαδικασίες για να είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Έχουμε στην μέση διάταξη το σημείο 5 και το σημείο 6. Έχει ζητηθεί από ορισμένε πολιτικέ ομάδε να αποσυρθούν αυτά τα δύο σημεία από την μέση διάταξη. Επομένω, αυτό που θα ψηφίσουμε τώρα είναι ηλεκτρονικά, όχι με ονομαστική κλίση. Ηλεκτρονικά λοιπόν θα ψηφίσουμε ναι, όποιοι είναι υπέρ τη απόσυρση, όχι όσοι είναι κατά τη απόσυρση αυτών των σημείων. Άρχεται η ψηφοφορία. Le vote est Πέρας ψηφοφορίας. παραμένει η ημερήσια διάταξη όπως ε, ήταν. Παραμένουν τα δύο σημεία δηλαδή, είναι ξεκάθαρο. Πρώτη ψηφοφορία. Απόσπαση οδηγών. για να τα πω πάλι ξεκάθαρα. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που είχαν κατατεθεί και τις έχει συμπεριλάβει η Επιτροπή Τραν, άρα δεν νομίζω ότι δεν κρίνω ότι μπορούμε να τις ψηφίσουμε εδώ πάλι. Πάλι κάποιες άλλες σε συμβιβασμούς της Τραν έχουν περιληφθεί, κάποιες όχι και αυτές είναι στον, κατά, στον κατάλογο ψηφοφοριών. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 έως 41 και 43. Άρα, ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Le vote est clos. Πέρας ψηφοφορίας. Υπέρ, λοιπόν, 29 κατά 18. Δεύτερο. Για το χρόνο διάρκεια οδήγησης. Έχουμε τις τροπολογίες εδώ που είναι σε συμβιβασμούς. Άρα θα τοποθετούμε στη 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. εγκρίνονται. 32 υπέρ 16 κατά. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν με τις ψηφοφορίες. Περνάμε στο σημείο 7. Είναι έκθεση του κυρίου Καλβέτ Σαμπόν. Θα κάνω ένα διάλειμμα, κάνα δύο λεπτά για να μπορέσουν ησύχως να αποχωρήσουν οι συνάδελφοι που θέλουν να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 Λοιπόν, διαφανής και προβλέψιμη ώρα εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το σημείο αυτό το λόγο ο κύριος Καλβέ Σαμπόν. Gracias. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. αξιότιμοι συνάδελφοι, αξιότιμοι σκιώδεις ηγητές, θα ήθελα να κάνω μια πολύ γενική παρουσίαση αυτή τη στιγμή της δικής μου τοποθέτησης και του έργου που έχω επιτελέσει. Για ένα σημαντικό φάκελο, κατά με τουλάχιστον, το θέμα των διαφανών και προβλέψιμων όρων εργασίας. Όποιοι έχετε μελετήσει την έκθεση και καταθέτετε τροπολογίες, θέλω να θεωρήσετε αυτήν την έκθεση ως ένα πρώτο σχέδιο έκθεσης. Είμαι απόλυτα ευέλικτος δηλαδή και μπορεί να βελτιωθεί φυσικά το κείμενο αυτό χάρη και στη δική σας συμβολή. Όμως, που έβαλα την ε, έμφαση. Εστίασα σε τρεις μεγάλους στόχους οι άξονες της οδηγίας αυτής της Κομισιόν. Πρώτο σημαντικό στόχος και λόγος, είναι ο λόγος ύπαρξης. Για την κοινή δουλειά. Θέλω να σας πω ότι θα καταβάλω σημαντικές προσπάθειες και θα δείξω την απαιτούμενη ευελιξία με απόλυτη αμεροληψία και χωρίς να με επηρεάζει η ιδεολογία μου γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ενώπιση των ευρωεκλογών για την Ευρώπη και για όλους αυτό ακριβώς που είναι και ένα από τα δύο σημεία από τον Γκέτεμπουργκ και τον κοινωνικό πυλώνα, πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτήν, πρέπει να αντικατοπτριστεί το έργο μα. Θέλουμε να έχουμε τουλάχιστον ε, κάποια στοιχειώδη ελάχιστα δικαιώματα για τους Ευρωπαίους ε, το κατοχυρωμένα. Άρα απόλυτα ανοιχτό λοιπόν και έχω επισκεφθεί και πολλούς, πολλές χώρες και έχω ακούσει και όλες εσάς με μεγάλη προσοχή και θα συνεχίσω να το κάνω. Αυτή λοιπόν είναι αφετηρία, ότι θέλουμε να έχουμε ένα πλαίσιο κατώτατων ελάχιστων δικαιωμάτων για τους Ευρωπαίους πολίτες. Όλοι οι πολίτες που εργάζονται είτε επικοινωνιακούν στην αγορά εργασίας ή ήταν στην αγορά εργασίας θα έχει επιπτώσεις ε, να βιώσει από όλες αυτές τις διατάξεις. Θέλουμε λοιπόν ένα το πλαίσιο για όλους τους Ευρωπαίους πολίτε Δεύτερο άξονα. Ίσως να μην και τόσο ξεκάθαρο, αλλά και αυτό σημαντικό στο πλαίσιο εξέλιξη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να κατοχυρώσουμε το ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού level playing field όπω λέγεται στα αγγλικά για την ενιαία αγορά. Νομίζω ότι υπάρχει πραγματική επίθεση κατά της κινητικότητας, κάτι πολύ εσφαλμένο. Αυτό θα σημαίνει το τέλος Ευρώπης. Αυτή η επίθεση κατά της ε, κινητικότητας στόχο έχει όταν υπάρχει διαφορετικό κόστος εργασίας να εμποδίσει αυτή την κινητικότητα. Και όταν υπάρχουν και μισθολογικές διαφορές, αυτό φυσικά αντιβαίνει ε, πλήρως στην έννοια τη μια αγοράς που ε, έχει, χαρακτηρίζεται από πλήρη κινητικότητα και δεν είναι βέβαια και δίκαιο για όλους τους εργαζομένους, καθότι δεν επιτυχάνεται σύγκληση. Για να το αποφύγουμε αυτό, πρέπει να επιβάλλουμε ένα σύστημα παιχνιδιού όρου παιχνιδιού ισότιμους, ίσους, για να μην υπάρχει ποτέ ανταγωνισμός πάνω στα δικαιώματα των εργαζομένων, όσο και αν κοστίζει. Κάθε χώρα θα πρέπει να προβεί στις δικέ τη ρυθμίσεις. Σίγουρα καλό είναι να υπάρχει βέβαια ευρωπαϊκή οικονομική αλληλεγγύη και όλα αυτά που θέλετε, αλλά δεν μπορεί να γίνει ανταγωνισμό ε, πάνω στα βασικά δικαιώματα των εργαζομένων. Όταν κάποιο είναι Ευρωπαίο πολίτη και Ευρωπαίο εργαζόμενο, σημαίνει ότι υπάρχει μια κοινή βάση και από εκεί και πέρα ξεκινά το παιχνίδι. Αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντική πτυχή και πρέπει να συμφωνήσουμε σε σχέση με αυτή τη βάση, τη βέλτιστη βάση που περιλαμβάνει βέβαια και τις διαφορετικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες ε, των κρατών μελών. Από οικονομικές μέχρι και κλιματικές συνθήκες. Και βέβαια όταν έχουμε καταλήξει τα βασικά, φυσικά έρχεται μια στιγμή, αφού έχουμε πλέον κατοχυρώσει τα βασικά δικαιώματα των εργαζομένων, φτάνει λοιπόν η στιγμή που λειτουργεί η αποκέντρωση, η επικουρικότητα θα έλεγα, κυρίω η αποκέντρωση στη δικασία λήψη αποφάσεων. Αν είναι κάποιο εργαζόμενο στην Εστρεμαδούρα, δεν είναι το ίδιο με τον είναι εργαζόμενο στο Τούρκου, στη Φιλανδία. Τυχαία τα πήρα αυτά τα, δύο μέρη παρά. Γιατί υπάρχει και το κρύο στο Τούρκου, τέλο πάντων. Αλλά εγώ εδώ μιλάω για την πρακτική εφαρμογή που γίνεται επί τόπου φυσικά. Αλλά τα δικαιώματα πρέπει να είναι τα ίδια και μπορούν να είναι τα ίδια. Τρίτον, προφανέστερο και σημαντικό στόχος ε, της οδηγίας αυτής και είμαι και ευέλικτος και θα είμαι στη σας για προτάσεις. Ότι δηλαδή de dar una βάση, μια κατώτατη βάση δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά όλες αυτές τις νέες μορφές εργασίας που ήδη γνωρίζουμε. Ή που δεν γνωρίζουμε, αλλά θα έρθουν λόγω της τεχνολογίας που ξελίσσεται τάχιστα. Μιλώ δηλαδή για τους προσωρινούς εργαζόμενους, ε, για τα voucher, για τα zero hours, για τις πλατφόρμες και άλλα που μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή. Η Κομισιό προσπαθεί να κάνει ένα, ε, φτιάξει ένα πλαίσιο με όλες αυτές τις νέες μορφές συμβατικών σχέσεων. Ωραία όλα αυτά. Αλλά αν υπάρχει σχέση οικονομικής εξάρτησης ε, και οργανωτικής Οργάνωση εργασίας ή σε ό,τι αφορά το ωράριο. Υπάρχουν δικαιώματα που πρέπει να εφαρμόζονται όπου και αν βρίσκεται ο εργαζόμενο σε όποια χώρα τη Ευρώπη και αν εργάζεται. Εκεί που δεν θα είμαι ευέλικτο είναι στο εξή. Αυτοί οι εργαζόμενοι που εργάζονται με νέες μορφές εργασία. νυν και επόμενες και μελλοντικέ. Αν δεν κατοχυρώνω τα δικαιώματα αυτών των εργαζομένων, εγώ δεν θα ψηφίσω, δεν θα υπογράψω την οδηγία αυτή. Αυτό είναι το μόνο στο οποίο δεν θα είμαι ευέλικτος και παρακαλώ να συμφωνήσουμε όλοι ως προς αυτό. Και να θεωρήσουμε ότι είναι ένας στόχος. Τώρα πώς θα προχωρήσουμε, πώς θα το διατυπώσουμε και πώς θα εφαρμοστεί, αυτά όλα είναι υποδιαπραγμάτευση. Τότε που έκανα τι προτάσει μου, έχω μιλήσει με πολλού και έχω πάει σε πολλέ χώρε γιατί. επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ε, θέλω να πω ότι αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ είναι να προχωρήσουν προς τα εμπρός και να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό. Έχοντας υπόψη βέβαια ότι το καλύτερο είναι εχθρό του καλού. Τούτων λεχθέντων Έχω καταθέσει κάποιε τροπολογίε για το προσχέδιο αυτό. Που επαναλαμβάνω ότι θα εμπλουτιστεί με τι δικέ σα ε, ε, συνεισφορέ και με την επισκέψη που έχω να κάνω ακόμη. Όλε σα τι προτάσει λαμβάνω υπόψη. Έχω ήδη καταθέσει και εγώ τροπολογίε. Αν διαιρέσουμε, σε τα τρία έχουμε ένα πρόβλημα. Τρει άξονε. Δικαιώματα, μάλιστα να τελειοποιήσουμε αυτό το κομμάτι. Όλα είναι διαπραγματεύσιμα, είμαι ευέλικτο, ε, θα βρούμε πιστεύω το σημείο ισορροπίας για τα κατώτατα ε, δικαιώματα. Το ίδιο ισχύει και για το δικαίωμα στην πληροφόρηση. Μετά έχουμε όμως την εφαρμογή. Εκεί νομίζω πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να βρούμε αυτή την ισορροπία μεταξύ επικουρικότητας και αναπόφευκτης υποχρέωσης δημιουργίας αυτού του πλησίου ε, στην Ευρώπη. Δεν θα σας ε, πω ψέματα και ολοκληρώνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Βλέπω ένα μεγάλο κίνδυνο. Το πρόβλημα δηλαδή του ορισμού θα εργαστούμε σκληρά, υπάρχουν λύσεις, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι τόσο να δούμε ε, πώς θα λύσουμε όλα τα νομικά προβλήματα και πώς ε, θα ρυθμίσουμε όλες τις λεπτομέρειες. Έχουμε το φυσικό δίκαιο, έχουμε το bargaining κτλ. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει το πεδίο εφαρμογή. Αν όλοι καταβάλουμε προσπάθεια για να φτάσουμε στο κεντρικό αυτό στόχο, το πεδίο εφαρμογή, νομίζω ότι το μεγάλο αυτό πρόβλημα του ορισμού θα το λύσουμε. Ευχαριστώ. Merci pour le PPE, Denis Radke για το έλκο ο κυρίος ε, Ντένις Ράτκε. Ναι, ευχαριστώ πολύ αξιότιμη εισηγητά, αξιότιμοι συνάδελφοι. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς θερμά τον εισηγητή για το έργο του. Διάβασα το σχέδιο έκθεσης ε, προσεκτικά και θέλω να τον ευχαριστήσω διότι σε ό,τι αφορά αυτή τη βασική κατεύθυνση της οδηγίας ε, έχει ακολουθήσει το σωστό δρόμο. Πραγματικά. Διαμφισβείται δηλαδή, τα σωστά αυτά που είπε Εμείς ως νομοθέτες τώρα θα πρέπει να αντιδράσουμε πέτσα αυτή τη θεμελιώδη, την άρδην αλλαγή που βλέπουμε τα τελευταία 25 χρόνια στο πλαίσιο της ενίας αγοράς. Και δεν μιλάω μόνο για κάποιες εθνικές αγορές εργασίας, αλλά και την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Εμείς ως νομοθέτε εδώ ε, δεν ε, θα πρέπει να ε, απολαμβάνουμε μόνο των προνομίων μας, αλλά να βλέπουμε τι γίνεται στην αγορά εργασίας και να προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τους εργαζομένους. Και θέλουμε το σχέδιο αυτό να πηγαίνει προς σωστή κατεύθυνση. Θέλω να αφαιρθώ σε κάποια σημεία, για τα οποία δεν είμαι και τόσο σίγουρος κατά πόσον είμαστε στη σωστή κατεύθυνση ή μήπως δημιουργούμε προβλήματα. Και αρχικά ε, θα μιλήσω για την νομική ισχύ και εφαρμογή σε ό,τι αφορά τον ορισμό του εργαζόμενου στην οδηγία. Δεν μπορούσε να δώσει κανείς ε, μια νομικά δεσμευτική απάντηση για το ποιε είναι οι νομικέ επιπτώσεις ε, του ορισμού και τι επιπτώσεις θα υπήρχαν σε ό,τι αφορά και τον ορισμό ε, του εργαζόμενου στο αστικό δίκαιο. Από, μιλάω για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας εδώ. Αλλά έχουμε και κάποιες ε, άλλες, έχουμε έναν άλλον ορισμό για, συνταγματικό για τον εργαζόμενο στη Γερμανία. Θα πρέπει να τα δούμε και μέχρι τώρα δεν κατάφερε κανείς να δώσει μια δεσμευτική ε, απάντηση στο πώς συνδυάζονται ενδεχομένως ή όχι αυτοί οι δύο ορισμοί. Και αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο το οποίο θέλω να το θέσω στο τραπέζι. Το δεύτερο σημείο που για μένα είναι σημαντικό σε ό,τι αφορά την ε, διεύρυνση του καταλόγου για το δικαίωμα στην πληροφόρηση. Ε, το δικαίωμα όλων των εργαζομένων στην πληροφόρηση φυσικά είναι ένα διαφυσβήτητο ε, στόχος. Πρέπει να διευρυνθεί ο κατάλογος. Η ε, δοκιμαστική περίοδος είναι μεγαλύτερη και τι γίνεται με τις αμοιβέ. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα συζητήσουμε και θα πρέπει και νομικά να ρυθμιστούν αυτά. Το θέμα είναι αν δει κανείς το κατάλογο συνολικά δεν ξέρω αν έχει νόημα να κάνουμε αυτή την τομή και να πούμε από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μέρα ε, θα πρέπει ε, να ισχύουν αυτά ή να κάνουμε μια διάκριση και να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες βασικές πληροφορίες για την αμοιβή, για τις περορίες κτλ. κτλ που από την πρώτη μέρα θα πρέπει να οριστούν και υπάρχουν άλλες πληροφορίες όπως είναι η επιμόρφωση για παράδειγμα που μπορεί να δοθεί σε μεταγενέστερο στάδιο αυτή η πληροφορία. Αυτό είναι μια ερώτηση που φαντάζομαι ότι στις ε, διαπραγματεύσεις που θα έχουμε θα διευκρινίσουμε. Άρα, βασική κατεύθυνση, λέω, ναι, να διευρυνθεί ο κατάλογος, ε, αυτό δεν το θεωρώ επίμαχο ή αμφιλεγόμενο, το θέμα είναι πώς θα γίνει αυτό από οργανωτικής πλευράς. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς. Για το επόμενο, το ερώτημα μερική απασχόληση. αν αυτό δεν λέγεται στην αρχή. Και είναι νομική ερμηνεία. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θα πρέπει να τα επεξεργαστούμε, να τα διατυπώσουμε μεγαλύτερη ακρίβεια. και να δούμε και τις ασφαλιστικές δικλείδες. Επίσης, ό,τι αφορά τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, σε ό,τι αφορά συλλογικέ συμβάσει εργασία. Δεν μπορούμε να ε, ανατρέψουμε αυτό που έχουν συμφωνήσει οι κοινωνικοί εταίροι. Αυτό είναι το απόλυτα βασικό και σημαντικό. Αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και στην οδηγία αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριος Λόπες, για τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο του τις τελευταίες εβδομάδες και τους τελευταίους ε, μήνες. Και εμείς ε, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και συμφωνούμε με το φιλοπορίας που συζητούμε σήμερα. Καταρχήν αυτός είναι ένας φάκελος ε, που θα πρέπει να μπορέσουμε να τον εγκρίνουμε κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα από τα νομοθετικά εργαλεία που κατορθώνει να παγιώσει τον ε, πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Επίσης, θα πρέπει να ανανεώσουμε το ελάχιστο πλαίσιο των εργασιακών όρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουμε νομοθετήσει τα τελευταία 15 χρόνια ε, στον τομέα. Αυτή η οδηγία είναι από τη δεκαετία του 90 και επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις βαθιές αλλαγές που υφίσταται η έργα εργασίας όπως ε, το προσωρινό χαρακτήρα της εργασίας, πώς ε, δημιουργούνται οι εργασιακές σχέσεις. Είναι δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου, την αποδυνάμωση των δικαιωμάτων και στις συλλογικέ διαπραγματεύσεις. Και επομένω θα πρέπει να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αλλαγέ και τι ε, τροποποιήσεις ε, στου όρου εργασία. Θα ήθελα τώρα να μπω σε λεπτομέρειες σε κάποιες πτυχές. Καταρχήν θα αναφέρω τα θετικά στοιχεία που πιστεύω ότι συμπεριλαμβάνει η πρόταση του εισηγητή και στη συνέχεια θα αναφερθώ σε κάποια στοιχεία που θεωρούμε ότι πρέπει να συζητηθούν τις επόμενες εβδομάδες. Καταρχήν μας φαίνεται ότι είναι πολύ καλά που σχετίζουμε ξεκάθαρα το φάκελο με τον κοινωνικό πυλώνα και επίσης ε, ότι υπάρχει ε, έτοιμα για περισσότερη πληροφορία για ε, την κοινωνική ασφάλιση και το υποχρεωτικό μητρό. Γίνεται μια μικρή αναφορά, θολή αναφορά στην δυνατότητα να προβλέπονται συμβάσεις μηδενικών ορών. Εμεί νομίζουμε ότι πρέπει να ενισχυθεί αυτό το στοιχείο. Επίσης είναι θετικό το να αναφέρονται οι επιθεωρητές ε, ε, των κρατών μελών, γιατί αυτοί θα είναι οι πρωταγωνιστές που θα εφαρμόσουν συνέχεια την εργασιακή νομοθεσία. Επίσης, οι βελτιώσεις που γίνονται στην ε, παροχή ενημέρωσης, πληροφόρησης, τόσο και γραπτός, όσο και επιγραμμικά. Θεωρούμε ότι και αυτό είναι θετικό. Επίσης, οι περιορισμοί παράλληλης εργασίας και η αναγκαιότητα να εμπλακούν οι κοινωνικοί εταίροι στην εφαρμογή της οδηγίας. Αυτά είναι νέα στοιχεία σε αντίθεση με την πρόταση της Κομισιόν ε, που πιστεύουμε ότι πρέπει να τονιστούν γιατί είναι θετικά. Τώρα, πού θα κάνουμε κάποια συζήτηση και θα αναφερθώ και σε κάποια στοιχεία που αναφέρθηκε ο συνάδελφος ε, στο ΕΛΚ. Με κάποια στοιχεία συμφωνώ, έχουμε κάποια κεντρικά στοιχεία ε, στη συζήτηση και σίγουρα ο ορισμός θα είναι κεντρικό στοιχείο. Γιατί είναι ένα ευρωπαϊκό ορισμό. Καταρχήν ε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ήδη υπάρχει ένας ε, ορισμός. Έχουμε την ομολογία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων για την εργασιακή νομοθεσία και για την ευρωπαϊκή νομοθεσία ήδη υπάρχει ένας ορισμός για τον εργαζόμενο μέσω των δικαστικών αποφάσεων. Τι κάνει αυτή η οδηγία ε, βάζοντας τον ορισμό Δηλαδή, καθώς είναι μια οδηγία που ρυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις, ουσιαστικά διασφαλίζει ποιοι θα είναι εντός του πεδίου εφαρμογή της Δηλαδή, η συζήτηση δεν αφορά το ποιος είναι εργαζόμενος, αλλά το πόσο το πόση ασφάλεια δικαίου θέλουμε, τι κάλυψη θέλουμε και τι πραγματική επιβολή θέλουμε για αυτήν την οδηγία. Δεν αφορά ε, ουσιαστικά τον ορισμό συζήτηση, αλλά η συζήτηση πρέπει να επικεντρωθεί στο ποιο θέλουμε να καλύπτεται από την οδηγία, ποια θα είναι η ασφάλεια δικαίου και πώ θα γίνει η επιβολή. Και πρέπει να βρούμε ένα πραγματικό μηχανισμό, γιατί σίγουρα υπάρχουν οι ορισμοί των εργασιακών σχέσεων. Αυτό δεν θα αλλάξει και υπάρχει ήδη ένας ορισμός ε, από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Πολύ γρήγορα να προσθέσω. Εμείς ε, δεν θεωρούμε ότι πρέπει να εξαιρέσουμε την ε, εφαρμογή ε, για τους δημοσίους υπαλλήλου ή για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι αυστηροί οι όροι και πρέπει να συνδέσουμε την ενημέρωση με τα ελάχιστα δικαιώματα και θα πρέπει και να ενισχύσουμε ίσως αυτά τα ελάχιστα δικαιώματα. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε τις λογικέ διαπραγματεύσεις και να εντοπίσουμε την υπερβολική ευελιξία ε, και ξέρετε ότι είναι πρωταγωνιστικό το θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε κάποιες χώρες. Πρέπει να το ενισχύσουμε και θα πρέπει να ενισχύσουμε και την εφαρμογή γιατί αυτό κάνει τη διαφορά. Το ότι συζητάμε εδώ, αν στη συνέχεια δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί στην πράξη, δεν έχει κάποιο νόημα. Ευχαριστούμε κυρία Μακεντάιρ για τους ε, για το ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το πλήρες σχέδιο έκθεσης. Φυσικά έχουμε πολύ σημαντική δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της παροχής της απαραίτητης ευελιξίας για τις επιχειρήσεις προκειμένου να κάνουν τη δουλειά τους και να διασφαλίσουμε ότι μένουμε και εντός του πεδίου εφαρμογής ε, της, οδηγίας, της οδηγίας. Εμείς στην ομάδα μου έχουμε κάποιες ανησυχίες ε, που θα τις θέσουμε σταδιακά. Η προτεραιότητά μου είναι να διασφαλίσουμε ότι η έκθεση της Επιτροπής ε, και οι τροπολογίες που καταθέτω εξυπηρετούν την αρχική πρόθεση της πρότασης δηλαδή να θεσπιστούν ελάχιστα δικαιώματα για να προωθηθεί ασφάλεια και προβλεψιμότητα σε εργασιακές σχέσεις στα κράτη-μέλη. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ως συνομοθέτες να θυμόμαστε ότι μιλάμε για ελάχιστα δικαιώματα που προωθούνται από μια οδηγία και τα κράτη-μέλη στην πραγματικότητα είναι αυτά που θα μεταφέρουν τις λεπτομέρειες διατάξεις στο ιστορικό τους δίκαιο και ε, θα είναι σίγουρα ότι ταιριάζουν με την ιστορική τους νομοθεσία. Δηλαδή θα πρέπει να αποφύγουμε να έχουμε ουσιαστικά έβρισκε ε, και περιοριστικές ε, απαιτήσει. Ε, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ευελιξία στην νομοθεσία. Φυσικά χρειαζόμαστε το ελάχιστα πρότυπα, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει και επαρκή ευελιξία, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη θα μπορούν ε, αυτές τις ε, απαιτήσει ε, να τις εμπεδώσουν ήδη στις καθιερωμένες πρακτικές τους. Είναι ενδιαφέρον ότι η Σουηδία έθεσε μια κεντρική κάρτα σε αυτό το φάκελο. Στην περίπτωση αυτή δεν αφορά μόνο τους εργαζομένους και τους εργοδότες και τα συνδικάτα. Ουσιαστικά εμπλέκονται σε αυτό. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα, παραδείγματο χάρη στις δοκιμαστικές περιόδους. Η πρόθεση της Κομισιόν είναι να διασφαλίσει ότι η μετάβαση σε μια νέα θέση δεν ε, θέτει έναν εργαζόμενο σε παρατετεμένη περίοδο ανασφάλειας. Αν ε, δείτε τι συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, τα περισσότερα καθεστώτα ε, προστασία σχετίζονται με δοκιμαστική περίοδο και με τη διάρκεια της ε, παροχής συνεχούς υπηρεσίας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει ε, ουσιαστικά να σεβαστούμε την δυνατότητα του κράτους μέλους να ρυθμίζει αυτές τις δοκιμαστικές περιόδους. Άλλο παράδειγμα είναι όπου δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ο εργαζόμενος στη δοκιμαστική περίοδο και ο εργοδότης θέλει να δώσει μια παράδειγμα παράταση ως δεύτερη ευκαιρία και οι δύο θα μπορούν ε, να επιλέξουν να το δεκτούν αν είναι προ εξυπηρετήσει των συμφερόντων του. Έτσι λοιπόν εδώ δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την οδηγία ω ευκαιρία για να πούμε ακριβώ τα κράτη-μέλη πώ θα το κάνουν αυτό, αλλά θα πρέπει να του δώσουμε ένα πλαίσιο ελάχιστων προτύπων και θα πρέπει να σεβαστούμε την αρχή τη επικουρικότητα. Έχω ανησυχίε ε, με το άρθρο 2 και τον ορισμό του εργαζομένου. Θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό προσεκτικά. Όλοι οι απασχολούμενοι είναι εργαζόμενοι, αλλά δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι απασχολούμενοι. Επίσης, με ανησυχεί ε, ο ορισμός του εργοδότη. Η πρόταση και η πρόταση του εισηγητή να βάλουμε πρόσθετη διατύπωση ε, για όλους τους λοιπούς φορείς, όλες τις λοιπές οντότητες. Έχω λοιπόν αυτές τις ανησυχίες, ε, αλλά έχω και ανησυχίες για πολλά άλλα άρθρα. Παραδείγματο χάρη. Με ανησυχεί το άρθρο 11 για την κατάρτιση. Είναι ένα πολύ μικρό άρθρο. Όμως, Ε, επικοινώνησαν ε, μαζί μου κάποιες ενώσεις ε, πιλότων και πρέπει να διασφαλίσουμε την η νομοθεσία θα έχει και τις απαιτούμενες συνέπειες στο να προστατεύει τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν θα καταθέσω κάποιες τροπολογίες και υπομονώ να συζητήσουμε περαιτέρω επί αυτού του φακέλου. Ευχαριστώ. Για την ΚΟΕ, όχι. ο κύριος Μέζεριξ τους πράσινους. Ευχαριστώ. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Να τονίσω ότι συμφωνούμε και με τον οδικό χάρτη. Είναι σημαντικό ο Ευρωπαϊκό ε, Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων να μεταφραστεί σε οδηγίε. Και αυτή είναι η πρώτη μεγάλη οδηγία. Αν χάσουμε εδώ, τότε κινδυνεύει όλο το πρόγραμμα. Να πω επίσης ότι καλωσορίζουμε την ε, αρχική πρόθεση της Κομισιόν. Δεν ε, υπάρχει κάποια διάνοιξη εδώ, όμως ε, συμμερίζομαι κάποιες ανησυχίες που έθεσαν οι συνάδελφοι. Δεν θα τα επαναλάβω όλα αυτά για να γλιτώσουμε χρόνο. Όμως, ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία και αυτό αφορά την ε, περίπτωση υπερβολικής ευελιξίας ε, και αφορά τη σύμβαση μηδενικών ορών. Θα πρέπει να απαγορευτούν ε, αυτές οι συμβάσεις. Ε, θα πρέπει κάποιες εταιρείες να δοκιμάσουν κάποια άλλη μορφή ε, υλοποίησης των εργασιών τους σε σχέση με την κίτρινη κάρτα από τη Σουηδία. Το έθεσε η κυρία Μακεντάιρ. Είμαι κάπως απογοητευμένος που όσοι ενδιαφέρονται για το θέμα της κοινωνικής ολοκλήρωσης Ευρώπης και μεγαλύτερης πρόοδου θα πρέπει να συζητήσουν όχι ε, μόνο που ε, υπερισχύει η αγορά αλλά και με αυτό που θεωρούνται η προοδευτική πλευρά της Ευρώπης. Στις σκανδιναβικές χώρες ε, φαίνεται να προσυπογράφουν το σημερινό η οφθαλμαπάτη της απομόνωσης. Μέσω της απομόνωσης δεν μπορείς να πετύχεις σε αυτόν τον κόσμο. Ο ε, αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα. Λοιπόν, για τις ε, τροπολογίες θέλουμε οι, τα ε, άτομα υποκατάρτιση, οι μαθητευόμενοι να συμπεριληφθούν. Εργαζόμαστε τώρα για το πώς, όμως θέλουμε οι μαθητευόμενοι και τα άτομα που ασκούν πρακτική ε, έχουν το δικαίωμα ε, αλλά και είναι και στο συμφέρον μας ε, να τους συμπεριφερόμαστε όσο ισότιμοι εργαζόμενοι στην αγορά εργασίας είναι στην αγορά εργασίας όταν κάνουν την πρακτική τους έτσι λοιπόν πρέπει να ισχύουν και, αυτούς και, και για αυτούς τα ελάχιστα πρότυπα. πρότυπα. Επίσης θέλουμε να ενδυναμώσουμε τη θέση των κοινωνικών εταίρων και να υπάρχουν και εγγύησει ότι θα εφαρμοστεί η οδηγία και θα γίνει σεβαστή ακόμη και στην πιο απομακρυσμένη περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης ε, θέλουμε μια πιο εύρωστη οδηγία χωρίς ε, τα συνήθη ε, παραθυράκια που συνοδεύουν πολλές από αυτές τις οδηγίες και φυσικά θα υποβάλουμε και τις κατάλληλες τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω κυρίως τον συνάδελφο Αντρίκε Καλβέ Σαμπον για την πρόταση και για την προσπάθεια δημιουργίας μιας ισχυρής βάσης για αυτή την ευρωπαϊκή νομοθεσία με μια πρόταση νομοθετική που πραγματικά νομίζω βάζει τα θεμέλια αυτό που μέχρι τώρα ήταν ε, ισχυρό περιεχόμενο χωρίς πρακτική εφαρμογή, δηλαδή τα βασικά κοινωνικά δικαιώματα, τα ευρωπαϊκά. Ένα περιεχόμενο λοιπόν ενδιαφέρον συμπληρώθηκε, εμπλουτίστηκε και νομίζω σε αυτή την περίπτωση αυτά που είπαμε και συζητάμε για την διαφάνεια είναι σημαντικά. Εξάλλου θα πρέπει να υπάρχει και μια ελάχιστη βάση για τα δικαιώματα των εργαζομένων και θα πρέπει όταν χρησιμοποιούμε αυτή την λέξη να είμαστε πιο συγκεκριμένοι γιατί λείπει σαφήνεια σήμερα. Πολλά άτομα δηλαδή παρόλο που εργάζονται δεν απολαμβάνουν αυτής τη ιδιότητας των εργαζομένων. Οπότε το να αρχίζουμε να βάζουμε κάποια βάση, κάποια θεμέλια είναι κάτω καθοριστικής σημασίας. Εμάς μας ενδιαφέρουν δύο πράγματα. Καταρχάς να διευρύνουμε το φάσμα των δικαιωμάτων εργαζομένων και μετά να εντάξουμε και τους νέους εργαζόμενους με τις εξελίξεις που έχουμε στην αγορά εργασίας, με τις πλατφόρμες και άλλες μορφές νέες, ε, νέες μορφές εργασίας. Θα πρέπει στην Ευρώπη να υπάρχει μια αναφορά στο ότι δεν θέλουμε να αφήσουμε κανένα πίσω. Δηλαδή να θεσπίσουμε ελάχιστα δικαιώματα, θα πρέπει να προστατεύουν τα εργατικά του δικαιώματα ακόμα και σε περίπτωση απόλυση. Γιατί υπάρχουν ε, κάποιες συνθήκες οι οποίες θα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένε και να διασφαλίζονται και να πούμε ότι αυτέ είμαστε ανυποχώρητοι. Έχουμε και κάποια άλλα σχόλια, απορίες και παρατηρήσεις που θα θέλαμε να υποβάλουμε προς τον εισηγητή. Καταρχάς, η διάρκεια της δοκιμαστικής περίοδου. Έξι μήνες είναι πολύ μεγάλη περίοδος για δοκιμή. Οπότε και εδώ θα πρέπει να βρούμε μια σύγκληση μεταξύ των διαφορών αναγκών και θέσεων που υπάρχουν. Η ανάγκη της προστασίας των εργαζομένων με οποιαδήποτε μορφή εργασίας, με πλατφόρμες, με στάζ, με εκμάθησης, οι μαθητευόμενοι κλπ. Θα πρέπει εδώ να καλύπτουμε όλους αυτούς, ιδιαίτερα αυτούς που κάνουν στάζ, κάνουν διάφορες ε, περίοδους εκμάθησης και είναι απροστάτευτοι. Οι ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας και αυτές δεν περιλαμβάνουν καμία προστασία εργατικών δικαιωμάτων. Θα πρέπει λοιπόν οι εργαζόμενοι αυτοί και αυτοί να περιληφθούν εδώ στην οδηγία. Οι ντελιβεράδες στην Ιταλία είδαμε ότι τα ίδια τα συνδικάτα δεν τους θεωρούν ως εκπροσώπους αυτών των νέων κατηγοριών εργαζομένων. Είναι λοιπόν απαραίτητο τα ίδια τα συνδικάτα να μας βοηθήσουν εδώ. Θα πρέπει τα συνδικάτα να εκπροσωπούν όλους αυτούς τους εργαζομένους. Γιατί όλες αυτές οι κατηγορίες εργαζομένων χρειάζονται διαφάνεια και ενημέρωση όσον αφορά την περίοδο εκμάθησης, τις συνθήκε εργασίας, τα, τις περιορίες, τις αμοιβέ, τον προγραμματισμό ε, της εργασίας όσον αφορά τις, ε, τους ε, συμβασιούχους και θα πρέπει να δίδεται και απαραίτητες πληροφορίες σε σχέση με την κατάρτισή τους γιατί είναι πολύ βασικό αυτό ιδιαίτερα για αυτούς στις νέες μορφές οικονομίας θα πρέπει να υπάρχει μια πρόβλεψη ώστε ώστε να μην εξαρτώνται από το κινητό μέσω, μέσω του οποίου τους ενημερώνω ότι ε, τους θέλουν για δουλειά. Θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο μεγαλύτερο περιθώριο ελευθερίας και ασφάλειας. Επίσης, για να μην πληβαρούμε και τους εργοδότες, θα πρέπει οι χώρες μέλη ακριβώς να διευκολύνουν την διαδικασία όσον αφορά τις ε, γραφειοκρατικές διαδικασίες σε με τους ε, εργαζόμενους και θα πρέπει να υπάρχουν και οι απαραίτητες συνθήκες οι οποίες απορρέουν από τις συλλογικέ συμβάσεις διαθέσιμες με τρόπο ευκολονόητο και απλό. Αυτά πρώτα ευχαριστώ. Merci. Pour Ευχαριστώ. Κύριε Μελάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οπωσδήποτε χρειαζόταν να αναθεωρήσουμε αυτή την οδηγία για τις ε, συνθήκε εργασίας, τις προβλέψιμες και τι διαφανεί. και οι σχέσει που ρυθμίζονται μέσω σύμβαση μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου. Η ψηφιοποίηση, η χρήση των μηχανών, των ρομπότ και τα λοιπά στην εργασία προκαλούν πολλά ερωτηματικά και απορίες. Εξού και η ανάγκη ε, προσέγγιση όσον αφορά τις, ε, και σύγκληση όσον αφορά τις διάφορες προσεγγίσεις τις νομοθετικές. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε πιο δυσχερείς τις εργασιακές σχέσεις και για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζομένους. Ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτές που δηλαδή ε, προσφέρουν μεγαλύτερο αριθμό θέσεων εργασία. Επίσης θεωρούμε ότι οι χώρες μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν αποτελεσματικέ και προσαρμοσμένες λύσεις αναπερίπτωση. Πρέπει όμως να συμφωνήσουμε για τον ορισμό των εργαζομένων και της εργασίας η οποία αναζητείται και αποδέχεται και η εργασιακή εξάρτηση. Γιατί οι νέε θέσει εργασία, οι νέε μορφέ όπω οι πλατφόρμε κτλ. ακριβώ ε, διαγράφουν αυτή την εργασιακή εξάρτηση. Κάποια σημεία μας βοηθούν να το διευκρινίσουμε. Αλλά βλέπουμε ότι και άλλοι, όπως ο πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος είναι ξεκάθαρα φιλευρωπαίος, έχει προετοιμάσει ένα κειμένο με ένα ειδικό καθεστώς για τους αυτοαπασχολόμενους, το οποίο θα πάει στη Βουλή, ιδιαίτερα για αυτούς τους δελιβεράδες, οι οποίοι δεν έχουν καμία σύμβαση, δεν εφαρμόζεται για αυτούς κανένα εργασιακό δικαίωμα και δεν υπάρχει καμία νομική σύμβαση ή συμφωνία με καμία κοινωνική, μορφή κοινωνικής πρόνοιας ή κοινωνικής προστασίας, ένσημα κλπ. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν τεράστια προβλήματα και δεν θα πρέπει το γαλλικό κείμενο να επιβληθεί στην Ευρώπη. Το αντίθετο μάλλον. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε τι γίνεται και με τους δημόσιου υπαλλήλου, με το δημόσιο, ιδιαίτερα αυτούς που εργάζονται στον τομέα της άμυνας, που έχουν ιδιαίτερο καθεστώς. Ξέρουμε τι γίνεται με τους αποσπασμένου ή με παρόμοιες μορφές εργασίες όπου υπάρχει μη προβλέψιμος χαρακτήρας εργασίας. Και τέλος, θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα ώστε οι εργασίες που θα προκύψουν να μην επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την εργασιακή ανασφάλεια. Γιατί μεταξύ 10 και 30% των θέσεων αυτές της εργασίας τα επόμενα 10 χρόνια αντιμετωπίζουν κίνδυνο, ακόμα και στο δημόσιο, όχι αμέσα αλλά στο μέλλον, ναι. Και η νομοθεσία λοιπόν δεν θα πρέπει να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο αυτή την ε, κατάσταση η οποία θα κυριαρχεί στα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τέσσερις ζήτησαν τον λόγο και θα προτείνω να περιοριστούμε στα δύο λεπτά ώστε να ακούσουμε και την αρμόδια Γενική Διεύθυνση και τον εισηγητή μα ώστε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Κυρία Σαντέρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον εισηγητή για την εργασία που έκανε. Και εγώ θα ήθελα βεβαίως να χαιρετήσω αυτό το κείμενο που έρχεται όταν έχουμε βαθιές αλλαγές στην αγορά εργασίας. Οπότε εμείς θα πρέπει να αντιδράσουμε, θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε και να ξεχρονίσουμε τα κείμενα και αυτό βεβαίω είναι σύμφωνα είναι σύμφωνο με τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Στόχος μας είναι να προσδώσουμε μεγαλύτερη σταθερότητα στους εργαζομένους. Εγώ θα ήθελα να επιμείνω στην ανάγκη οι διατάξεις που θα θεσπίσουμε να εφαρμόζονται πλήρως σε εθνικό επίπεδο και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και ιδιαίτερα όσον αφορά την πραγματικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορά την τεράστια πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Μιλήσαμε για κάποιε πληροφορίε οι οποίε θα πρέπει να παρέχονται σε συγκεκριμένο σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτέ οι πληροφορίε βεβαίω θα πρέπει να παρέχονται στου εργαζομένου, δεν υπάρχει μια αμφιβολία. Αντίθετα θεωρώ ότι για να είμαστε πιο ρεαλιστέ, θα έπρεπε να θεσπίσουμε μία διαφοροποίηση μεταξύ αυτών των πληροφοριών που παρέχονται άμεσα και αυτών που θα πρέπει να παρέχονται στη συνέχεια και να υπάρχει μια προθεσμία μεταξύ μια ημέρα ή μια εβδομάδα, δύο εβδομάδων ενδεχομένω, ώστε να έχουμε κάποια ευελιξία. Πάντω, ε, συμφωνώ για, με του ανθρώπου για αυτά που υπόθηκαν για το κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καταρχάς, να αναφέρω κάτι που είπαν και άλλοι. Η νομοθεσία αυτή είναι προοδευτική, το οποίο σημαίνει ότι οι μελλοντικοί εργαζόμενοι στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας θα έχουν καλύτερη ζωή στο μέλλον από ό,τι έχουν τώρα. Και αυτό είναι καλό. Όμως, η πρόταση παρόλα αυτά μπορεί να βελτιωθεί και δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Να πω μόνο συνοπτικά ότι θα πρέπει να καλύπτουμε και το δημόσιο και το ιδιωτικό τομέα. Το δημόσιο δεν θα πρέπει να εξαιρείται. Και βεβαίως θα πρέπει να περιλάβουμε και τους αυταπασχολούμενους. για τους ορομίστους και τις συμβάσεις μηδενικών ορών. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να απογορευτούν, να καταργηθούν, όμως υπάρχουν και αλλού, όπως στη Νέα Ζηλανδία, όπου είχαν ένα επιτυχές παράδειγμα για το πώς εφαρμόζονται αυτές οι συμβάσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια αυτό το μοντέλο θα μπορούσε να μεταφερθεί και να ισχύσει σε αυτή την νομοθεσία. Εγώ θα έλεγα θα έπρεπε. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Ενρίκε που είπε ότι θέλει να ακούσει και να είναι ευέλικτο για την εξέβρεση λύσεων. Και με την συζήτηση που προηγήθηκε νομίζω ότι ε, υπάρχουν θέματα από των οποίων συμφωνούμε και είναι πολλά αυτά. σε ό,τι αφορά τον ορισμό, αν θα πρέπει να είναι ε, διευρυμένος ορισμός ή αν θα πρέπει να ε, είναι πιο ομοιογενοποιημένος, εναρμονισμένος. Υπάρχει η απόφαση του ε, δικαστηρίου ε, που αναφέρθηκε, αλλά εκεί λέει ότι θα πρέπει ε, να μην προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά σε εθνικό επίπεδο. Δεν υπάρχει ουσιαστικά ένας ευνίος ορισμός. Το θέμα είναι οι απολαβές, οι απερορίε. Οι δοκιμαστικές περίοδοι δεν μπορεί να είναι τρεις, έξι μήνες. Δεν έχουμε ε, ξεκαθαρίσει ακόμη. Πρέπει να μιλήσουμε όμως ε, για την ε, δοκιμαστική περίοδο και να πούμε ότι δεν μπορεί να παρατείνεται επαόριστον γιατί αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά δεν έχουν κάποια σχέση σταθερής απασχόλησης και καμία πρόπτικη και αυτό είναι απαράδεκτο, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν από αυτού. Ε, κάτι άλλο που θεωρώ σημαντικό είναι ε, ότι πράγματι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τεθούν υπό αμφισβήτηση οι συλλογικέ συμβάσει εργασία, οι κοινωνικοί εταίρ και τα δικαιώματά του. Ε, έχουμε εμπειρία, όχι βέβαια σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την ίδια εμπειρία γιατί υπάρχουν διαφορέ και ιδιαιτερότητε. Όμω σίγουρα υπάρχουν οι συλλογικέ συμβάσει που είναι η βάση και από εκεί πρέπει να βγουν οι ε, διάφορε ρυθμίσει. Τα δικαιώματα των κοινωνικών εταίρων σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να τα απεμπολίσουν και επίσης καλό είναι να λάβουμε υπόψη μας και τις νέες τεχνολογίες, αυτές οι ε, συμβάσεις μηδανικών ορών κτλ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία διαφωνία μεταξύ μας, αλλά είναι κάποιες χώρες οποίες υπάρχουν ακόμη αυτές οι συμβάσεις ε, και πρέπει να βρεθεί μια λύση, γιατί δεν μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ κύριε Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Πολλά υπόθηκαν. Αλλά και η κυρία Ουλσκοκ έχει να κάνει μια σημαντική δήλωση την οποία βέβαια αντικαθιστώ και εγώ είμαι συμπατριώτης σας από την Έμβη. Λέει λοιπόν κύριε Λοφσκό ότι η πρόταση αυτή είναι πολύ σημαντική και το ανέφερα πολύ σήμερα. Η αγορά εργασία ήδη έχει αλλάξει πολύ μετά από την υιοθέτηση προσφάτων οδηγιών που οδήγησαν σε αυτή την αθεώρηση της οδηγίας. Θεωρώ λοιπόν ότι με αυτή την οδηγία νέε μορφές μπορούν να ρυθμιστούν. Παρ' όλα αυτά, οι αναλύσει των οργανώσεων εργοδοτών και συνδικάτων από τη Σουηδία είναι ξεκάθαρη ότι υπάρχει ένα σαφή κίνδυνο ότι η πρόταση τη Κομισιόν θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στι βασικέ αρχέ του Σουηδικού μοντέλου συλλογικών συμβάσεων και θα επηρεάσει σοβαρά την ισορροπία μεταξύ κοινωνικών εταίρων και το δικαίωμα αυτορύθμιση. Και αυτό προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Υπάρχουν κυρίως τρία σημεία τα οποία θα ήθελα να τονίσω. Πρώτον, ο ορισμός των εργαζομένων, οι εργασιακές σχέσεις και οι εργοδότες. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την τωρινή ισορροπία όπου η έννοια του εργοδότη καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο μέσω της νομολογίας του δικαστηρίου όπως ακριβώς ισχύει σήμερα. Ο ορισμός λοιπόν του εργαζόμενου σχετίζεται άμεσα με τις ίδιες παραδόσεις και νομικά συστήματα της κάθε χώρας και σε εθνικό ακριβώς επίπεδο έχουν συγκροτηθεί αυτά τα εθνικά εργασιακά μοντέλα τα οποία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν με το βέλτιστο τρόπο και πολλοί συνάδελφοι τον έπαιξαν αυτό σήμερα. Επίση, η συγκεκριμένη πρόταση για τον ορισμό έχει επιπτώσει οι οποίε δεν θα μπορούσαν να αναθεωρηθούν υπό την εθνική νομοθεσία. Που κατ' επέκταση αυτό θα μπορούσε να έχει σημαντικέ επιπτώσει σε άλλε μορφέ νομοθεσία όπω ε, κοινωνική πρόνοια και φορολογία. Δύο, η αυτονομία των κοινωνικών εταίρων θα πρέπει να τηρείται. Επ' αυτού θα ήθελα να καλωσορίσω κάποιε από τι προτάσει που έκανε ο εισηγητή για την ενίσχυση τη εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων. Αλλά χρειάζονται περισσότερε ουσιώδει αλλαγέ, ιδιαίτερα στο άρθρο 12. Τρίτον, είναι εξίσου σημαντικό το, κοινωνικό το δίκαιο μέσω εξωτερικών συμβάσεων να διαμορφώνεται και από τι εθνικέ νομοθεσίε. Καταλήγοντα, θα έλεγα ότι εμεί σχεδιάζουμε και η Μαρίτα, η συναδελφό μου, σχεδιάζει να καταθέσει πολλέ τροπολογίε για αυτό το θέμα, για του λόγου που σα ανέφερα. Και θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα αυτό για μα στην Σουηδία. Πρέπει λοιπόν να είναι σεβαστά τα εθνικά μοντέλα Αγορά εργασία και να στηρίζεται η αυτονομία των κοινωνικών εταίρων. Από τη Γενική Διεύθυνση, παρακαλώ, σύντομα εσεί. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και από πλευρά Κομισιόν τόσο τον εισηγητή όσο και του κοιόδη εισηγητέ και όλου όσου έλαβαν το λόγο. Είναι πολύ επικοδομητική συζήτηση και βλέπω ότι ήδη έχετε αναλύσει σε βάθο την πρόταση αυτή. Δεν θα επαναλάβω γιατί είναι τόσο σημαντικό για την Κομισιόν, το είπαν όμω και οι ομιλητέ, ούτως ή άλλως ε, με εύκολο τρόπο. Θέλω να αναφερθώ σε ορισμένα ζητήματα και κάποιες απορίες σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν. Το εύρος της πρότασης και ο ορισμός του άρθρου 2 για τον εργαζόμενο. Είπαν και πολλοί ομιλητές ότι αυξάνεται ε, η ευαλωτότητα για πολλούς ε, και ιδίω αυτού που αποκλείονται την αγορά εργασία και από το καθεστώ εργαζομένων. Αυτό το βλέπουμε στην εργατική οικονομία, στην αλληλέγγυη οικονομία, σε κάποιε άλλε μορφέ εργασία, ε, μερική απασχόληση, ε, με κουπόνια κτλ. Και πραγματικά πρέπει να δούμε κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια που φε, λέγει, αναφέρει απόφαση του δικαστηρίου και δικαιούνται προστασία δυνάμει αυτή τη οδηγία. Προστατεύει και τους εργαζόμενους από μελλοντικές ε, εξελίξεις στον τομέα της αγοράς εργασίας. Ο ορισμός κωδικοποιεί, όπως είπαν και οι προλήσαντες, την έννοια του εργαζόμενου που χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί ε, τα τελευταία 30 χρόνια το δικαστήριο για τον οικονομικά ενεργό πολίτη που έχει καθώς ε, απασχολουμένο. Είναι κάτι που εφαρμόστηκε στα εθνικά συστήματα ως ορισμό. Και για τον κύριο και να πω ότι δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι ένα κάτω μέλος θα πρέπει να αλλάξει τους δικούς του ορισμούς. Αφορά συγκεκριμένα το πεδίο εφαρμογή αυτή τη οδηγία ορισμό αυτό. Άρα, ένα κάτω μέλο μπορεί να πει αυτή η οδηγία, σε ό,τι αφορά το ψυχικό πεδίο εφαρμογή, ε, έχει να κάνει με τον κοινωνικό εργασιακό κώδικα, οργατικό κώδικα, πώς ορίζει τους εργαζόμενους ε, και τους εγχώρεους, ε, τους εργαζόμενους ε, διαφόρων κατηγοριών να τους καλύψει. Και η επικαλύψη σε θέματα φορολογικά κοινωνική ασφάλειας είναι κάτι που έτσι θα αποφευχθεί. Πάντα στο παιδί εφαρμογή. Συμφωνούμε με αυτού που ανησυχούν πω υπάρχουν δηλαδή να εξαιρείται ο δημόσιος τομέας ή η ναυτική για παράδειγμα. Εμείς θεωρούμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να υπόκειται στην προστασία αυτή θα πρέπει να υπάρχουν ολιγμένοι αντικειμενικοί λόγοι και οι καταστάσει αυτέ και οι συνθήκε θα πρέπει να δικαιολογούνται με αντικειμενικού λόγου. Ε, ο χρονισμός της πληροφοριών είναι θέμα θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Πρέπει να γνωρίζουν ποιε είναι οι συνθήκε, ποιοι είναι οι όροι απασχόληση του εργαζόμενοι και από πότε ξεκινούν τα δικαιώματά του. Αυτό το έχουν προσυπογράψει όλε οι χώρε και στο πλαίσιο του κοινωνικού πυλώνα και θα εφαρμοστεί με το, την οδηγία αυτή στην πράξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει και στην έκθεση του Κοινοβουλίου να υπάρξει υποστήριξη για την διάθεση ευθύ εξ αρχή από την έναρξη τη επαγγελματική σχέση των βασικών πληροφοριών. Και να μην υπάρχει καθυστέρηση στην παροχή αυτών των πληροφοριών. Καταλαβαίνω το ερώτημα. Αν θα πρέπει ήδη από την πρώτη μέρα παρέχονται όλε τι πληροφορίε ε, του καταλόγου. Αυτό το καταλαβαίνω. Και για το θέμα των κοινωνικών εταίρων, αναγνωρίζουμε τον πολύ σημαντικό του ρόλο σε πολλά κράτη-μέλη για τη ρυθμίση τη αγορά εργασία εξού Ήδη η πρόταση δίνει περιθώρια στους κοινωνικούς εταίρους για να μπορούν να τροποποιούν τα υλικά δικαιώματα του κεφαλαίου 3 στις ανάγκες των τομέων αυτό. Μεγάλο το πεδίο. Το ίδιο και για την εφαρμογή της οδηγίας μέσω συλλογικών συμβάσεων. Το θέμα είναι να υπάρχει θέση προστασία στον αυξανόμενο αριθμό που δεν καλύπτονται από τις ε, Συλλογικέ συμβάσεις που δεν είναι συνδικαλισμένοι. Αν τα ελάχιστα πρότυπα των Ευρωπαίων Ομοθετών εφαρμοστούν με συλλογικές ή εφαρμόζονται με συλλογικές συμβάσεις, θα πρέπει να είναι δυνατόν επίσης να ελέγχεται ότι διατηρούνται αυτά τα πρότυπα και κανόνε. κανόνες. Και αυτό θα πρέπει να υπόκειται στις εθνικέ και στην ευρωπαϊκή δικαιοδοσία. Άρα συμφωνώ και εγώ το αίτημα του συγκριτού και των σκιωδών να συνεχιστεί αυτή η πολύ οικοδομική συζήτηση. για εργαζομένους που πολύ μεγάλος αριθμός αυτών είναι σε πολύ δύσκολη επισφαλή θέση. Και εμείς φυσικά και θέλουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σας ε, στο πλαίσιο και αυτού του φιλόδοξου παρόλα αυτά χρονοδιαγράμματο. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα ο εισηγητή να πει δύο λόγια. Ναι, Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται μισή ώρα να εξηγήσω τώρα τις απαντήσεις μου. Λοιπόν, υπάρχουν Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστώ πολύ και είμαι αισιόδοξο γιατί βλέπω όλα όσα άκουσα είναι επικοδομητικά και όλοι πιστεύουν ότι μπορεί να προχωρήσει. Όποιο θέλει μπορεί και με αυτό κερδίζουμε ήδη πολλά. Υπάρχουν πολλά θέματα, πολύ συγκεκριμένα που αναφέρθηκαν και είναι σημαντικά. Δεν αμφιβάλλω ότι μπορούμε να βρούμε την ε, κατάλληλη ισορροπία. Πριν το σχάρι αναφέρθηκαν ε, ιδιαίτερε δυσκολίε των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ. Τι έχω λάβει υπόψη. Μπορώ φυσικά και παραπάνω. Επίση, άλλα θέματα για πρώτη μέρα ή όχι την πρώτη μέρα, ανάλογα με τι θα το συζητήσουμε αυτό και θα βρούμε ισορροπία. Πόσο καιρό θα διαρκεί η κατάρτιση να βρούμε μια ισορροπία και σε αυτό ίσως θα έχουμε ε, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Θα τα δούμε όλα αυτά τα θέματα με τις συναντήσεις με τους σκιώδεις. Φυσικά τους εμπιστεύομαι και σίγουρα θα φτάσουμε σε συμφωνία. Τώρα, πιο κεντρικά ζητήματα. Το θέμα του ορισμού, το περιβόητο. Χάρηκα πολύ όπως άκουσα από τον κύριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φοβάμαι ότι μετατρέπουμε ένα πρόβλημα και αγγίζουμε ε, το καυτό σημείο των νομοθετών των δικηγόρων. Μετατρέπουμε λοιπόν ένα κοινωνικό θέμα σε ένα θέμα ε, με, σύγκρισης ε, νομοτεχνικής για να επιβάλλουμε στους ε, εθνικούς ε, κώδικες ένα συγκεκριμένο ορισμό που θα έχει συγκεκριμένη νομική αξία, αυτό δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Επομένως, ε, αυτό που υπόθηκε ότι αφορά μόνο την πρόταση, δηλαδή ορίζεται ο εργαζόμενος μόνο για αυτή την πρόταση, ίσως θα πρέπει να αποφύγουμε τον, τη λέξη ορισμός αλλά να πούμε ότι αυτή η πρόταση θίγει οποιοδήποτε άτομο που έχει μία σχέση εξάρτησης οικονομική κτλ. Τώρα, για τις ε, συμβάσεις μηδενικών νερών. Δεν υπάρχει στην Ισπανία δεν είναι πρόβλημα. Αν το αποφασίσει το Κοινοβούλιο ε, θα καταργηθεί. Αν ε, και άκουσα ότι είπε ο συνάδελφος Σάιμον, δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι το κατάλληλο πλαίσιο για να απαγορεύσουμε αυτές τις συμβάσεις. Αντίθετα, κάνουμε μία σειρά πραγμάτων ε, για να υποχρεώσουμε κάποιους να σεβαστούν. Λοιπόν, τώρα για το δημόσιο τομέα. Ένα είναι όσοι εργάζονται για το δημόσιο ή για δημόσιες εταιρείε που δεν ε, μπορούν να θεωρηθούν κάτι ξεχωριστό και είναι κάτι διαφορετικό ε, η άμυνα και οι δυνάμεις ασφαλείας. Αυτό θα τα δούμε. Και έχουμε και το πρόβλημα της Σουηδίας. Πριν 15 μέρες εγώ πήγα στη Στοκχόλμη και μάλιστα συνάντησα μέχρι και την Υπουργό Απασχόληση και κανένας δεν μου μίλησε για αυτή την κίτρινη κάρτα. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι από τότε, 18 Μαρτίου μας εστάλει αυτό, εξελίσσονται τα πράγματα παντού. Κανένας ε, δεν μου μίλησε για την κίτρινη κάρτα. Υπήρχε ένας κύριος ε, μάλιστα που εκπροσωπούσε του κοινωνικού εταίρου και μου είπε ότι εγώ δολοφονούσα το κοινωνικό μοντέλο, ενώ εγώ είμαι θαυμαστής αυτού του μοντέλου. Λοιπόν, εγώ θα βάλω τα δυνατά μου έτσι ώστε να τους ξεκαθαριστεί ότι ενισχύουμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα αναπτυχθούν και θα ελέγξουν και θα εφαρμόσουν την νομοθεσία, δηλαδή αυτοί είναι που θα δημιουργήσουν την νομοθεσία. Μόνο μη μου ζητήσετε το δικαίωμα ε, να μπορούν να διαπραγματευτούν κάτω από τα ελάχιστα πρότυπα. Εγώ έτσι λοιπόν πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα γίνει και επομένως θα βρούμε μια λύση. Σας ευχαριστώ. Σε σχέση τώρα με το χρονοδιάγραμμα προθεσμία για τις τροπολογίες 26 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι και θα εξετάσουμε τις τροπολογίες 29-30 Αυγούστου η ψηφοφορία θα γίνει στις 18 Οκτωβρίου του 2018 στην Επιτροπή μας. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν στο σημείο 8 της ημερική διάταξη που αφορά το Πανευρωπαϊκό Ατομικό Συνταξιδικό Προϊόν και προτείνω να δώσουμε αμέσως το λόγο στο Heinz Μπέκερ από το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Thank you very much, uh, Chair. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω όλους ε, ε, για την πολύ καλή συνεργασία, τους κοιόδης εισηγητές ε, και την γραμματεία για την εξωτερική υποστήριξη. Ήταν μια πολύ επικοδομητική διαδικασία μέχρι τώρα. Είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι το Πανευρωπαϊκό Τομικό Συνταξιδοτικό Προϊόν το ΠΕΠ θα ε, αποτελέσει μια θεματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα θεματικό επίτευγμα. Δεν υπάρχει συγκρίσιμο προϊόν με αυτό. Και με ελέγχεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμπεριλαμβανομένης ε, και της επιλογής ε, ευρωπαϊκής εγγύησης κεφαλαίου που να ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω του ΕΙΟΠΑ, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα λοιπόν αυτό και δεν ε, έχει υπάρξει ποτέ στη συνταξιδοτική αγορά. Εμείς ως Επιτροπή Απασχόλησης δεχόμενοι ότι η αρμόδια επιτροπή είναι η ΕΚΟΝ και συμμετέχει και η ΙΜΚΟ με γνωμοδότηση. Όλες ε, οι πτυχές ε, των χρηματοοικονομικών αγορών και των αγορών ασφαλίσεων ε, θα είναι αντικείμενο εκείνων των επιτροπών. Εμείς λοιπόν επικεντρωνόμαστε στη σκοπιά της απασχόλησης και στη διάσταση της κοινωνικής πολιτικής. να εξηγήσω ότι έχουμε δύο ε, κυρίες ομάδες στόχου. Καταρχήν ε, θα είναι αυτοί που θέλουν ε, να έχουν μία πρόσθετη ε, διασφάλιση μετά τη συνταξιδότηση σε σχέση με την ποιότητα ζωής τους οι υπόλοιποι. Και νομίζω ότι επίση είναι σημαντική. Είναι αυτοί που ζουν σε χώρες όπου δεν είναι καλά αναπτυγμένος ο πρώτος και δεύτερος πυλώνας των συντάξεων. Αν ε, δεν ε, υπάρχει ένα καλά αναπτυγμένο σύστημα, τότε αυτό το προϊόν μπορεί να είναι μια πολύ καλή επιλογή για το μέλλον, για να υποστηριχθούν κυρίως οι νέοι και οι γυναίκες. Το ΠΕΠ ε, θα συνεισφέρει στο να καλύψει τις ανάγκες ανθρώπων ε, που θέλουν ε, να έχουν ε, επαρκείς συντάξεις θα αντιμετωπιστεί το δημογραφικό πρόβλημα και τα εφιστάμενα στα εξοδοτικά κενά. Επίσης, συμπεριλαμβάνουμε μία πτυχή μακροπρόθεσμης αποταμίευσης για το ΠΕΠ και μία βιώσιμη επενδυτική πολιτική συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών επενδύσεων. Το ΠΕΠ έχει σχεδιαστεί ως ένα κινητό προϊόν, δηλαδή ε, να εξυπηρετεί ανθρώπους που μετακινούνται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, που εργάζονται ή ζουν εκεί και συμπεριλαμβάνουμε πολλές ε, πτυχές ε, στο να διαφυλάξουμε στην κινητικότητα αυτή καθ' αυτή. Αν ο πάροχος του εξωτερικού προϊόντος, ΠΕΠ, δεν παρέχει ένα ε, προϊόν στην νέα χώρα, ο αποταμιευτής ΠΕΠ μπορεί να αποφασίσει από μόνος του ποιον ε, νέο πάροχο θα διαλέξει στην καινούργια χώρα. Και όλα αυτά θα πρέπει να είναι δωρεάν. Υπάρχουν ε, διάφορες πληροφορίες που θα είναι υποχρεωτικές, παραδείγματος χάρη, μία δήλωση των συνταξιδοτικών παροχών, που, όπου αναφέρονται όλες οι υποχρεώσεις ε, και επίσης και το τι εννοούμε με τη συμπληρωματική σύνταξη. Το ΠΕΠ επίσης, όπως είπα, θα συμπεριλαμβάνει περιβαλλοντικό, κοινωνικό παράγοντα και παράγοντα διακυβέρνησης και επίσης ε, θα πρέπει να διατίθεται και μία αξιολόγηση κινδύνου στην ΕΙΟΠΑ ε, στις αρμόδιες αρχές καθώς και στους ε, αποτεμιευτές ε, θα πρέπει να αναφέρονται όλες οι πιθανές συνέπειες. Υπάρχει και μια σημαντική πτυχή, η βασική επενδυτική επιλογή. Συχνά αυτό σημαίνει ότι υπάρχει προστασία του κεφαλαίου για το πανευρωπαϊκό τομικό συνταξιδοτικό προϊόν. Έχουμε συμπεριλάβει τον κανονισμό ότι η ενημέρωση για τον αποταμιευτή ΠΕΠ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις σχετικές πτυχές ε, με πάσα λεπτομέρεια και μπορεί να χρειαστούν περισσότεροι συμβιβασμοί γιατί αυτές οι πληροφορίες ε, συμπεριλαμβάνονται ε, στο λεγόμενο βασικό έγγραφο πληροφοριών ΠΕΠ, έτσι δηλαδή μπορεί να έχουμε ε, παραπάνω από ε, μια συμβιβαστική λύση γι' αυτό. Αλλά έχουμε ήδη ένα συμβιβασμό. Και τέλος, θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα ευχάριστο ότι έχουμε συμφωνήσει να κάνουμε την εξή πρόταση. Οι να πρέπει να εγγυώνται στον αποταμιευτή ΠΕΠ ε, ότι το κεφάλαιο που θα έχει συσσωρευτεί μέχρι την αρχή της περίοδου ε, πληρωμών θα είναι ίσο με το ποσό των εισφορών που έχουν καταβληθεί συμπεριλαμβανομένου όλου του κόστους ε, συν το κόστος του πληθωρισμού που το υπολογίζουμε ως ένα ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού του 4%. Δεν υπάρχει κανένα άλλο συντοξιδοτικό προϊόν στην αγορά ακόμη και θα μπορούσε, όπως είπα, να αποτελεί ένα πολύ καλό ευρωπαϊκό προϊόν ναυαρχίδα. Έχουμε ε, περίπου 25-30 συμβιβασμούς και πολλές τροπολογίες. Η ΥΜΚΟ σήμερα ψηφίζει η ΕΜΠΛΕ ψηφίζει στις 28 Ιουνίου και η ΕΚΟΝ στις 11 Ιουλίου έτσι ώστε να μπορούμε να το συζητήσουμε στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστώ όλους για το επικοινωνικό έργο. Θα δώσω τώρα το λόγο στου. συνάδελφου που το λόγο, αλλά πάρα πολύ σύντομη να είστε παρακαλώ ένα λεπτό, γιατί έρχεται ο κύριος ε, Κατάινεν όπου να είναι και ζητώ συγγνώμη που θα πρέπει να σας ζητήσω να είστε τόσο σύντομοι. Για τους σοσιαλιστέ, ε, υπάρχει κάποιο, Α, ωραία, γλιτώσαμε ένα λεπτό. Για την ομάδα ECR, Μάκιν Μάκιντάιρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη σκιώδης εκτίση τον κύριο Γκέρι και δεν μπορούσα να είναι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω εξ ονόματό του τον κύριο Μπέκερ για το έργο του. Εγώ προσωπικά είμαι οπαδό ε, των ε, συντάξεων αυτών ε, και καλό είναι να υπάρχει κάποια πρόταση. Το είχα πει και στην προηγούμενη συζήτηση. Στηρίζουμε σε μεγάλο βαθμό αυτή τη γνωμοδότηση. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι οποιοδήποτε τέτοιο προϊόν να είναι συμπληρωματικό και να μην εναρμονεί στα εφιστάμενα στα εκδοτικά ζητήματα. Αυτό κάνει ο εισηγητή ε, και γι' αυτό στηρίζουμε το σχέδιο των συμβαστικών προτάσεων. Ίσως να έχουμε κάποια θεματάκια με ένα-δύο πράγματα που νομίζουμε ότι υπερβαίνουν το πεδίο αρμοδιοτήτων τη Επιτροπή μα. Θα βράζω με τη ευκαιρία ε, να ζητήσω να στηρίξετε τη δική μου τροπολογία που δεν έχει περιληφθεί σε μία συμβιβαστική τροπολογία, την υπαρθμόν 63. Ειδικά δε αυτό που θέλουν να μειωθούν τα έξοδα, το κόστος προς τον καταναλωτή. Σε σχέση με οποιοδήποτε τέτοιο προσωπικό στέξοδοτικό πρόγραμμα, που μπορεί να είναι μια πραγματική λύση στην Ευρώπη, αλλά υπάρχουν και κάποια αντικίνητρα, ένα από τα οποία είναι το πρόσθετο κόστος που θα μπορούσε να αποτελέσει δυνητικά αντικίνητρο. Αν αυτό το λύσουμε, θα έχουμε ένα πολύ καλό προϊόν. Ευχαριστώ. κύριος Καλβέ Σαμπών για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα τα πω γαλλικά για να τα πω πιο γρήγορα. Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους, ε, κυρίως ε, τον εισηγητή, τον ε, κύριο Μπέκερ. Όλοι επίσης ήμασταν υποδομητικοί και πετύχαμε σημαντικά πράγματα που θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε. Πρώτον, πολύ σημαντικό, Default Investment Option, η προεπιλογή, επενδυτικής επιλογής. στους ε, ευάλωτους ταξιούχους να μπορούν να κτίσουν το κεφάλαιό τους ε, σε περίπτωση πτώχευσης. Δεύτερο, δεν θα θέλαμε να υπάρχει επίδυση, να υπάρχουν επίδυση σε παράγωγα και άλλα τέτοια ε, προϊόντα με μεγάλο ρίσκο. Θέλουμε επίσης εγγύηση ε, κατά ε, μόνιμης αναπηρίας θανάτου στην φάση της συσσόρευσης κεφαλαίου για τα επενδυτικά πρότυπα. Και επίσης στηρίζουμε το άρθρο 5, τους πρασίνους, S&D το άρθρο 10 κτλ. Σημαντικό να μπει η προσέγγιση της εταιρικής σχέσης. Αλλιώς Περισσότερε από τι μεγάλε εθνικέ ασφαλιστικέ εταιρείε δεν θα μπορέσουν να θέσουν στο εμπόριο αυτά τα προϊόντα, εάν του ζητηθεί να έχουν, παραδείγματο χάρη, γραφείο σε κάθε χώρα. Μόνο η BlackRock και άλλοι τέτοιοι μεγάλοι όμιλοι μπορούν να το πετύχουν. Εμείς θα στηρίξουμε ένα σύστημα εταιρική σχέση όπως και ο κύριο ε, Μπέκε και έτσι θα έχουμε κάτι απτό και πολύ καλό για τους Ευρωπαίους πολίτες. Καλωσορίζουμε τους ε, προσκεκριμένους κυρίας Μελέν που μόλις ήρθα. Εσείς από την ε, Γκουε, κυρία Κάρικ. Øh, Ευχαριστώ. Αντικαθιστώ το συνάδελφό μου που δεν μπορούσε να είναι εδώ θα μιλήσω για τα σημαντικότερα. Το πανευρωπαϊκό στεξιδοτικό προϊόν είναι μια προσπάθεια προώθησης ε, της ιδιωτικής σύνταξης. Τα στεξιδοτικά συστήματα δηλαδή ε, πλέον μεταφέρονται, ε, μετατοπίζονται σε μια χρηματοπιστωτική αγορά ουσιαστικά. Όμως θα έπρεπε να ενισχυθεί και η απασχόληση και η ασφάλιση των εργαζομένων από τα κράτη. Γι' αυτό και δεν μας ε, φαίνεται σωστή η πρόταση της Κομισιόν. Αυτή η ιδιωτική σύνταξη που θα στηρίζει τα έσοδα των χρηματιστήρων δεν είναι μια καλή λύση για τους συνταξιούχους. Γι' αυτό πρέπει να στηριχθούν τροπολογίες που υποστηρίζουν δημόσιες κρατικές συντάξεις. Τα κρατικά συνταξιωτικά στήματα έχουν πρόβλημα. Γιατί όμως? γιατί είναι τέτοιες οι συγκυρίες και υπάρχουν και αυτά τα νέα καθεστώτα, υπάρχει παρεκονομία, απλήρωτη, αδήλωτη εργασία, ανεργία κτλ. Είμαστε κατά των προτάσεων που θα έδωσαν στους διαχειριστές κεφαλαίων τη δυνατότητα να κερδοσκοπούν με τις αποταμιεύσεις των συνταξιούχων. Είναι ένα γκρίζο προϊόν που ουσιαστικά αποφέρει κέρδη στις παγκόσμιες αγορές. Δεν είναι συνταξιδοτικό προϊόν και βάζουμε σε κίνδυνο δισεκατομμύρια με αυτό του είδους τα προϊόντα. Δεν βλέπω να εκπροσωπούνται άλλες πολιτικές ομάδες. Η κυρία Μελέν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι. Επειδή ε, δεν έχουμε ε, και πολύ δυνατότητα δεν μπόρεσε να περιληφθεί καμία από τις τροπολογίες μας συμβασικές προτάσεις. Ε, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αυτό το έγγραφο ε, ουσιαστικά ε, θα έχει boomerang, ε, θα αποτελέσει ένα boomerang γιατί ουσιαστικά επηρεάζει και ε, τα εθνικά δίκαια, παρεμβαίνει στην εθνική νομοθεσία. Το ίδιο, η ίδια κατασκευή του ε, κάνει το προϊόν αυτό να μην είναι επωφελές για αυτούς που θέλουμε να βοηθήσουμε. Είναι επισφαλές, δεν δημιουργεί παραπάνω οικονομίες και αποταμιευσή. Επίση ε, θα είναι ανταγωνιστικό αυτό το προϊόν και η Ευρωπαϊκή Αρχή Επαγγελματικών των Συντάξεων δεν θα φροντίσει να καλύψει τους μικρούς ασφαλισμένους, αλλά τους μεγάλους ομίλους και συμφωνώ με τη συνάδελφο για γκρίζα ζώνη, γκρίζα προϊόντα. Σίγουρα τα εθνικά κοινωνικά δικαιώματα δέχονται πλήγμα και γι' αυτό έχουμε έντονες επιφυλάξεις. Γι' αυτό το κείμενο πραγματικά δεν είμαστε υπέρ, αν και ο συγκτής έκανε πολύ καλή δουλειά. Κυρία Ρέγνερ, ναι, είπα, θα είμαι σύντομη. Η Μαριά Ρενά ήταν η σκιώδη από την ομάδα μας. Δεν μπορούσε να είναι εδώ. Πάρα πολύ σύντομα λοιπόν φυσικά δεν είναι αντικατάσταση, υποκατάσταση του πρώτου και δεύτερου πυλών αυτό το ΠΕΠΑ σε καμία περίπτωση επομένως ε, από κάθε πλευρά αυτό πρέπει να το λέμε πανευρωπαϊκή προοπτική θετική αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει ε, επένδυση, επενδυτική επιλογή. Αυτό το πρόγραμμα ε, είναι συμπληρωματικό και σίγουρα ο πρώτος και ο δεύτερος πυλώνες σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δεχθούν πλήγμα από αυτό το προϊόν που είναι συμπληρωματικό και όχι υποκατάστατο. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Συγγνώμη, ζητώ και πάλι που σας ε, έβαλα να μιλήσετε για πολύ λίγο σε ό,τι αφορά τις ε, τροπολογίες. 2 ε, Μαΐου λέει ο 22 ε, Ιουνίου στην Επιτροπή ΕΚΟΝ 11 Ιουλίου Ολομέλεια δεν έχουμε ακόμη ημερομηνία. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο. Ανταλλαγή απόψε στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου με τον κύριο κατά είναι αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Για να μην καταχραστώ το χρόνο σας, να πω ότι πάντοτε είναι μια σημαντική στιγμή για εμάς η παρουσία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανταλλαγή αυτή απόψεων, για τον διαθρωμένο αυτό διάλογο. Σημαντικό ε, ορόσημο του διαλόγου ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Κατάινεν, καλώς ήρθατε. Θα σας δώσω λίγο χρόνο να καθίσετε. Ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα πόσο μας πιέζει ο χρόνος πολλές φορές. Θα σας δώσω ευθύ αμέσως το λόγο. Αν θέλετε, Δέκα λεπτά παρακαλώ. Mr. President, honorable members, ladies and gentlemen. Πρόεδρε, κύριε βουλευτές, και κύριοι, ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο για να μιλήσω για διάφορα ζητήματα και θα μιλήσω ιδιαίτερα για θέματα εργασιακά και εκπαίδευση με στόχο να καλύψουμε θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για το μέλλον για τις ε, κοινωνίες μας όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η γυριακή οικονομία. Αυτές είναι οι δύο μεγατάσεις στην οικονομία που θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο στις κοινωνίε μα και θα πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτέ τι αλλαγέ. Οι αλλαγέ βέβαια μπορούν να είναι θετικέ αλλά και αρνητικέ ανάλογα με το πόσο προετοιμασμένοι είμαστε και πόσο θα προβλέψουμε σωστά τι αλλαγέ αυτέ. Αν δούμε την τεχνητή νοημοσύνη και την ψηφιοποίηση, υπάρχουν διάφοροι υπολογισμοί, διάφορε εκτιμήσει για το πόσε θέσει εργασία θα χαθούν ανάλογα με το χρονισμό αν δούμε δηλαδή την πενταετία, θα έχουμε διαφορετικά στοιχεία σε σχέση με την δεκαπενταετία. Ακόμα και αν δούμε το θέμα βραχυπρόθεσμα, υπάρχει μεγάλη ποικιλία εκτιμήσεων. Όσα είχε υπολογίσει τελευταία ότι το 9% των υπαρχιστών θέσεων εργασία απελούνται από την αυτοματοποίηση είναι το μικρότερο ποσοστό που έχω δει, το 9%. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα αντικαταστηθεί ολόκληρη θέση εργασία, αλλά κομμάτια τη εργασία. Δηλαδή δεν θα χαθούν οι ίδιε οι θέσει τη εργασία από μόνε του. Αλλά θα πρέπει να προσέχουμε. Επίση, η ψηφιοποίηση και η τεχνική νοημοσύνη θα μπορούσε να οδηγήσει στην αντικατάσταση πολλών υποεργασιών που δεξάγονται από τους εργάτες. Δεν ξέρουμε όμως ακόμα τι θα γίνει ακριβώς, κάνουμε εκτιμήσεις και αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορούμε να προετοιμαστούμε για αυτές τις αλλαγές. Δεν έχει νόημα να προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε τα μελλοντικά επαγγέλματα επειδή δεν ξέραμε, δεν ξέραμε ποτέ. Αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε τους εργάτες να είναι πιο εύκολο προσάρμοστοι σε αυτές τις αλλαγές και να αποκτήσουν νέες δεξιοτεχνίες. Γι' αυτό ακριβώς ε, εγώ λέω βάσει αυτής της ανάλυσης ότι θα πρέπει να ανθαρρύνουμε τις χώρες μέλη σήμερα να ενισχύσουν την εκπαίδευση, ακόμα και την βασική εκπαίδευση, περισσότερο από ό,τι έκανα στο παρελθόν. Δεν μιλάω για τις και τα προσόντα. Στη συνέχεια θα το κάνω αυτό. Μιλάω για τη βασική εκπαίδευση και την κατάρτιση. Δυστυχώ η εκπαίδευση δεν αποτέλεσε τομέα προτεραιότητα σε πολλέ χώρε μέλη και αυτό θα το δείτε εύκολα από τα αποτελέσματα στο τομέα τη εκπαίδευση στι χώρε μέλη. Επίσης, αν δείτε και τις αρμοδιότητες ή τις δεξιότητες των διδασκόντων, υπάρχουν τεράστιες αποκλήσεις. Το 25% των ενηλίκων Ευρωπαίων έχουν σοβαρά ελλείμματα στην μόρφωση. Οπότε, τι μπορούμε να προσδοκάμε από ενήλικες, από άτομα, από πολίτες, αν δεν ξέρουν να γράψουν και να διαβάσουν σωστά. Αυτά σε σχέση με την εκπαίδευση. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι είμαι αρκετά ικανοποιημένο ότι καταφέραμε να στοχεύσουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο στα κοινωνικά θέματα και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση. Αυτή είναι η πρώτη χρονιά που αυξήσαμε σημαντικά τις συστάσεις και τις προσεγγίσεις για τα εκπαιδευτικά συστήματα στις χώρες μέλη. Όπω ξέρετε, δεν έχουμε αρμοδιότητα ω Ένωση στα θέματα εκπαίδευση. Δεν σημαίνει όμω αυτό ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για την εκπαίδευση αν δούμε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην εκπαίδευση και να θεωρούμε τι χώρε να κάνουμε μεταρρυθμίσει. Όπω ακριβώ κάναμε και για τα συνταξιδοτικά συστήματα στι διάφορε χώρε ή οτιδήποτε άλλο κοινωνικό θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να μας στηρίξετε στην αποστολή μας αυτή να περιλάβουμε την εκπαίδευση και να της δώσουμε ένα πιο ισχυρό ρόλο, μια πιο ισχυρή θέση στη δικασία του εξαμήνου. Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να εξετάσουμε και τις δεξιότητες, τα προσόντα των εργαζομένων. Ήδη ζούμε στην ψηφιακή εποχή και η ζήτηση για ψηφιακές δεξιότητες έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία και η τάση είναι αυξητική. Πάνω από 750.000 ε, θέσεις εργασίας καινές ε, αφορούν τον τομέα αυτό και καλύπτει την περίοδο μέχρι το 2020. Επίσης, οι ψηφιακές δεξιότητες ζητούνται πια ως προσόντα για όλες τις θέσεις εργασίας. Παρ' όλα αυτά, 4 στους 10 Ευρωπαίου σήμερα δεν έχουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Δεν χρειάζεται όμω βέβαια μόνο αυτό. Χρειάζονται δεξιότητες τεχνικές και ψηφιακέ, όπως και άλλε δεξιότητες, επιχειρηματικότητα, κριτική σκέψη κλπ. Για τα άτομα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουν την κατάρτιση τους διαδίου Γι' αυτό ακριβώ εμεί ω Κομισιόν επενδύουμε τόσο πολύ στι δεξιότητε. Έχουμε το θεματολόγιο που ξεκίνησε το 2016 για την ε, δεξιότητε στην Ευρώπη που αποβλέπει την ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων για όλου μα από το χαμηλότερο στο ψηλότερο επίπεδο Στοχεύοντα τι προσαρμογέ και στι τεχνικέ και τεχνολογικέ αλλαγέ. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν και απαραίτητα μέτρα που θα στηρίξουν αυτές τις δέκα δράσεις για, αυτές τις, ε, για αυτούς τους τομείς και θα μιλήσω στη συνέχεια για κάποιες πρωτοβουλίες. Οι ψηφιακές δεξιότητες και η βελτίωσή τους ήταν το κύριο κίνητρό μας όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασία και των κύριων δράσεων σε αυτό το θεματολόγιο. Από το 16 λοιπόν το Δεκεμβρίου. Έχουμε 21 εθνικά κέντρα και το πιο πρόσφατο ήταν ένα κέντρο μεταξύ Σουηδίας, Κατοχωρών και Ελλάδας. Οι κυβερνήσεις δεν είναι μόνες οι οποίες πρέπει να δράσουν. Έχουμε και πρωτοβουλίες από κοινωνικούς εταίρους, από επιχειρήσεις λοιπά για την παροχή αυτών των ψηφιακών δεξιοτήτων. Έχουμε δει παραδείγματα στο Βέλγιο όπου είχαμε αριστούχους σε αυτές τις ε, πρωτοβουλίες με την παροχή αυτών δεξιοτήτων στα παιδιά. Έχουμε ένα παραδειγματικό ένα υποδηματικό πρόγραμμα στην ε, Ιρλανδία για να, για να βελτιωθούν οι δεξιότητες αυτές με, που βοήθησε μάλλον 12.500 άνεργους. Προσπαθούμε λοιπόν να ευκολύνουμε τις χώρες μέλη στο να βελτιώσουν τις δεξιότητες των εργαζομένων και γι' αυτό ακριβώς ε, είχαμε την σύσταση ε, φέτος για την ε, διαβίου μάθηση και το πλαίσιο το οποίο θετήθηκε το αντίστοιχο στις χώρες μέλη. Έχουμε επίση και το θέμα των τομεακών δεξιοτήτων. Το οποίο σημαίνει ότι συγκεκριμένοι οικονομικοί τομεί χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή ακριβώς για να καλυφθούν αυτές οι ελλείψεις που υπάρχουν σε δεξιότητε. και καλύψαμε ήδη από πέρσι μίσο όπως μηχανία, τουρισμό, θάλασσες μεταφορές κλπ. Έχουμε ένα δεύτερο κύμα προγραμμάτων το οποίο θα ξεκινήσει στο τέλος του τρέχοντος έτους, θα καλύψει την μεταποίηση, οικοδομές, ε, χάλιβα, ναυτιλία και οι χώρες μελή πρέπει να πούμε ότι έχουν δεσμευτεί για μέτρα τα οποία θα αυξήσουν ακριβώς αυτές τις δεξιότητες μέχρι το 2020. Η Κομισιόν κάλεσε τις χώρες μέλη να το κάνουν αυτό μέχρι το, τα μέσα του Ιούλη. Βοηθάμε και τους ανειδίκευτους να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, τις, τη βασική τους μόρφωση, ώστε να τους βοηθήσουμε να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Κύριοι βουλευτές, τα κονδύλια και τα μία της Ένωσης ε, θα διαδραματώσουν ένα κέριο ρόλο επίσης στην ε, στήριξη αυτού του πυλώνα. Πρέπει να επενδύσουμε στους πολίτες μας ώστε όλοι οι πολίτες μας να έχουν τα κατάλληλα προσόντα για την αγορά εργασίας στο μέλλον. Έχουμε στο επόμενο πι δελτα πι με 101 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε και τι προτεραιότητες του αντίστοιχου πυλώνα, τις οποίες θα εποπτεύουμε πολύ προσεκτικά σε σχέση με τις δραστηριότητε του εξαμήνου. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε όλε τι δράσει οι οποίε απολέπουν ακριβώ τη βελτίωση όλων των προσεωτήτων, κυρίω των ε, τεχνολογικών και ψηφιακών δεξιοτήτων που θα βοηθήσει του εργαζόμενου για πρόσβαση στην εργασία εργασία. Το Κοινωνικό Ταμείο Plus θα δώσει ακριβώ την ε, στήριξη μέσω του 25% για μέτρα τα οποία ακριβώ απολέπουν στην ενίσχυση των ε, κοινωνικών δράσεων για αυτού που τα χρειάζονται περισσότερα. Και το 10% θα αφορά κυρίως την ε, ανεργία των νέων και θα ενισχύσει ακριβώ την προσθέμενη αξία το ταμείο αυτό, το κοινωνικό ταμείο Plus ε, και θα, αποβλε... θα συνδέεται επίσης και με, τις, ε, με το ταμείο για τους, για τους πιο φτωχούς, για τους νέους, για την κοινωνική φτώχεια και η και το πρόγραμμα για την ε, υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, το κοινωνικό πρόγραμμα Plus θα είναι πιο συνεκτικό και πιο συμπληρωματικό σε σχέση με άλλα ταμεία τα οποία αυτή τη στιγμή παρέχουν στήριξη στους πολίτες, όπως ακριβώς το Ταμείο προσαρμογή στην, ε, στην Παγκοσμιοποίηση, Εράσμο κλπ. Το τελευταίο που θα ήθελα να θίξω είναι το Ταμείο για την επένδυση στην Ευρωπαϊκή, για την επένδυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο θα είναι πιο στοχευμένο σε πολιτικές. Η στόχη μας είναι ακριβώς η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα της οικονομικής ανάκαμψης, η, η κοινωνική ανθεκτικότητα και η υπερεκτικότητα, η περίληψη, η ένταξη των ατόμων αυτών. Και στοχεύουμε στην, στον διπλασιασμό ακριβώς της ε, στήριξης από 2 δις αυτή τη στιγμή στα 4 δισεκατομμύρια τα οποία έχουν ε, στοχευθεί για, αυτούς τους, για αυτές τις δράσεις. Και από τα 26 στο γενικό Ταμείο θα πάμε στα γύρω 50 στο πάνω πι. Και ελπίζουμε να το πετύχουμε αυτό σε συνεργασία με πολλούς ε, εταίρους, εθνικά κέντρα ας πούμε πρόθεση αυτό το δράσιο, τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένω να χρηματοδοτήσουν πιο μικρά, πιο τοπικά προγράμματα. Επίσης θα θέλαμε να είμαστε και ευέλικτοι, δηλαδή θα θέλαμε να στηρίξουμε και τις υποδομές αλλά και τις επιχειρήσεις και να μην ξεχνάμε ακριβώς αυτές τις τάσεις. Και αυτό βεβαίως σχετίζεται και με το ταμείο που σα έλεγα το, για τι επενδύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα δραματίσει σημαντικό ρόλο εδώ. Οπότε, κύριε και κύριοι βουλευτέ, τα κύρια σημεία εδώ είναι η ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα, ποιότητα εκπαίδευσης, ε, κατάρτιση διαβίου, εκπαίδευση, ακριβώς για να ενισχύσουμε και να προωθήσουμε την κοινωνική μας δομή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την προδραστική εστίαση κυρίως στα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, την κατάρτιση και των ε, ικανοτήτων. Είναι σημαντικά αυτά τα θέματα και για μας εδώ στην Επιτροπή Επασχόλησης. Να δώσω τώρα το λόγο στους συντονιστές ε, ή τους εκπροσώπους τους για δύο λεπτά. Ο κύριος Μπέκερ. Καλώς ορίσατε κύριε Αντιπρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για όλες τις ε, προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε σε επίπεδο κομισιών. Καλώς ορίζω το ότι εστιάζεται στις βασικές ε, εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς ε, είναι γεγονός ότι η αναγνώση και η γραφή θα πρέπει να συμπληρώνεται και από τις ψηφιακές δεξιότητες ως προτεραιότητα νούμερο ένα, όπως είπατε. Οι αυριανές αλλαγές συμβαίνουν σήμερα και η ψηφιοποίηση η ρομποτική και η ε, τεχνητή νοημοσύνη προσφέρουν μεγάλες ευκαιρίες στην Ευρώπη, όμως ε, φυσικά ε, θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε και ενώ βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να υπάρχουν αποκλήσεις μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχει κατακαιρματισμός της αγοράς και χαμηλή κινητικότητα ε, και βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, και αναντιστοιχίες ε, σε ό,τι αφορά τις δεξιότητες και επίσης οι στόχοι που είχαμε θέσει πριν 20 χρόνια για την απασχολησιμότητα δεν έχουν επιτευχθεί. Η δημοσίευση της Κομισιόν τον περασμένο μήνα των συγκεκριμένων συστάσεων αναχώρα τα θέτει αυτά τα προβλήματα. Να ρωτήσω πώς σκοπεύει να διασφαλίσει η Κομισιόν ότι τα κράτη-μέλη ε, θα κάνουν τι απαραίτητε μεταρρυθμίσει ε, στην αγορά εργασίας και στα εκπαιδευτικά συστήματα για να προετοιμαστούν ε, για ε, τις ταχύς αυτές αλλαγές και πώς η Κομισιόν ε, σκοπεύει να διευκολύνει την απόκτηση νέων δεξιοτήτων από το εργατικό δυναμικό προκειμένου να αντιμετωπίσει την ψηφιακή μεταλλαγή που συμβαίνει στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Αντιπρόεδρο για την παρουσίασή σας. διαφοροποιούμενος από τον κύριο Μπέκερ. Πιστεύω ότι δεν ε, επικεντρωθήκατε ορθώς ε, στις δεξιότητες και στην τεχνητή νοημοσύνη. Μας καλέσατε να σκεφτούμε τον ευρύτερο ορίζοντα, το ευρύτερο τοπίο. Πιστεύω ότι ε, στο έγγραφο που αφορά την δυσάθευση της παγκοσμιοποίηση, είπατε ότι ο κύριος παράγοντας για τη δυσάθευση της παγκοσμιοποίηση ε, είναι ε, κάποια εύρωστα καράτη προνοίας και κοινωνική Ευρώπη και φυσικά χρειαζόμαστε επενδύσεις και κοινωνικές επενδύσεις πολύ συγκεκριμένα καθώς οι επενδύσεις είναι πολύ σημαντικό τμήμα του χαρτοφυλακίου σας, νομίζω ότι θα έπρεπε να έχετε επικεντρωθεί σε αυτή την κυρία πρόκληση. τελευταία αξιολόγηση που έγινε, ανεξάρτητη αξιολόγηση που έγινε ε, αυτό το μήνα για το ΕΦΣΥ, μας λέει ότι στο καλύτερο σενάριο υπάρχει σχεδόν επίτευξη του στόχου ε, των ε, ε, αποδεδειγμένων επενδύσεων Το FC Plus ε, που αναφέρατε φαίνεται ότι θα έχει μείωση τουλάχιστον 60% σε σχέση με την σημερινή προγραμματική περίοδο των κονδύλιων ε, που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τα δύο λεπτά τελειώνουν αλλά θα ήθελα να αναφερθείτε στην κύρια πρόκληση των αυξανόμενων ανισοτήτων, της φτώχεια που επιμένει και ε, για νέες μορφές ανισοτήτων που έχουν να κάνουν και με την ψηφιοποίηση. Αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει έλλειψη εστίασης και από την πλευρά της Κομισιόν, γιατί θέτει ως μεγαλύτερη πρόκληση και θέτοντας ακριβώς ως μεγαλύτερη πρόκληση ακριβώς τις ανισότητες. Σας ευχαριστώ, η κυρία Μακεντάρ, για το CR. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω τη δήλωσή σας, κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε στις δεξιότητες και στην εκπαίδευση και στην επιχειρηματικότητα. Ήμουν σε μια συνεδρίαση της ΤΟΑ πρόσφατα όπου υπόθηκε πόσο σημαντικό είναι να διδάσκουμε τους ανθρώπους κριτική σκέψη και κάποιοι μάλιστα είπαν να διδάξουμε τους ανθρώπους να σκέφτονται είναι σημαντικό. Έτσι λοιπόν ε, πραγματικά σας ε, συγχαίρω γι' αυτό. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ε, έχουμε περίπου το χάρη 2 εκατομμύρια καινές θέσεις εργασίας και έχουμε 700.000 ελλείψεις σε δεξιότητες που αφορούν την πληροφορική και ε, περιμένουμε ουσιαστικά πολλούς ανθρώπους μέχρι το 2020 να αποκτήσουν ε, βασικά προσόντα. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα ε, με τις μαθητείες και θα πρέπει νομίζω να διδάσκουμε επιχειρηματικά προσόντα έτσι ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να δημιουργήσουν τις δικές τους ε, δουλειές. Θα μπορούσαμε να διδάσκουμε επιχειρηματικότητα και στα σχολεία. Υπάρχουν πολλοί παραδείγματα που διδάσκουμε του ανθρώπους πώς θα διευθύνουν μια επιχείρηση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε το Young Enterprise που μαθαίνει στους ανθρώπους πώς ε, μόνοι τους να μπορούν να λειτουργούν μια επιχείρηση. Τι κάνει η Κομισιόν σε σχέση με πρωτοβουλίες ε, που θα συμβάλλουν στη δημιουργία συνεργατικών σχέσεων ε, μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων προκειμένου να μπορούν οι πολίτες να έχουν ε, πρόσβαση ε, σε ε, δουλειές ε, που σχετίζονται ε, με τις τεχνολογίες των πληροφοριών και την πληροφορική. Επίσης, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την παγκόσμια απασχόληση. Είδαμε μείωση στη γεωργία, γιατί υπησέρχεται η τεχνολογία. Όμως, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε, παραδείγματος χάρη, σε μια συγκεκριμένη περιοχή περισσότερους απασχολούμενους από ό,τι πριν 200 χρόνια. Έτσι, λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε πείτε ποιε είναι οι προτάσει σα για δημιουργία θέσεων εργασία στον αγροτικό τομέα. Βλέπω ότι δεν έχω κανέναν για του φιλελεύθερου. Ε, κυρία Κάρη, για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Καταρχήν, καλώς ήρθατε, κυρία Κατάινεν, στο Κοινοβούλιο. Βλέπω ότι όλοι συμφωνούμε για το ότι χρειαζόμαστε μεγάλες επενδύσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα. Όλοι θα πρέπει να συμμετέχουμε, αλλά θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Εδώ ε, δεν μιλάμε για όσους ε, έχουν χαμηλή κατάρτιση. Ακόμη και οι δικηγόροι θα μπορούσαν ε, να αντικατασταθούν από τη τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, οι θύματα δεν είναι μόνο οι μορφωμένοι. Η ανεργία των νέων είναι επίσης πολύ μεγάλη και μεταξύ αυτών που έχουν πολλά έτη μόρφωσης. Εσείς ε, αναφερθήκατε και στην ε, μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και σε άλλες μεταρρυθμίσεις που θα επιμηκύνουν το χρόνο εργασίας. Επίσης, ε, ζητάμε μεγαλύτερη κινητικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Βλέπουμε και συρρήκνωση των μισθών όμως. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Στην Κομισιόν ε, σκέφτεστε να αλλάξετε τη στόχευση των προτάσεών σας, αντί δηλαδή να αναγκάσετε τους ανθρώπους να εργάζονται πιο σκληρά και περισσότερο, ίσως θα μπορούσε να γίνει μια κατανομή της εργασίας. Υπάρχουν ε, νέε μηχανές που κάνουν ε, καλή δουλειά, θα μπορούσαμε, πολλή δουλειά, θα μπορούσαμε όλοι να δουλεύουμε λιγότερο, να μοιράσουμε καλύτερα την εργασία για να μπορούν όλοι να συμμετέχουν και να δώσουμε περαιτέρω ευκαιρίες ε, για να υπάρχουν επενδύσεις στα νοσοκομεία, στα σχολεία. Μήπως ε, θα μπορούσατε να αλλάξετε στόχευση από την πλευρά της Κομισιόν. Μάλιστα, δεν βλέπω κανένα για τους πρασίνους. Η κυρία Γκιά για το EFTD. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα, Επίτροπε. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τα όσα αναφέρονται για την Ιταλία στις ειδικές συστάσεις χώρα κατέγραψε μικρή πρόοδο σε σχέση με το Job Act στην Ιταλία και είναι αλήθεια γιατί δημιουργήθηκε μια επισφαλής αγορά εργασίας, όπου σήμερα οι νέες μορφές εργασίας αποτελούν ένα σημαντικό ε, μέρος ανθρώπων ε, που δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι είναι καθοριστικό να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε και την οδηγία για τους διαφανείς όρους εργασίας προκειμένου να μπορέσουμε να προλάβουμε τις αλλαγές ε, ε, στον εργασιακό τομέα. Ήδη έχουμε νέες μορφές εργασίας στην κοινωνία μας και εγώ πιστεύω ότι να δημιουργήσουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο που να ρυθμίζει αυτές τις νέες ε, θέσεις εργασίας, παραδείγματος χάρη αναφέρομαι στους εργαζομένους, στις ψηφιακές πλατφόρμες και σε μία σειρά εργαζομένων με μηδενικές συμβάσεις, όλα αυτά θα πρέπει να καταργηθούν με τα οι εργαζόμενοι με τα δελτία, με τα βάουτσερ, όλοι αυτοί θα πρέπει να προστατεύονται και θα πρέπει να προβλέπουμε όρους ε, διαφανής. Ε, επίσης, ε, θα πρέπει να έχουν και ένα πολύ σημαντικό ρόλο τα συνδικάτα εμείς στο πρόγραμμά μας έχουμε προβλέψει ένα νέο διάταγμα. Ε, ο Υπουργός Εργασίας ε, θέλει να διορθώσει τις τρευλώσεις που προκαλεί το νομοσχέδιο για την απασχόληση, το Job Act. Επίσης, για τις συντάξεις μας λέει η Κομισιόν σήμερα ε, ότι αν έχουμε συντάξεις πάνω από ένα όριο δημιουργεί στρεβλώσεις αυτό. Ε, εμείς ε, το εξετάζουμε αυτό στην κυβέρνησή μας. Πρέπει να προβλέψουμε ε, και τις ανισορροπίες του συστήματος κοινωνικής προηνίας που εισήχθησαν από το σύστημα Φορνέρο. Επίσης, θέλουμε να εγγυηθούμε ελάχιστο εισόδημα που ενέκρινε πέρσι στην Ολομέλεια το Κοινοβούλιο. Αυτό πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και πρέπει να ζητηθεί από την Κομισιόν να επιτρέψει στα κράτη-μέλη που δεν έχουν ε, μορφή ε, κοινωνικής προστασίας ε, το ελάχιστο εισόδημα να μπορέσουν να εισαγάγουν αυτή τη μεταρρύθμιση και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν και κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να χρηματοδοτήσουν αυτό το ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα. Είμαι πεπισμένη ότι είναι πολύ σημαντικές και μεταρρυθμίσεις ε, στο εκπαιδευτικό σύστημα, ε, αλλά ε, δεν πρέπει να δούμε μόνο απλώς ποιες είναι οι ανάγκες της αγοράς εργασίας, αλλά να δημιουργήσουμε ένα σύστημα προστασίας και για τους μαθητευόμενους, αλλά και για τους αρμόδιους της κατάρτισης το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί πραγματικά να υποστεί μια σημαντική μεταρρύθμιση. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μαρτέν για το ΙΕΝΕΦ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Κατάινεν που ήρθε εδώ να συναντήσει τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών λαών και να μας ε, παρουσιάσει τη συνήθη λιτανία των στόχων Ευρώπη 2020. Κύριε Κατάινεν, είχα την εντύπωση ότι άκουγα έναν υποψήφιο σε προκλογική εκστρατεία. Γιατί από ό,τι φαίνεται είστε υποψήφιος για την Προεδρία της Κομισιόν το επόμενο έτος. Και Ξέρετε, όσο αποτυχάνουν οι άνθρωποι, τόσο του ε, προσλαμβάνει η Κομισιόν. Να σα υπενθυμίσω τον κύριο Μπαρόζο, ο οποίο ε, βήθησε ε, την Πορτογαλία και μετά δέχτηκε τελικά τη βρύθμιση τη Τράπεζα και κατέληξε στην Goldman Sachs και ο κύριος Γιούνκερ ήταν πρόεδρος του Λουξεμβούργου, φορολογικού παραδείσου και στη συνέχεια έγινε πρόεδρος μιας κομισιόν που μιλάει για φορολογική ελληνική ο ε, επικεφαλής ε, της βελγικής αστυνομίας ε, μας έδειξε ότι ήταν ανίκανος στην αντιμετωπίση της τρομοκρατικής επιθέσεις και έγινε επικεφαλής της Europol. Και στη Φιλανδία η Νόκια εξαγοράστηκε για να την κλείσουν. Έτσι είχαμε 27.000 απολυμμένους χωρίς να υπολογίσουμε ε, στην ε, Εξαλκατέλ τι έγινε στη Γαλλία και πώς ε, τις θέσεις εργασίας χάθηκαν. Έτσι λοιπόν, σας, σας αναθέτουν στις Βρυξέλλες το χαρτοφυλάκιο που αφορά την απασχόληση, την αντιγωνιστικότητα και το κόμμα σας κλείνει ε, τα κινητά νοσοκομεία στη Φιλανδία. Ε, να λοιπόν το μέλλον της Φιλανδίας. Έτσι λοιπόν ε, κύριε υποψηφία Κατάιναν έχετε κάθε πιθανότητα να διοριστείτε ε, του χρόνου. Βέβαια υπάρχουν και εκλογές του Μαΐου του 2019 και οι λαοί θα εκφραστούν εκ νέου και θα κρίνουν τις πολιτικές αυτές που απλώς καταστρέφουν τους κυρίαρχους λαούς που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, να πω εδώ ότι είναι πολιτική συζήτηση για το προσανατολισμό που παρουσιάστηκε και όχι να αναφέρουμε τα διάφορα οράματα στη συγγνώμη. Κύριε Μαρτέν, εγώ έχω το λόγο, σας τον έδωσα το λόγο. Κύριε Αντιπρόεδρε, για να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Για τα θέματα που έθεσε ο κύριος Μπέκερ καταρχήν. Πώ να διασφαλίσουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για να αποκτήσουν περισσότερα προσόντα ε, οι εργαζόμενοι και να αυξηθεί η προσαρμοστικότητα πρέπει να επιδιωχθούν από τα κράτη-μέλη. Όπως είπα, φέτος, ως μέρος ε, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, δώσαμε περισσότερη προσοχή στην εκπαίδευση. Αυτή ήταν μια προσωπική μου αποστολή. Πιστεύω ότι όχι μόνο οι δεξιότητες αλλά και η βασική εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό στοιχείο για μια ευημερούσα κοινωνία στο μέλλον. Επίσης, είναι σημαντικό από τη σκοπιά της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αν δείτε την μελέτη του ΩΣΑ για την πίζα, βλέπετε τεράστιες διαφορές στη βασική εκπαίδευση μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό είναι απαράδεκτο σε πολλά κράτη-μέλη, αν η εκπαίδευση δεν ήταν πολιτική, η εκπαίδευση δεν ήταν πολιτική προτεραιότητα για πολλά ε, χρόνια. Ε, οι επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο δεν ε, ήταν ιδιαίτερα αποδοτικέ σε προκλογική περίοδο. Και αυτό στο παρελθόν ίσχυε γιατί ήταν κάπως ε, πιο απλή ζωή, ενώ τώρα γίνεται πιο πολύπλοκη. Πολλοί από εμάς είναι υπέρ μιας πιο ανοιχτής κοινωνίας χωρίς ε, σύνορα και επίσης οι νέες τεχνολογίες θα κάνουν τη ζωή μας ταυτόχρονα πιο εύκολη αλλά και πιο σταθή. Για αυτό προσωπικά λέω ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση σε θέματα που φορούν το ανθρώπινο κεφάλαιο από ό,τι στο παρελθόν, λόγω των ε, αλλαγών που γίνονται στην κοινωνία μας. Γι' αυτό οι ειδικέ συστάσεις αναχώρας είναι το ένα. Τώρα το δεύτερο. Έχουμε μία υπηρεσία που υποστηρίζει τις ευθεωτικές μεταρρυθμίσεις, λειτουργεί αρκετά καλά, και μάλιστα θα προσφέρει ακόμη περισσότερε υπηρεσίε στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Θέλουμε να ενισχύσουμε την ε, υπηρεσία ε, στήριξης ε, των μεταρρυθμίσεων σαν την παρουσιάσουμε σε μια τακτική υπηρεσία για τα κράτη-μέλη και θέλουμε να αλλάξουμε και τη φήμη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που είχαν αρνητική θεώρηση για διάφορους λόγους. Θέλουμε να αλλάξουμε λοιπόν αυτή την ε, φήμη και επειδή έχουμε μετασχηματισμούς ε, στην στον κόσμο μας πρέπει να αλλάξουμε και τις δικές μας κοινωνίες. Γι' αυτό η στήριξη της Κομισιόν στα κράτη-μέλη είναι πολύ πιο σημαντική σήμερα από ό,τι στο παρελθόν. Επίσης έχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για το θέμα αυτό και φαίνεται να λειτουργεί αρκετά καλά. Αυτός είναι ένας τρόπος λοιπόν να βλέπει κανείς τα πράγματα. Για τα προσόντα και την ε, εκπαίδευση. Έχουμε μία υπηρεσία δωρεάν για τα κρατη και εντελώ εκούσια. Παραδείγματο χάρη, κάποια κράτη-μέλη θέλουν να μεταρρυθμίσουν το εκπαιδευτικό του σύστημα. Η Κομισιόν μαζί με τον ΟΣΑ μπορεί να δημιουργήσει μία task force μαζί με τον ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ε, για να ε, αξιολογήσει το σημερινό σύστημα και να δώσει κάποιες συμβουλές ε, για τις μεταρρυθμίσεις. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί τόσο πολύ. Υπάρχει ήδη όμως εδώ και δύο χρόνια. Αν σας αρέσει η ιδέα λοιπόν, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Η μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών συστημάτων φέρνει αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα στην Πορτογαλία, παραδείγματο χάρη, και στην Ιστονία. Οι χώρε αυτέ μεταρρύθμισαν το εκπαιδευτικό του σύστημα και βλέπουμε ήδη ωφέλη. πέντε έτη μετά τι μεταρρυθμίσει. Αξίζει λοιπόν. Τώρα, πόσο κομισιόν διευκολύνει την αποκτήση περισσότερων προσόντων. Ε, όλο το θεματολόγιο για τα νέα προσόντα μας δίνει συγκεκριμένο παραδείγματος χάρη, παραδείγματος χάρη ε, ο συνασπισμός ε, για την απασχόληση και τα ψηφιακά προσόντα ε, και το δημο, ο δημόσιο αλλά και ο ιδιωτικό τομέα μπορεί να μα δώσει βαλτιστέ πρακτικέ. Αναφέρθηκε το τι έγινε εδώ στο Βέλγιο, παραδείγματο χάρη. και υπάρχει ε, μεγάλο ποσοστό εκπαίδευσης ε, ε, στα σχολεία στο Βέλγιο. Παραδείγματο χάρη και στην Ιρλανδία έχουν προσλάβει κάποιους ανέργους με καλά αποτελέσματα. Και τέλος, για τις επενδύσεις. έχουμε τα Ευρωπαϊκά Διευθυντικά Ταμεία, είναι το νέο Ταμείο Επενδύσεων. Έχω συζητήσει με κάποιους ε, υπουργούς παιδείας και τους πρότεινα να σκεφτούν να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα Erasmus Plus, κυρίως για τους εκπαιδευτικούς και για όσους σπουδάζουν ε, παιδαγωγική. το χάρη, μια χώρα αποφασίσει ότι το 10% ή το 20% όσων ε, σπουδάζουν παιδαγωγικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το Erasmus ή ένα συγκεκριμένο ποσοστό των εκπαιδευτικών θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το Erasmus Plus. Φανταστείτε ε, τι θα σήμαινε αυτό για το κοινωνικό κεφάλαιο. Όχι δηλαδή ότι πρέπει να μαθαίνεις πάντα από το εκπαιδευτικό σύστημα των άλλων χωρών, αλλά ε, όταν, εφόσον γίνονται πιο διεθνοποιημένε οι κοινωνίε μας, είναι πολύ σημαντικό και οι εκπαιδευτικοί μας να μπορούν να παρακολουθούν αυτές τις εξελίξεις. Το Erasmus Plus, ιδιαίτερα στην επόμενη ε, προγραμματική περίοδο, ε, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και από τους φοιτητέ παιδαγωγική αλλά και από τους εκπαιδευτικούς. Τώρα, αναφερθήκατε στη φτώχεια και στις ανισότητες. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά από τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη, αλλά μπορεί να κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλά εδώ, κυρίως στοχεύοντας ε, τις επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές. Θέλουμε να αντικαταστήσουμε το ΕΦΣΥ με το InvestEU Fund, που θα είναι πιο προσανατολισμένο προς επενδύσεις. Θα έχουμε τέσσερις θηρίδες επένδυσης, ε, την έρευνα και την ανάπτυξη, το κοινωνικό, τις βιώσιμες υποδομές και τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Το You Fund θα ε, αφορά περισσότερο τις πολιτικές. Φυσικά θα πρέπει κάποιος να ενδιαφέρεται να επενδύσει στο κοινωνικό κομμάτι. Όμως ε, θέλουμε να επικεντρωθούμε στο να χρησιμοποιήσουμε περισσότερα αυτά τα εργαλεία σε σχέση με το ΕΦΣΥ. Εκτός και αν το Κοινοβούλιο αλλάξει την πρότασή μας, στοχεύουμε να διπλασιάσουμε ε, τα ποσά που αφορούν ε, τα προσόντα και τις κοινωνικές υποδομές από 2 σε 4 δισεκατομμύρια. Δεν είναι τέλος πάντων τόσο πολλά αλλά θα φτάσουμε από τα 26 δισεκατομμύρια σε 50 εκατομμύρια με όρους πραγματικών επενδύσεων. Λοιπόν, για την ε, μαθητεία. Νομίζω ότι η μαθητεία είναι ένας πολύ καλός τρόπος και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ευρύτερα στα κράτη-μέλη μας, γιατί είναι ένας από τους πιο δυναμικούς τρόπους να οργανώσουμε την ε, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Επίσης, ε, τα προσόντα της επιχειρηματικότητας είναι σημαντικά μέχρι τώρα ε, το, η κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα φαινόταν ε, ως ε, το δεύτερο καλύτερο. να δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο, μπορείς να γίνει επιχειρηματίας το χάρη. Αλλά αν δείτε το στόχο των νέων, ουσιαστικά θέλουν μια δουλειά που να έχει νόημα. Και μερικές φορές το να γίνει κανείς επιχειρηματίας είναι ο τρόπος να κάνει κάτι που να έχει νόημα. Η επιχειρηματικότητα δεν είναι σημαντική αυτή καθ' αυτή, αλλά είναι ένας τρόπος να οργανώσω τη βούλησή μου να κάνω κάτι που θέλω. Και γι' αυτό ε, επιχειρηματικότητα συμπεριλαμβάνεται στα προγράμματα σπουδών, ε, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στα προγράμματα σπουδών με καλύτερο τρόπο για το μέλλον τα ψηφιακά προσόντα και ο συνασπισμός για την απασχόληση είναι ένας ε, τρόπος ε, να ε, φέρουμε σε συνεργασία τις δημόσιες αρχές με τους κοινωνικούς εταίρους έτσι ώστε να αποκτήσουν ευκαιρίες οι άνθρωποι για απόκτηση περαιτέρω προσόντων. Όταν αλλάζουν τα προσόντα που χρειαζόμαστε, Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι όλα μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς φορείς. Γι' αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί και ο ιδιωτικό τομέα. Και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Λοιπόν, τώρα, για την Ήπεθρο. Βλέπω ότι σε σχέση με το παρελθόν όλες αυτές οι διαφορετικές αλλαγές που κάναμε θα βελτιώσουν την προσβασιμότητα στην Ήπεθρο. Παραδείγματο χάρη, τα χιλιόμετρα μεταξύ των αστικών περιοχών και των χωριών δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία όπως το παρελθόν. Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η προσβασιμότητα βελτιώνεται, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλες οι αγροτικές περιοχές ε, αποτελούν προορισμό επενδύσεων Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, πρέπει όλοι να έχουν τι ίδιε ευκαιρίε σε σχέση με την ψηφιακή σύνδεση. Για το θέμα τη κατανομής τη εργασία. Επειδή αλλάζει η φύση τη δουλειά. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει νέα κατανομή εργασίας. Απλά θα πρέπει να δυσφαλίσουμε ότι οι συνθήκες εργασίας είναι δίκαιες Δεν πιστεύω ότι έχει νόημα οι δημόσιες αρχές να αρχίσουν ε, να μοιράζουν τις ε, υφιστάμενες ε, θέσεις απασχόλησης για να δώσουν δουλειά σε κάποιους που δεν έχουν. Αλλά θα πρέπει να δούμε το εξή. Τα συστήματα κοινωνικής μας ασφάλισης είτε επιτρέπουν να συνδυαστούν οι προσωρινές της απασχόλησης ε, η η ημερική απασχόληση πρέπει να μπορεί να επιτρέπει να συνδυάζεται καλύτερα σε σχέση με σήμερα. Έχαν συνδυαστεί αυτά τα συστήματα όταν ε, κάποτε είχαν ε, όλη δουλειά και πήγαιναν για δουλειά στις 8 το πρωί και γύρναγαν στις 4 5 το απόγευμα. Έτσι λοιπόν τα συστήματα Κοινωνική πρόνοια ήταν κάπως ε, εύκολο να δημιουργηθούν τότε που ήταν μονολυθικό ο κόσμος. Ε, τώρα όμω έχουν αλλάξει τα πράγματα και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τα συστήματα κοινωνική ε, προστασία με έναν μεταλλασσόμενο κόσμο. Μερικές φορές τις λύσεις τις διαπραγματεύονται και οι κοινωνικοί εταίροι. Και ένα τελευταίο θέμα, το οποίο το σημείωσα, που δεν ήταν και τόσο εντός θέματος. Υπήρξε τέλο πάντων ένα θέμα, σημείωσα τι ήθελε να μου πει ο μιλητή. Σας ευχαριστώ, δύο άτομα έχουν ζητήσει ακόμη το λόγο για τις προκλήσεις που αναφέρατε. Είναι αλήθεια ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν μεγάλες προκλήσεις. Τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλά μέσα για να διορθώσουμε όσα δεν πήγαν καλά, αλλά αν δούμε ε, τις διάφορες σπουδέ που υπάρχουν σε διάφορα κρατημέλη και βλέπω και ε, τις ε, διαφορές μεταξύ των νέων που βγαίνουν από το σχολείο χωρίς απολυτήριο είτε επειδή το έχουν εγκαταλείψει είτε γιατί έχουν αποκλειστεί νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό για να αποφύγουμε ακριβώς ε, να ακολουθήσουν ε, οι άνθρωποι αυτοί μια καταστροφική πορεία. Σοφία Ριμπέρο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, κύριε Επίτροπε. Η αρχική σας ομιλία για τις επενδύσεις ε, στην εκπαίδευση και στην αναγκαιότητα να ενταχθεί αυτό στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ξαμήνου και να έχουμε συνεχή κατάρτιση για τους εκπαιδευτικούς και επίση, ε, αναφέρεται ότι έχουμε μεγάλε προκλήσεις, ε, τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική. Όλα αυτά απαιτούν να έχουμε τους καλύτερους εκπαιδευτικούς στα σχολεία. Όμως για να έχουμε τους καλύτερους καθηγητές στα σχολεία θα πρέπει να έχουμε πολιτικές που να δίνουν κίνητρο για να έχουμε τους καλύτερους εκπαιδευτικούς. Και αυτό δεν μπορεί να συμβεί με μειώσεις των μισθών ή όταν ε, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος εργασίας ή η οταν δεν λαμβανεται υποψη ο χρόνο εργασιας η η δουλεια που κάνουν οι καθηγητές. Χρειάζεται λοιπόν να φέρουμε τους καλύτερους εκπαιδευτικού, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε εγγύησει ότι θα κάνουμε την καλύτερη δυνατή δουλειά και θα μπορούμε να διαδώσουμε τη γνώση με τον καλύτερο τρόπο. Αυτές οι πολιτικές δεν είναι συμβατές με την μείωση των ε, κονδυλίων ε, στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο ε, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είχαμε μια συζήτηση με τις τρέχουσες τιμές και τις συνεχείς τιμές, όμως ουσιαστικά εδώ συγκρίνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ταμείο με το ESF ε, Plus και αυτό οδηγεί σε ε, απομείωση της αξίας τους. Όμως είναι απαραίτητο εμείς να, και τις, να έχουμε και τις κατάλληλες πολιτικές ε, για, τις, για την Ήπεθρο. αυτό φυσικά δεν συνάδει με τις περικοπές στο Ταμείο Συνοχής της τάξης του 45%. Τώρα, ε, ακούσαμε ότι έχουμε το Brexit ε, και ότι πρέπει να εστιάσουμε στην άμυνα ε, και επομένως πρέπει να υποστούμε αυτές τις απώλειες. Όμως, εντό της πολιτικής συνοχής έχουμε χώρες που χάνουν κονδύλια για άλλες που κερδίζουν. Αυτό και στην Πορτογαλία. Είπατε, βελτιώσατε τους δείκτες σας. Όμως, το 2013 προσπαθούσαμε να βγούμε από μια χεροκοπία και Όλη η προσπάθεια που έγινε ήταν μια βαθιά προσπάθεια, σκληρή προσπάθεια για τους Πορτογάλους. Και τώρα, αν ε, δεν δουν ότι τους βοηθά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ε, αισθανθούν εντελώς εγκαταλελειμμένοι. Έτσι λοιπόν, αυτό πρέπει να δούμε. Η οικονομική και η κοινωνική και επενδυτική πολιτική θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα κονδύλια, κυρίω στι περιοχέ με τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τι ανισότητε, αλλά θα τι αξίσουμε εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Κύριε Πυρίνσκι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κατάινεν που απάντησε σε ένα ερώτημα που έθεσα για τις κοινωνικές επενδύσεις συγκεκριμένα. Πολύ σωστά λέτε ότι κοινωνικές πολιτικές είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά ε, στόχο έχει να δίνει κίνητρα και να υποστηρίζει με οικονομικό τρόπο τους μίζωνες κοινωνικούς στόχους. Όμως, μιλώντας για κοινωνική ευθύνη. Μιλήσατε κι εσείς για τα εκπαιδευτικά συστήματα, συστήματα για τα οποία πλήσαν περισσότερο από τις πολιτικές λιτότητας και τα σχετικά μέτρα. Και είπατε ότι ήταν έτσι πιο προβεβλημένο το να χτίζει κανείς δρόμους ή κάτι τέτοιο. Ε, έχοντας υπόψη μας και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και την αυξανόμενη προσοχή που δίνεται στα κοινωνικά ζητήματα λόγω και του κοινωνικού πυλώνα. Έχω να σας ρωτήσω το εξή. Οι ανισότητε και η κινητικότητα στον πίνακα, το scoreboard, δεν θα έπρεπε να ε, περιλαμβάνει και τον ε, συντελεστή Τζίνι που δείχνει τις ε, ανισότητες ώστε να γνωρίζει κάθε χώρα. Να γνωρίζουμε τι γίνεται σε κάθε χώρα. Στη Βουλγαρία, για παράδειγμα, αυτός ο δείκτης αυξάνεται. Είναι ένας από τους υψηλότερους. Έχοντας υπόψη ότι πρέπει να πιάσει και τους άλλους ε, η Βουλγαρία στους στόχους. Επίσης για 2,4 δις ε, από το 2016 να πάνε στα 50 δις ε, είπατε. Υπάρχει έκθεση ψηλού επίπεδου αρχές του έτους που υπολογίζει σε 100 με 150 δις ε, την τρύπα στις επενδύσεις ετησίως. 1,53 μέχρι το 2030 νομίζω είναι τα ποσά τα οποία υπολογίζονται. Και αυτό το οποίο τώρα έχει σχεδιαστεί είναι να καλυφθεί το μισό αυτού του κενού της τρύπα. Αν όμως ο στόχος είναι τα μισά ε, για να αποφύγουμε την τρύπα, πέφτουμε μέσα στην τρύπα. Και επομένως αυτή η λύση δεν είναι λύση. Επίσης αναφέρατε συνολικά την ε, εμπειρία μας από το ΕΦΣΙ, το Ταμείο Στρατικών Επενδύσεων. Στην προηγούμενη παρέμβασή μου μίλησα για τις τεράστιες γεωγραφικές ανισορροπίες ό,τι αφορά τις επενδύσεις. Γνωρίζω ποιε είναι οι εξηγήσεις που δίνονται ε, για το ΑΕΠ, για το μέγεθος των χωρών, αλλά όποιες και αν είναι οι εξηγήσεις, το αποτέλεσμα παραμένει. Παραμένουν και ανισότητες. Οι αγροτικές περιοχές πλήττονται κυρίως, το είπε και η κυρία Μάκιντάιρ. Επομένω, πιστεύω ότι εάν πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πετύχει ε, αλλαγή και στροφή, θα πρέπει να υπάρξουν προσπάθειες ε, εκ νέου στον τομέα της ε, κοινωνικής συνοχής και της συνοχής εν γέννη. Τέλος. Μιλήσατε για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις παραδοσιακά όταν αναφέρονται συσχετίζονται με την άρση των φραγμών ε, στον ανταγωνισμό, φεξέλικτες αγορές, ε, εργασίες κτλ. κτλ. Η Επιτροπή ε, ε, κύριε Αντιπρόεδρε, επασχόληση ανέκρινε μια έκθεση η οποία είχε να κάνει ακριβώ με το πρόγραμμα υποστήριξη των διαθροτικών μεταρρυθμίσεων και στην ε, εκθέση αυτή πολύ ξεκάθαρα τονίσαμε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται ε, μεταρρυθμίσεις στον τομέα της στέγασης, της υγείας και της εκπαίδευση επομένω. καλά κάνετε και νεύετε ε, θετικά σε αυτά που λέω, αλλά θέλω να υπάρξουν ε, και πράξεις ε, σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Όπως είπατε, είναι και σημαντικός παράγοντας για να γίνει αυτή η στροφή στα κράτη-μέλη. Τέλος, στη Σόφια το Φεβρουάριο έγινε μια διάσκεψη με μεγάλη συμμετοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα φασμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επένδυση στους ανθρώπους, ο δρόμος που τα μπρος. Αυτός ήταν ε, ο τίτλος, ήταν το σλόγγαν. Ας προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εσείς ε, κύριε Κατάινεν ε, για τελευταία φορά για να απαντήσετε. Ναι, ευχαριστώ. Για την κυρία Ριμπέιρο ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρξουν κίνητρα για τους δασκάλους, εκπαιδευτικούς, είπατε για τους μισθούς των εκπαιδευτικών. Φυσικά είναι ένα σημαντικό κομμάτι για τη δημιουργία κινήτρων. Γιατί κάποιος να θέλει να γίνει εκπαιδευτικός. Θέλουμε τους πιο ταλαντούχους και αφοσιωμένους ή κάτι άλλο. Θα ήθελα να τα συσχετήσω αυτά σε αυτό που είπε ο κύριος Πυρίνσκι για τις διαθετικές μεταρρυθμίσεις στον κοινωνικό τομέα και την εκπαίδευση μεταξύ άλλων. Πρέπει να σας πω ότι εξεπλάγει κάπως βλέποντας κάποιο στατιστικό στοιχείο που λέει ότι η Φιλανδία χρησιμοποιεί λιγότερο από το μισό, ε, από το μέσο όρο του ΩΣΑ ε, για την εκπαίδευση, αλλά με πολύ καλά αποτελέσματα. Επομένως, ε, τα χρήματα δεν είναι το μόνο που εξηγεί. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν θα πρέπει οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί να παίρνουν ε, υψηλούς μισθούς ή να μην αμείβονται σωστά. Σίγουρα δεν είναι, αλλά... Το θέμα είναι πώς θα γίνει να είναι και σεβαστό και καλά αμοιβόμενο το επάγγελμα. Ε, όταν ήμουν πρωθυπουργό στη χώρα μου, η κόρη μου πήγαινε σχολείο και ήταν έξι ετών τότε. Μια από τις πρώτες μέρες λοιπόν στο σχολείο εγώ με την κυβέρνηση ε, κάναμε μια συνέντευξη τύπου τον Αύγουστο ε, και παρουσιάσαμε τον προϋπολογισμό. Με έπαιρνε τηλέφωνο ε, ε, κόρη μου ε, και βγήκα έξω για να συζητήσω μαζί της, ε, γιατί νόμιζα ότι κάτι συμβαίνει. Ήθελα να πω για τον δάσκαλό της. Ε, Γενικώ είναι πάρα πολύ σημαντική εκπαιδευτική λοιπόν και όχι μόνο για τα χρήματα. Λέμε πάντα ότι πρέπει να αξιοποιούνται καλύτερα οι πόροι και οι επαγγελματίε, καθηγητέ, εκπαιδευτικοί να είναι ε, ε, καλύτερα αμοιβόμενοι, να έχουν μεγαλύτερο σώμα και, και τα κτλ. Σίγουρα προ αυτές τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις κοινωνικέ θα πρέπει να προχωρήσουμε και η Πορτογαλία είναι ένα καλό παράδειγμα. Τουλάχιστον με βάση τον όσα. Έχει καλή απόδοση η Πορτογαλία. Και ναι, πράγματι υπάρχουν αυτές οι εκτιμήσει. Τα κοινωνικά κονδύλια θα είναι πάνω από 100 δις, λέει ο κύριος Κατάιν. Και θα έχουμε και άλλες επενδύσεις. Έχει βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση, καλά νέα και αυτά. Δεν είναι τα κονδύλια που προβλέπονται στην Επιτροπή βέβαια ε, για τη συνοχή, αλλά τέλος πάντων. Τέλος. Επενδυτικό κενό. 100 δις, 50 δις κτλ. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν τη δική τους δουλειά. Δεν μπορούν να βγαίνουν όλα τα χρήματα από τον ενωσιακό Προϋπολογισμό. Για το ΕΦΣΥ, τέλος, γεωγραφικές ανισορροπίες. Ο πιο ρεαλιστικός τρόπος να εξετάσει κανεί αυτό το θέμα είναι να δει τι επενδύσει σαν ΑΕΠ. Ε, how much a country για να δούμε πώς κάθε χώρα αξιοποίησε τα κονδύλια του ΕΦΣΥ δεδομένου του μεγέθους οικονομίας της. Ο μεγαλύτερος χρήστης του ΕΦΣΥ ανά είναι η Ελλάδα, με δεύτερη τη Βουλγαρία. Όχι, λάθος, Εστονία, Βουλγαρία, Πορτογαλία, Ισπανία. Και έξι, στην έκτη θέση η Φιλανδία. Και ξέρετε κάτι, είναι το καλύτερο κρυμμένο μυστικό, δεν το ξέρει κανένας. Ευχαριστώ που το ρωτήσατε κιόλας παρότι κινείται με βάση τη ζήτηση το ΕΦΣΥ, έχει ε, καταφέρει να κάνει αυτό που όλοι θέλαμε, να δώσει χρηματοδότηση, να αντιμετωπίσει τι αστοχίες αγορά. Και χρηματοδοτεί όχι μόνο ΜΜΕ, ε, βέβαια, αλλά και άλλε και άλλα project. Όλες τις λεπτομέρειε μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα και πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Αυτά είχα να πω πολύ καλή συζήτηση. En tous les cas, c'est nous qui vous remercions de, de vous prêter à cet exercice, mais je le redis, je l'ai dit en σας είπα και το ξαναλέω και τώρα, είναι ένα εγχείρημα αυτό στο διαδρομένο διάλογος πάρα πολύ σημαντικός ε, για εμάς. Σας ευχαριστούμε, θα τα ξαναπούμε και ευχαριστούμε για αυτή τη μόνιμη ανταλλαγή μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν. Και τώρα φτάνουμε στο τελευταίο σημείο που έχουμε στην ημερήσια διάταξη για σήμερα το πρωί. Είναι ένα κάπως ιδιαίτερο σημείο, σημείο ε, στην ημερήσια διάταξη, γιατί δεν αφορά ε, έκθεση ή γνωμοδότηση για ένα κείμενο από το οποίο έχουμε τροπολογίες. Όμως, στην τελευταία ε, συνεδρίαση της επιτροπή απασχόληση είχαμε τη δυνατότητα ε, και έλαβαν το λόγο διάφοροι βουλευτέ να συζητήσουμε την διαμάχη, τη διένεξη που υπάρχει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, υπάρχει μια εργασιακή κοινωνική διένεξη ε, με του διερμηνεί. την κατηγορία αυτή του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έγινε την τελευταία εβδομάδα στο Στρασβούργο μια συνάντηση για το θέμα και αποφασίσαμε να αφιερώσουμε χρόνο, περιορισμένο μεν, αλλά να έχουμε μια δυνατότητα ανταλλαγή απόψεων με του στην πρώτη γραμμή ενδιαφερομένου του, εκπροσώπους των διερμηνέων. Θέλαμε να αφιερώσουμε ένα μισάωρο λοιπόν στην ε, ε, περίπτωση, υπόθεση αυτή, σε δύο μέρη θα χωριστεί. Καταρχάς θα ακούσουμε τους εκπροσώπους των διερμηνέων στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο τέταρτο, θα μπορέσουμε να ακούσουμε παρεμβάσεις από τους ε, συντονιστές και άλλους συναδέλφου που ενδεχομένως είναι παρόντες. Θέλω να ευχαριστήσω τους διερμηνείς πρώτα απ' όλα για το έργο τους, για τη δουλειά τους, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ε, ακόμη και στην στιγμή αυτή που, βρίσκεται, που υπάρχει αυτή η διένεξη Θέλουμε να μας παρουσιάσετε την κατάσταση και τα αιτήματά σας. Αυτό ε, που θέλω να πω εγώ, νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι βουλευτέ ε, δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ό,τι το περιεχόμενο τη δικαστικής, ε, της εργασιακή αυτής διένεξη μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι ένα είδο εταιρεία, επιχείρηση σε κάποιο βαθμό, αλλά επειδή άκουσα τις παρεμβάσεις της τελευταίας της Επιτροπής μας, είναι νομίζω σημαντικό στο Κοινοβούλιο που προάγει την αρχή της διαβούλευσης και του κοινωνικού διαλόγου να ε, είμαστε βέβαιοι ότι μπορεί αυτός ο διάλογος να γίνεται με πλήρη και σωστό τρόπο. Θα σας δώσω λοιπόν το λόγο σε 15 λεπτά. Έχετε το λόγο κύριε Ρομπέρτο Ακουίνο ε, και οι κυρίες Άστρικτ Κνόκε και Άννα Μπίβας Μπάιλο Ελπίζω να προφέρω σωστά τα ονόματά σα. Δεν είμαι δυστυχώ εγώ γλωσσολόγος, γλωσσομαθής. σα δίνω λοιπόν το λόγο για ένα τέταρτο. Εσεί ξέρετε πώ θα τον μοιράσετε μεταξύ σας. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία και ευχαριστώ όλα τα μέλη τη Επιτροπή που μα ε, υποδεχθήκατε τόσο σύντομα. Θα είμαι σύντομο κι εγώ και στο συγγνώμη εκ των προτέρων από τους αδέλφους αν η παρουσίαση θα είναι στα αγγλικά, αλλά δυστυχώς έτσι πρέπει να είναι. Καταρχάς το κυριότερο που θα ήθελα να πω από την αρχή είναι ότι είμαστε μια ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού. Αυτό το αναγνωρίζει και το καταστατικό και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε ιδιαίτερε συνθήκε εργασία Για ποιο λόγο. Γιατί όπως αναγνωρίστηκε από πολλέ ιατρικές μελέτες έχουμε υψηλό επίπεδο άγχους, εργασιακούς, ε, χρειάζεται να αφήσει υψηλό επίπεδο συγκέντρωση γιατί κάνουμε διάφορε εργασίε ταυτόχρονα. ακούμε, επεξεργαζόμαστε και ταυτόχρονα μεταφράζουμε σε πολλέ γλώσσε. Και δεν έχουμε ε, έλεγχο για το αριθμό τη εργασία μα, ο οποίο καθορίζεται από του ομιλητέ. Οπότε θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε οποιαδήποτε ταχύτητα θα αντιμετωπίσουμε. Και αντίθετα με το υπόλοιπο προσωπικό, δεν έχουμε γραφεία, δηλαδή είμαστε ένα περιοδεύον επάγγελμα το οποίο εργάζεται σε κλειστό χώρο. Υπάρχουν επίση συγκεκριμένε προκλήσει που σχετίζονται με το Κοινοβούλιο και την διερμηνία. Καταρχάς ξέρετε ότι έχουμε πολύ σύντομο χρονομιλία το οποίο οδηγεί σε πολύ υψηλέ ταχύτητε όταν διαβάζετε ομιλίε και θα δείτε ότι ο μέσο όρο σε ένα συνήθε περιβάλλον, περιβάλλον, εδώ αυτό ο αριθμό που βλέπετε ότι είναι αρκετά φύσικος. 225 δηλαδή λέξεις ένα λεπτό. Προσπαθούμε όλα αυτά να τα συνδυάσουμε με την αντιμετώπιση και άλλων προκλήσεων, τεχνικές συνεδριάσεις εδώ που θα πρέπει να προετοιμάσουμε και οι νέες συνθήκες εργασίες που επιβλήθηκαν τον περασμένο Αύγουστο δεν αφήνουν αρκετό χρόνο προετοιμασίας και αυτό θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα της υπηρεσίας μας. Έχουμε και υψηλό άγχος λόγω ε, τηλεδιασκέψεων. Πολλές ε, συνεδριάσεις ε, μεταδίδονται. Οπότε δεν περιζόμαστε μόνο ως ακροατές στους παρόντες και δεν έχουμε κανένα έλεγχο και στο πρόγραμμα εργασία μας, το οποίο καθορίζεται από την μονάδα προγραμματισμού και θα πρέπει να προσαρμοστούμε γιατί συχνά έχουμε αλλαγές τελευταίας στιγμής. Περμαστε και ευέλικτοι. Γιατί διαμορφωνόμαστε λοιπόν. Επειδή είμαστε λοιπόν μια πολύ ιδιαίτερη κατηγορία εργαζομένων, ήμασταν πάρα πολύ ευέλικτοι εδώ και δεκαετίε και τώρα διαμαρτυρόμαστε διάφορους λόγους. Καταρχάς υπάρχουν νομικά ζητήματα. Οι νέες συνθήκε εργασία επιβλήθηκαν μόνο μερό κατά παράβαση διαφόρων κανόνων, καταρχάς την ρήτρα αναθεώρηση των προηγούμενων συνθήκων εργασία που προέβλεπε μια συμφωνία με τους διερμηνεί, κανονισμούς που αφορούν το προσωπικό, επειδή υπάρχει μια διάταξη η οποία καθορίζει ακριβώ την ανάγκη για διαβούλευση όσον αφορά την Επιτροπή Προσωπικού πριν γίνουν αυτέ οι αλλαγέ. Αυτή η διαβούλευση δεν έλαβε χώρα. Και επίση υπάρχει ένα συγκεκριμένο ζήτημα στο νέο κείμενο το οποίο παραβιάζει την οδηγία για το ωράριο εργασίας, ιδιαίτερα για τον χρόνο ανάπαυσης. Υπάρχει επίσης παράβαση συμφωνίας, ε, της συμφωνίας μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και δερμηνών freelance αυτοπασχολουμένων. Από και εκεί δεν τηρείται ακριβώς ο χρόνος εργασίας. Φτάσαμε στο οποίο που είμαστε επειδή δεν υπήρχε επαρκή διάλογο. Όπω ξέρετε, είχαμε την ειδοποίηση για απεργία στι 29 Μαου και από τότε δεν είχαμε καμία συνάντηση μεταξύ δηλαδή τη διοίκηση του Ευρωκοινοβουλίου και των συνδικαστικών οργάνων ώστε να βρούμε μια συνετική λύση σε αυτή τη διένεξη. Επίσης, η διαβούλευση η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή υπό τη Γενική Γραμματέα της Διοίκησης και της Επιτροπής Προσωπικού και των συνδικαστικών οργάνων έπρεπε μάλλον να έχει ολοκληρωθεί στο, το 2017 δεν απέδεσε, απέδεσε κανένα καρπό μέχρι τώρα και ήταν μια μακροχρόνια διαδικασία χωρίς αυτά αποτελέσματα. Ας πάμε όμω λίγο πίσω στο παρελθόν, να δούμε ποια ήταν τα προβλήματα στο κοινωνικό διάλογο πριν πάμε στην ε, αναγγελία της ε, απεργίας. Η διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σταμάτησε τι διαπραγματεύσει δύο φορές μονομερός, και απέτρεψε την ανέβρεση συγκλήσεων. Άλλαξαν οι στόχοι της διοίκησης ε, συνεχώς. Μιλάμε για αδιαφάνεια σε σχέση με τι αρχικέ ε, συζητήσει. Υπήρχε έλλειψη διαφάνεια. Κανεί από του Ερμηνεί, ούτε η Επιτροπή Προσωπικού, δεν είχαν πλήρη πρόσβαση στι στατιστικέ και στα δεδομένα τη Γενική Διεύθυνση για να δουν κατά πόσο πραγματικά τα αιτήματα τη διοίκηση ήταν τεκμηριωμένα στον αφορά τη πραγματική ανάγκη του θεσμικού οργάνου. Και επίση υπήρξε μια στρεβλωμένη περιγραφή της κατάστασης, ιδιαίτερα στο Προεδρείο του Κοινοβουλίου τον Ιούνιο στο Στρασβούργο, όπου μόνο ε, μία πλευρά ε, της υπόθεσης, της ιστορίας αυτής, ε, αναφέρθηκε και η πλήρης εικόνα ήταν τελείως ε, διαστρεβλωμένη. Όπως θα δείτε σήμερα, υπάρχουν και πολλά, πολλές αφήσεις στις καμπίνες δερμίας θα τις δείτε γύρω-γύρω. Στο Στρασβούργο είχαμε μαζικές επιτάξεις συναδέλφων, γύρω στο 60% του συνόλου των παρόντων διερμηνέων ε, στο Στρασβούργο μια συγκεκριμένη μέρα, 60% επιτάξεις, είχαμε επιτάξεις ε, καταχρηστικές και αυτή την εβδομάδα. Πολλοί από τους παρόντες συνάδελφους εδώ στην αίθουσα ε, είναι αποτέλεσμα επίταξης και διαμαρτυρόμαστε λοιπόν για την ίδια τη φύση των συνθηκών εργασίας των οποίων, οι οποίες έχουν επιβληθεί. Θα θέλαμε να είμαστε σε θέση να παράσουμε μια υπηρεσία υψηλή ποιότητα, αλλά βεβαίω να διασφαλίσουμε και την προσωπική μα ζωή και την υγεία μα. Να σα αναφέρω ότι ο αριθμό των ωρών που περνάμε καθημερινά είναι στην Καπίνα είναι υψηλότερες, είναι περισσότερες από αντίστοιχου ε, οργανισμούς όπως ο ΙΕ, όπου έχουμε έξι ώρες με τέταρτο, το ένα τέταρτο των γλωσσών που εργάζονται αυτοί σε σχέση με εμά και ήδη βρισκόμαστε εκτός ε, παραδοσιακού ε, εργασιακού ωραρίου επειδή εργαζόμαστε νωρίτερα ή αργότερα. Επίσης θα πρέπει να είμαστε διαθέσιμοι για πολλές μέρες και να έχουμε διαθεσιμότητα για 12 ώρες εργασίας στο Κοινοβούλιο. Και αυτό χωρίς ε, την ε, η διαθεσιμότητά μας, διαθεσιμότητά μας να λαμβάνεται υπόψη στον πραγματικό χρόνο εργασίας, δηλαδή αυτός που παρέχεται προς εσάς. Όλα αυτά δηλαδή οδηγούν σε μεγάλες παρανοήσεις. Δηλαδή ότι εργαζόμαστε μόνο όταν βρισκόμαστε στην ε, καμπίνα. Αυτό είναι το ορατό κομμάτι της δουλειάς μας. Είναι σαν να έλεγα ότι, σαν να ότι οι ευρωβουλευτέ δουλεύουν μόνο όταν πάνε στι ε, συνεδριάσει των επιτροπών. Ε, ο υπόλοιπο χρόνο που βρίσκονται στα γραφεία, που μελετούν τα έγγραφα, που κάνουν πολιτική δουλειά, δεν μετράει. Εδώ πρέπει να πούμε ότι τα δύο τρίτα τη δουλειά μα δεν είναι ορατή, αλλά είναι απαραίτητη ακριβώ για να διασφαλίσουμε την υψηλή ποιότητα εργασία που αξίζετε εσεί και να διασφαλίσουμε την καλή λειτουργία όλου του συστήματο. Δεν θα αναφερθώ τώρα σε λεπτομέρειες που έχουμε εδώ στις διαφάνειες, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αναφέρονται εδώ διάφοροι λόγοι που εξηγούν για ποιο, γιατί είναι διαστερολωμένα τα στοιχεία που παρέχει η διοίκηση του, Ευρωπαϊκού, του Κοινοβουλίου και έχουμε και εδώ μια γραφική απεικόνηση της ε, δουλειά μας. Αυτό είναι το, ένα κλασικό πρόγραμμα, ένα παρουσιακό πρόγραμμα ενός ε, συναδέλφου της καθημερινή του εργασία. Αυτή η συνάδελφο σε συγκεκριμένη περίπτωση ήταν άτυχη γιατί έκανε πάρα πολύ τρει πολλέ τεχνικέ επιτροπέ συν τον τριμερή διάλογο την ίδια εβδομάδα. Οπότε η συνάδελφο θα έπρεπε να προετοιμαστεί εντατικά για αυτέ τι συνεδριάσει. Και αυτό που μετρά στι στατιστικέ είναι η παρουσία, η παραμονή στην ε, καμπίνα ε, όλα τα υπόλοιπα, η προετοιμασία, η εκπαίδευση στις γλώσσες, η καλλιεργία τους κτλ. δεν λαμβάνονται υπόψη. Υπόθηκε λοιπόν ότι οι διερμηνείς αντιστέκονται στις αλλαγές και θέλουν μόνο να συνεχίσουν να εργάζονται όπως εργαζόταν μέχρι τώρα. Αλλά αυτό απέχει πολύ από την πραγματικότητα γιατί όπως βλέπετε από το 2002 έχουμε χάσει 81 θέσεις ε, μελών προσωπικού από 350 σε 269 και έχουν διπλασιαστεί οι γλώσσες. Ε, κάνουμε λοιπόν πολύ περισσότερα με λιγότερα. Επίσης θα έχουμε εξοικονομήσεις με τις αντιπροτάσεις που υπέβαλαν οι διερμηνείς σε σχέση με τις ε, συνθήκες εργασίας. Θα έχουμε περισσότερη ευελιξία χάρη στις καινοτομίε οι οποίες έχουν εισαχθεί και για τις οποίες συμφωνήσαμε ευθύ εξ αρχής ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε περισσότερες συνεδριάσεις ας πούμε κατά διάρκεια των, ε, της ώρας των γευμάτων χωρίς να χρειαστεί να προσληφθούν περισσότεροι διερμηνείς. Επίσης έχουμε και την προσθήκη ε, νέων γλωσσών. Εμείς μελετάμε και μαθαίνουμε συνεχώς νέες γλώσσες. Πολλοί συναδελφοί έχουν 6-7 γλώσσες εργασίας ώστε να έχουμε περισσότερη κάλυψη. Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο και εκπαίδευση. Καταλήγοντας, να πω ότι ήδη έχουμε κάνει πάρα πολλές παραχωρήσεις για να συμβιβαστούμε να βρούμε μια λύση με το Κοινοβούλιο. Αντίστοιχη ανταπόκριση δεν υπήρξε από την διοίκηση. Δεν έχουν αποδεχτεί κανένα από τα κύρια αιτήματά μας και ε, θέλουν την πίτα ολόκληρη για αυτούς έχουν μειώσει τον αριθμό των διερμηνέων, των μονίμων διερμηνέων, θέλουν να μειώσουν και τις προσλήψεις των συναδέλφων freelance, αλλά ταυτόχρονα θέλουν να υπάρχει μια υπηρεσία η οποία θα καλύπτει ένα αυξανόμενο αριθμό συνεδριάσεων. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να τετραγωνίσουμε τον κύκλο και να πετύχουμε τα πάντα χωρίς να λύσουμε δομικά προβλήματα και χωρίς να λύσουμε βέβαια και να ρυθμίσουμε το θέμα των συνδικών εργασίας. Ποια είναι λοιπόν η θέση μας και κατά από το Σεπτέμβριο του 2017 η διοίκηση έχει εφαρμόσει αυτό που λέμε την software, την ήπια εκδοχή των νέων συνδικών εργασίας. Και αυτό ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις αντιπροτάσεις των διερμηνέων. Θεωρούμε λοιπόν ότι ένα συμβασμό μεταξύ των δύο θα μπορούσε να βρεθεί ώστε να εφαρμοστεί αυτή η λύση και να α, γίνει με ταχύ τρόπο θα θέλαμε να βρεθεί μια λύση μάλιστα πριν το καλοκαίρι γιατί έχει τραβήξει πολύ αυτή η ιστορία. Και είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε παραχωρήσεις. Είδαμε ας πούμε στην ε, μικρή Ολομέλεια εδώ στις Βρυξέλλες το Μάγιο ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε πέραν αυτών που προβλέπει το κείμενο των συνθηκών εργασία αν απαιτείται από τις συνθήκες. Βεβαίω, δεν θέλουμε περισσότερα χρήματα, μας ικανοποιούν οι απολαβές μας, όπω και το πολύ προσωπικό εδώ στο Κοινοβούλιο. Θέλουμε απλά και μόνο να βελτιώσουμε τι ειδικέ εργασίε μα. Γιατί θέλουμε να παρέχουμε άριστη ε, ποιότητα ε, η υπηρεσία και να διασφαλίσουμε την υγεία και την προσωπική μα ζωή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή που πραγματικά νομίζω μας ε, ε, έδωσε πολλά στοιχεία παρότι ήταν πολύ περιορισμένος ο χρόνος αλλά νομίζω ότι μάθαμε πολλά και τώρα θα ήθελα να δώσω ε, το λόγο στους συναδέλφους κανένα δύο λεπτά ο καθένας για να μπορέσουν να μιλήσουν όλοι για... Α, με συγχωρείτε, Νόμιζα ότι είχαμε ολοκληρώσει με την παρουσίαση των Δήμων. Ναι, ε, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας παρουσιάζω εγώ την ε, προοπτική των συναδέλφων ε, freelance. Πρόεδρε, θα σας παρακαλέσω να είστε πολύ σύντομοι γιατί νομίζω ότι είναι πραγματικά σημαντικό να ακούσετε και τις, ε, ε, την αντίδραση των συναδέλφων μου βολευτών. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Ε, ο Ρομπέρτο παρουσίασε πολύ καλά την κατάσταση για τις συνθήκες εργασίας. εγώ θα ήθελα να σας δώσω όσο την προοπτική των freelance συναδέλφων. Όταν μιλάμε για συνδίκε εργασία των ε, διερμηνών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, κανεί σκέφτεται του μονίμου που είναι 269. Όμω ε, το Κοινοβούλιο κάθε χρόνο δίνει συμβάσει σε 1.500 freelance διερμηνεί, οι οποίοι καλύπτουν πάνω από το 50% των ορών διερμηνία. Και αυτέ οι συνθήκε εργασία για τι οποίε μιλάμε θα εφαρμόζονται σε όλου αυτού του εργαζόμενου που οι περισσότεροι είναι αυτοαπασχολούμενοι οι freelance που λέγονται AIS που σημαίνει ε, διερμηνής συνεδρίων ε, είμαστε αυτόνομοι εργαζόμενοι με μεγάλα πολλά προσόντα έχουμε περάσει ε, πολύ απαιτητικές εξετάσεις καλύπτουμε όλες τις επίσημες γλώσσες και παρέχουμε απόλυτη ευελιξία και μας εκπροσωπεί η ΑΕΚ η μεγαλύτερη και παλαιότερη επαγγελματική Διεθνής Ένωση Διερμηνέων Συνεδρίων από το 1969 τα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μια σύμβαση με την ΑΕΚ που ρυθμίζει του ειδικού όρου εργασία των freelance συναδέλφων με βασικό όρο και αρχή την ισότιμη μεταχείριση. Όμω οι συνδίκε εργασίε που επιβλήθηκαν πέρυσι ε, δεν τηρούν αυτή την αρχή τη ισότητα. Ε, στο παράρτημα αυτών των συνδικών εργασία υπάρχουν εξαιρέσει για του freelance ό,τι αφορά αντισταθμιστική αποζημίωση για νυχτερινή εργασία ή πάρα πολύ κουραστικές αποστολές. Οι συγκεκριμένες αυτές ε, υποχρεώσεις ε, δεν ε, είναι προσαρμοσμένες ε, στη, στην ιδιαίτερη κατάσταση των freelance γιατί αφήνουν τους freelance χωρίς προστασία όταν ξέρουμε ότι τους προσλαμβάνει το Κοινοβούλιο για μία ή τρεις ημέρες και επομένως δεν μπορούν να, έχουν, να απολαμβάνουν όλων των άλλων διατάξεων για αντιστάθμιση. Ούτε λαμβάνεται υπόψη ο ειδικός χαρακτήρας του επαγγέλματός μας. Επίσης υπάρχει μια δεσπόζουσα θέση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στον αγορά, στην αγορά της διερμηνίας. Ε, επειδή υπάρχει πραγματικά μεγάλος όγκος προσλήψεων και ο βασικός στόχος των συνδικών εργασιών που επευλήθησαν ήταν να μειώσουν το κόστος. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα στερήσει αυτό τη δουλειά από πολλούς από εμάς. Η μείωση του κόστος μπορεί να είναι ένας θεμητός στόχος, αλλά όχι σε βάρος ε, είτε της ποιότητας είτε του απαιτούμενου χρόνου προετοιμασίας. Πρέπει να το ξέρετε αυτό ε, και θα σας το πω. Πολλές φορές πολλοί freelance προσλαμβάνονται 24 ώρες ή και λιγότερο πριν από την έναρξη τη συνεδρίασή του. Και αυτό ασκεί τεράστια πίεση και για την επαγγελματική ποιότητα, καθότι δεν είναι δυνατόν να προετοιμαστούμε καλά, αλλά και για την εργασιακή αξιοπρέπεια δημιουργείται όλο και πιο επισφαλή κατάσταση ε, και θέση εργασία για τους, ε, κατάσταση για του freelance. Αυτό που θέλω να πω όμω ε, όμως είναι ότι υπερβαίνει πολύ αυτό που γίνεται εδώ και το θεσμό αυτό και τους διερμηνείς του Κοινοβουλίου γιατί είναι σημείο αναφορά στι συνθήκε εργασία εδώ για πολλού freelance. Δεν θα πρέπει όμω να μα διαφύγει το βασικό ότι η διερμηνία είναι ένα επάγγελμα κυρίω για αυτοαπασχολήμου και όχι για μονίμου. Οι freelance διερμηνεί και κυριοποίοι ασκούν προσπίζοντας προασπίζονται αυτό το επάγγελμα σε κάθε γωνία τη Ευρώπη ε, έχουν στραμμένο το βλέμμα του εδώ. Εξαρτώνται από αυτό που θα συμβεί εδώ. Και ελπίζουμε να ε, μην προκύψει από όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ κάτι που θα αποτελέσει σκληρό πλήγμα για του freelance συναδέλφου. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν θα δώσω το λόγο στις διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Για το ΕΛΚ παρακαλώ έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Κλόντ. Δεν θα ήθελα εδώ να μιλήσω για τις πολύ μεγάλες ε, προκλήσεις ε, και για την γνώση που απαιτείται για τους διερμηνείς. Νομίζω το γνωρίζουμε εμείς ε, από την εμπειρία μας ως ευρωβουλευτές που συμμετέχουμε στις διάφορες επιτροπές και πραγματικά κάθε μέρα εκτιμούμε τη δουλειά των διερμηνέων. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, νομίζω ότι πράγματι είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και αυτό ε, είναι ένα θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει και τους αντιπροσώπους των δεδομένων αλλά και τα συνδικάτα. Ε, και το βασικό που μας απασχολεί εμάς είναι ο κοινωνικός διάλογος, πραγματικός κοινωνικός διάλογος που δεν υπάρχει και με λυπεί ιδιαίτερα πραγματικά το ότι εδώ στο Κοινοβούλιο μπορεί να δακτυλοδεικτούμε πάρα πολύ εύκολα άλλους επιχειρήσεις ε, που δεν τηρούν τις συνθήκες του κοινωνικού διαλόγου αλλά εμείς εμείς δεν μπορούμε εδώ στο Κοινοβούλιο να φέρουμε σε πέρας ε, πραγματικά ένα σωστό κοινωνικό διάλογο και το είπαν και εκπρόσωποι των διερμηνέων ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη απόκληση, η λύση είναι κοντά και νομίζω ότι μπορεί κανείς ε, να βρει ε, τη λύση πριν τις θερινές διακοπές στο πλαίσιο ενός διαλόγου ε, και σίγουρα ο στόχος είναι να καταλάβουμε ότι εδώ πρόκειται για μια παροχή υπηρεσιών. Το είπαν οι εκπρόσωποι των διερμηνέων, το δείχνουν κάθε μέρα πόσο ευέλικτοι είναι, πόσο προσαρμόζονται και πραγματικά νομίζω ότι το συντομότερο δυνατό θα πρέπει να βρεθεί ο δρόμος πίσω στον κοινωνικό διάλογο και να λυθεί το πρόβλημα πρόβλημα πριν τι euh, Ευχαριστώ, ο κύριος Μαρτάν, για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και του διερμηνείς για τις εξηγήσεις τους. Ήδη εν μέρη τα γνωρίζαμε αυτά. Εγώ διάβασα το φυλαδιό σας αυτό που θέλω να καταγγείλω είναι η στάση του Γενικού Γραμματέα, γιατί διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ένα δικαίωμα οποιαδήποτε επιχείρηση. Όμω, οποιαδήποτε επιχείρηση ε, μπορώ να σα το ότι ε, θα είχε μπλοκαριστεί ε, ουσιαστικά η λειτουργία τη επιχείρηση από την ε, απεργία. Όμω, εδώ έχουμε επίταξη. Πράγματι, πραγματικά στους ε, αντίποδες των δικών μας ε, αξιών ε, και ε, αυτό που συμβαίνει αντίκειται σε όλες τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας και εμείς ε, πώς ε, μπορούμε να το δεχτούμε αυτό και δείτε ότι είναι, μας λένε δείτε είναι άρρωστοι, δείτε πόσο φωνάζουν και πρέπει να τους εγκαταστήσουμε από ποιους από τους freelance και τελικά είναι σαν να έχουμε μιας χρήσης προϊόντα, τα παίρνουμε και τα πετάμε και πάντοτε έλεγα ότι η αξιοπιστία ενός εκλεγμένου είναι να εφαρμόζει για τον εαυτό του αυτά ε, που κηρύττει στους υπόλοιπους. Νομίζω ότι κανένας βουλευτής εδώ δεν θα διχόταν ε, τις ίδιες συνθήκες. Ε, θα πρέπει να το καταγγείλουμε αυτό, αλλά δεν αρκεί πια. Γιατί εγώ ε, πράγματι εξεπλάγει από το γεγονός της επίταξης. Ε, δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό και μαζί σας και μαζί τους εγώ θα εξετάσω τη δυνατότητα να κάνουμε μια ευρεία δράση που θα είναι δυναμική και ορατή και προς τα έξω και να καταγγείλουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ε, το Δεκέμβριο στο Γκέντεμπουργκ είχαμε τρεις υπογραφές από τρεις προέδρους, τους Κιούνκερ και Ταγιάννη, και το μελάνι τη υπογραφή του δεν έχει στεγνώσει ακόμη για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα ε, και τώρα έρχονται και αρνούνται τον κοινωνικό διάλογο. Αυτό πρέπει να το καταδικάσουμε. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι δεν είναι κανείς εδώ από το ΣΥΑΡ και από το ΑΛΔΕ. Η κυρία Κάρη για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους διαρμηνείς για την παρουσίασή τους και σας ευχαριστώ για την καθημερινή σας εργασία. Πράγματι όλοι συμφωνούμε, οι περισσότεροι από εμά αναγνωρίζουν ότι είναι πολύ δύσκολη η δουλειά σας, σε δύσκολες συνθήκες. Χαίρομαι λοιπόν που έμαθα πράγματα σήμερα. Η δική μου ομάδα, όπως και άλλοι, ανησυχούν και έχουν εξοργιστεί από τη στάση ε, του Γενικού Γραμματέα. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες, όμως έχετε δίκιο να ζητάτε να γίνουν σοβαρές κοινωνικές διαπραγματεύσεις. Ε, θα πρέπει η διοίκηση να μπει σε διαπραγματεύσεις και κατά προτίμηση πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Δεν μπορούμε να δεκτούμε αυτό από την πλευρά της διοίκησης και όπως και άλλες ομάδες και εμείς συμφωνούμε να πιέσουμε για να καταγγείλουμε αυτή τη στάση των ευρωπαϊκών οργάνων, αυτού του ευρωπαϊκού οργάνου. Αν ε, δεν υπάρχει κάποιος για τους πρασίνους και τη ο κύριος Μαρτέν για το ΙΕΝΕΦ. Ευχαριστώ. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ απλό. Είναι η έκφραση μιας άκρος φιλελεύθερης Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που με κάθε κόστος ε, θέλει να καταστήσει επισφαλή όλο τον κόσμο. Βλέπουμε μια απλή διαδικασία, αυξάνουμε τον αριθμό των freelance. Από ό,τι κατάλαβα, άνθρωποι που εργάζονται χωρίς πραγματική προστασία και ταυτόχρονα ασκούμε πίεση ε, στους μόνιμους υπαλλήλους και τους ε, επιβάλλουμε όλο ένα και πιο δύσκολες συνθήκες εργασίας και τους οδηγούμε στην ε, παρέτηση για να κάνει οικονομίες ε, ο κύριος Βέλεξ, οικονόμηση. Όμως είναι ντροπή για αυτό το θεσμικό όργανο που πρέπει να δίνει το παράδειγμα και σε όλες τις ομιλίες του λέει εντελώ το αντίθετο ενώ καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια άκρος φιλελεύθερη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που κάνει με τους διερμηνείς είναι η ίδια στρατηγική που με τους λαούς ε, πάντοτε ε, ωφελώντας έναν ακραίο φιλελευθερισμό, υπερβολική επισφάλεια, ε, ευελισφάλεια. Ε, ουσιαστικά αυτό χρησιμοποιείται και εντός του οίκου μας. Ε, είναι κάτι ντυροπιαστικό. Μάλιστα, δώσαμε το λόγο στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Η κυρία Ριμπέιρο, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους διερμηνείς ε, για όλη τη δουλειά και για την ποιότητα της δουλειάς τους ε, τώρα για αυτό το θέμα. Θέλω να θέσω δύο ζητήματα. Το ένα έχει να κάνει με τον κοινωνικό διάλογο Νομίζω ότι εμείς ε, έχουμε επαναλάβει ότι πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη δράση και αυτή η Επιτροπή έχει αυξημένη ε, ουσιαστικά αρμοδιότητα να ζητήσει να αναλυφθεί δράση έτσι ώστε οι υπηρεσίες επικοινωνίας του Κοινοβουλίου να μας πούν τι έχουν κάνει για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια σε αυτή τη διαδικασία πώς διαχειρίστηκε όλο το χρονοδιάγραμμα και ποιες ε, είναι οι προοπτικές της ίδιας της Γενικής Διεύθυνσης για να λυθεί αυτή η υπόθεση στο μέλλον. Και από την άλλη, ε, σε ό,τι αφορά τώρα την επίταξη που και εγώ θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη γιατί έχουμε δει σε όλες τις συνθήκες εργασίας ε, ε, ουσιαστικά αυτή η Επιτροπή Απασχόληση πρέπει να στραφεί στι αρμόδιε υπηρεσίε του Κοινοβουλίου και να ζητήσει εξηγήσει και να μα γνωστοποιήσουν ποιε ήταν οι διαδικασίε, τι υπήρξε πίσω δηλαδή από αυτή την επίταξη των διερμηνέων που εκ πρώτη όψεω ε, μα ε, φαίνεται παράδειγμα γιατί εδώ δεν μιλάμε για ελάχιστη υπηρεσία. Ελάχιστη υπηρεσία είναι όταν τίθεται θέματα ασφάλεια, άμυνα δεν ε, είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ουσιαστικά ε, δεν έχει τέτοιες, χρειάζεται τέτοιες ελάχιστες υπηρεσίες. Έτσι λοιπόν να ζητήσουμε τις εξηγήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες γιατί να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε μία ξεκάθαρη και κάθετη θέση κατά της δράσης αυτής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ ότι όλοι οι συνάδελφοι που στηρίζουν την απεργία και στηρίζουν τους εργαζόμενους ε, διαρμηνείς και στο Κοινοβούλιο και γενικά σαν ειδικότητα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό η υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία να τηρείται σε όλες οι υπηρεσίε και σε όλες τις ειδικότητες του Κοινοβούλιου και στα ευρωπαϊκά όργανα. Γιατί αυτό είναι ο κατρέφτης και αυτό είναι το πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν το χαλάσουμε αυτό, αν δεν το χτίσουμε αυτό, από κάτω οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα παρανομούν πολύ περισσότερο. Γι' αυτό υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. Πολύ σοβαρά θέμα, θέμα το οποίο δεν είναι καλά μελετημένο. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά πάνω σε αυτό. Θα αναφερθώ σε μια μελέτη που είχα, είχα διαβάσει πριν κάποιο καιρό που λέει ότι οι διερμηνείς η στιγμή της εργασίας του ο εγκέφαλός τους παρουσιάζει κατάσταση όμοια με την κατάσταση ένα εγκεφαλικού. Τόση επιβάρυνση έχει ο εγκέφαλός του. Αυτό πρέπει να μας βάζει και να σκεφτούμε λίγο πέρα από αυτό. Τι ζητάμε εμείς, εργασία ή πρέπει να τους οδηγήσουμε σε εξαντλήωση αρρώστιες και καταστροφή του ζωής. Νομίζω ότι όλες οι οργανώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι πρότυπα. Πρέπει να τηρούν όλες, όλα τα δικαιώματα και να προστατεύουν τους εργαζόμενους 100% ειδικά αυτές τις ειδικότητες που είναι τόσο δύσκολες και απαιτητικές. Και ρωτώ τους εισηγητές, οι αλλαγές που προτείνει ο Γενικός Γραμματέας το Ευρωκοινοβούλιο βασίζεται σε κάποια ατρική μελέτη που επιβεβαιώνει, επιβεβαιώνει πως η υγεία σας δεν τίθεται σε κίνδυνο. Διότι οι κανόνες εργασίας σας έχουν βασιστεί στις φυσικές δυνατότητες λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου. Δεύτερη ερώτηση. Πού κωδικοποιούνται οι νέοι κανόνες που εισηγείται ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωκοινοβούλιο Από πού φαίνεται αν οι κανόνες σέβονται τα διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα για την εργασία σας. Και τρίτη ερώτηση, αλητεύει πως δεν θα λάβετε μέρος στις προσεχείς διαπραγματεύσεις για την αλλαγή των εργασιακών σας συνθήκων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Κορούσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που οργανώσατε αυτή τη συνεδρίαση εδώ και πολλούς μήνες. Είδαμε το μήνυμα των διερμηνέων ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τις συνθήκες εργασίας και η δική μας Επιτροπή, αν και δεν συμμετέχει στη συζήτηση, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό όλοι οι βουλευτές να γνωρίζουν ξεκάθαρα ποια είναι η κατάσταση και περί τίνος πρόκειται. Δεν έχω καμία αμφιβολία γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο που θέλει να αλλάξει τον κόσμο αυτό που κάνει είναι να απευθύνει μία έκκληση στα κράτη-μέλη Και εμείς ε, τελικά ε, ουσιαστικά δεν δίνουμε το καλό παράδειγμα εμείς που θα έπρεπε να κάνουμε κάθε στιγμή, θα έπρεπε να δίνουμε το παράδειγμα ανα πάσα στιγμή και να δρούμε έτσι όπως ε, θα οφείλουμε. Χαίρομαι που υλοποιείται αυτή η συζήτηση. Είμαι πεπισμένη ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη και απαιτητική η δουλειά των διερμηνέων και οι συνθήκες εργασίας των διερμηνέων θα πρέπει να γίνονται σεβαστές επειδή είναι πολύ δύσκολη ακριβώς αυτή η δουλειά ε, το πώς ε, κάνουν διερμηνείς έχει επίπτωση και στο πώς μπορούμε να εργαστούμε εμείς ως βουλευτές μεταξύ των ε, διερμηνέων που εργάζονται στο Κοινοβούλιο υπάρχουν ε, πολλά κοινά στοιχεία. Δεν είναι μόνο οι διερμηνείς, ε, υπάρχουν πέρα από τους διερμηνείς και οι βουλευτές, αλλά και οι υπάλληλοι που πρέπει να εργάζονται με ένα πολύ γρήγορο ρυθμό. Πρέπει να δουλεύουμε μάλιστα και τη νύχτα. Αυτό μας επηρεάζει όλους. Και αν ε, υπάρχουν ε, κάποια ερωτηματικά. Εγώ νομίζω ότι αυτές οι αμφιβολίες θα πρέπει να απαντηθούν ευρύτερα και όχι μόνο σε σχέση με τους διερμηνείς. Ε, μεταφραστές παραδείγματος χάρη έχουν ε, τρεις εβδομάδες ε, για να μεταφραστούν κείμενο, αλλά εμείς ως βουλευτές ε, έχουμε παραδείγματος χάρη μία μέρα μόνο για να ετοιμάσουμε μία συμβιβαστική τροπολογία που πρέπει να μεταφραστεί στη συνέχεια και αν μιλήσουμε, πρέπει να μιλήσουμε για την οργάνωση των εργασιών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ευρύτερα και συνηθίζουμε να λέμε ότι η Επιτροπή Επασχόλησης είναι αυτή που εκπροσωπεί το τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ δυστυχώς έχω πάρα πολύ λίγα στοιχεία για να αξιολογήσω αυτό το διάλογο που έγινε μεταξύ της διοίκηση και των διερμηνέων. Ξέρω ότι τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια είχαμε δεκάδες συνεδριάσεις. Ε, το πορκέ αυτές οι συνεδριάσεις δεν μπορούν να ε, ονομαστούν κοινωνικό διάλογο. Είναι μια ερώτηση που πρέπει να θέσουμε, όμως ε, έγιναν αυτές οι συνεδριάσεις. Εμένα αυτό που μου λείπει είναι και το πώς βλέπει το θέμα η άλλη πλευρά. Θα ήθελα να ακούσω και την άλλη πλευρά, γιατί σε ένα κοινωνικό διάλογο συμμετέχουν δύο. Τώρα ακούμε μόνο το πώς το βλέπει μία πλευρά. Αυτό που λέτε μου φαίνεται ότι είναι ρεαλιστικό αλλά θα αισθανόμουν καλύτερα αν σε αυτή την ίδια συνεδρίαση θα μπορούσα να ακούσω και τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς για να μπορώ να συγκρίνω τα δύο επιχειρήματα. Ελπίζω ότι όλο αυτό θα μας χρησιμεύσει για να κατανοήσουμε πολύ καλύτερα αυτή την διαμάχη. Γιατί εμείς δεν είμαστε μέρος, δεν θα έπρεπε να είμαστε μέρος, καθώς δεν είναι η δική μας επιτροπή που ουσιαστικά προσλαμβάνει τους διερμηνείς. Εμείς Χρησιμοποιούμε τι υπηρεσίες σα, αλλά δεν σας προσλαμβάνουμε. Ελπίζουμε στο εγγύς μέλλον να μπορέσουμε να λάβουμε πιο πλήρες πληροφορίες για να μπορούμε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη και δίκαιη αξιολόγηση για να μπορέσει να βοηθήσει τον αγώνα σας. Σας ευχαριστώ. Έδωσα το λόγο λοιπόν στους διάφορους συναδέλφους που μου το είχαν συζητήσει και ως πρόεδρος της Επιτροπής ε, δεν θα φτάσω ένα συμπέρασμα τώρα γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς. Ε, ελπίζω να μπορέσει να υπάρξει στο τέλος ε, μια συμφωνία, να καλυφθούν τα αιτήματά σας και να υπάρχει πραγματικός κοινωνικός διάλογος. Όμως ε, μας ακούσατε, είμαστε αλληλεγγύοι με, δύο, με τις δύο έννοιες της λέξης. Όταν λέω με τις δύο έννοιες, καταρχήν υπάρχει η αλληλεγγύη της βούλησης, ε, δηλαδή ότι ακούμε τις διεκδικήσεις σας, ότι ε, ακούμε ότι υπάρχει έλλειψη ε, της διαδικασίας κοινωνικού διαλόγου, όμως είμαστε αλληλέγγυοι και με υλικό τρόπο ουσιαστικά με σωματικό τρόπο θα έλεγα. Χωρίς να είναι αρνητικό αυτό, μην με παρεξηγήσετε, αλλά ως ε, διερμηνείς είστε ένα μέρος από εμά. Αναφέρετε τις δικές σας συνθήκες εργασίας. Αυτές οι συνθήκες εργασίας οι δικές σας ε, σχετίζονται με τον τρόπο που εργαζόμαστε κι εμείς. Ε, χωρίς εσάς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κατά κάποιο τρόπο είστε η φωνή μας, ακόμη και δεν μπορείτε να αναπαράξετε τη φωνή μας, αλλά πρέπει να τη μεταφράσετε. Δεν ε, νομίζω ότι πρέπει να ε, εφησυχαστούμε στο να σας ακούμε απλώς, το να σας ακούμε. Ε, ναι, είναι τώρα και φυσικά θα ακούσουμε και τη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει και μια σειρά εγγράφων, όμως δεν έχω πρόβλημα στη συνεδρία των συντονιστών να αναφερθούμε σε αυτό το θέμα, να ακούσουμε και τη διοίκηση, γιατί το υποχρεώνει ο κοινωνικός διάλογος να έχουμε δύο μέρη που συνομιλούν, αν και δεν είμαστε εμείς ε, ένα από τα δύο αυτά μέρη. Και νομίζω ότι δεν ε, μπορούμε να μείνουμε σε αυτό. Θα σας πρότεινα, αν συμφωνείτε, τουλάχιστον ε, θα το παραπέμψω αυτό και στην συνεδρία των συντονιστών, αλλά νομίζω αφενός ότι από την Επιτροπή Απασχόλησης, αν και δεν αφορά μόνο αυτή την Επιτροπή, να απευθυνθούμε επίσημα και στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στη Γενική Διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και στους Προέδρους των διάφορων πολιτικών ομάδων, καθώς συμμετέχουν ε, στην διάσκεψη των Προέδρων και ε, όχι για να μπούμε στις διαπραγματεύσεις, δεν είναι ο δικός μας ρόλος, αλλά για να δηλώσουμε την λύπη μας για την κατάσταση αυτή. Και λυπούμαστε για αυτήν την κατάσταση γιατί μας εμποδίζει να λειτουργήσουμε σωστά, να ασκήσουμε τα καθήκοντα του βουλευτή. Είναι μια κατάσταση που εμποδίζει τη δημοκρατία να λειτουργήσει. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Από την άλλη, να επενθυμίσουμε τις αρχές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αναφερθήκατε ε, και στις αρχές αυτές και συνυπογράφησαν από τα τρία θεσμικά όργανα ε, μέσω του κοινωνικού πυλώνα, γιατί σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση, σε κάθε έκθεση και σήμερα το πρωί μάλιστα, νομίζω δεν υπήρξε κανένας ε, φάκελος που να μην αναφερθήκαμε στο θέμα του κοινωνικού διαλόγου. και επίσης ε, να δηλώσουμε την ενισχύα μας ε, κατά της αρχής της επίταξης, να ρωτήσουμε το γιατί. Ε, η ενδεχόμενη νομική βάση μπορεί να υπάρχει. Εσείς αναφερθήκατε στους ευρωπαϊκούς καλώνες, αλλά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και τις βασικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που πλαισιώνουν το δικαίωμα στην απεργία και υπάρχουν κάποιε δυνατότητε να προβλέπονται και συστήματα επίταξη. Και ακόμη και αν στα διάφορα κράτη-μέλη υπάρχουν διαφορετικοί κανόνε, εδώ ε, υπάρχουν ε, κάποια πράγματα που μπορεί να ε, διατηρούν πριν το σχάρι, κάποια στοιχεία, κάποιες εργασίες που αφορούν την ασφάλεια, την άμυνα κτλ. Επίσης, αναφερθήκε και συνάδελφος στο εξή, ε, στο ποια θα είναι ε, η πορεία της λήψης ε, αποφάσεων. Επίσης, να πούμε ξεκάθαρα ως Επιτροπή Επασχόλησης τι θέλουμε, απαιτούμε να υπάρχει σοβαρή επανέναρξη της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης και διαβούλευσης. Με όλη τι σημαίνει αυτό. Εμείς δεν Είμαστε ουσιαστικά εδώ για να ε, αναφέρουμε τις δικές σας ε, απαιτήσει, τις δικές σας διεκδικήσεις, όμως αυτό είναι δική σας δουλειά, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός απέναντι στο δικό μας θεσμικό όργανο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ αντικαθιστώ τη Μαρίτα και θα τα μεταφέρω όλα αυτά στους συντονιστές για να μπορέσουμε να τα κάνουμε πολύ γρήγορα. Και κάτι τελευταίο. Βγαίνω από το ρόλο του Πρόεδρου. Νομίζω ότι ο Έντουαρτ το ανέφερε. Να δούμε τι άλλα είδη δράσεις θα μπορούσαμε να έχουμε. Αλλά αυτό δεν το λέω ως πρόεδρος αυτής της Επιτροπής. Ξέρετε ότι μια σειρά βουλευτών είναι διαθετημένοι να σας στηρίξουν, είναι δική τους επιλογή. Έτσι λοιπόν, αν το επιθυμείτε, σας καλώ να έρθετε σε επαφή μαζί τους και πάντοτε, όχι ως πρόεδρος, ε, λέω ότι υπάρχουν ε, και άλλα θέματα στα οποία ζητάμε ε, την διαβούλευση. Μάλιστα, στο Στρασβούργο ε, πολλές φορές έχουμε κάποιους συμβασιούχους που δεν την χάνουν ορθής μεταχείρισης. Εγώ ήμουν συνδικαλιστής ε, όλη μου τη ζωή και θεωρώ ότι μία επιχείρηση, όποια και να είναι, θα πρέπει να αλλάζει και να προσαρμόζεται σε μία σειρά καταστάσεων και μάλιστα και με μερικές δυσάρεστες εξελίξεις όμως ε, αυτό θα πρέπει να γίνεται με απόλυτο σεβασμό και με την απαραίτητη διαβούλευση και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι μπορούμε να μείνουμε εδώ και είμαι και στη διάθεσή σας. Ε, ε, αν θέλετε να συνομιλήσετε με τους συναδέλφους για να σας βοηθήσουν έτσι ώστε να λαδοθεί κάπως ο μηχανισμός και να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει, μπορείτε να το κάνετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους βουλευτές που πήραν ε, το λόγο. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ζητώ την ε, ανοχή και από τους συνοδέλφους. Για μια φορά δεν θα σταματήσουν στην ακριβή ώρα. Για να απαντήσω στις ερωτήσεις. Δεν θα πω ότι συμφωνώ με το 99% των όσων είπατε σε ό,τι αφορά τη φύση του κοινωνικού διαλόγου μας ρωτήσατε πώς και δεν υπήρχε κοινωνικός διάλογος αν έγιναν τόσες συνεδριάσεις ε, εδώ. Ε, έχουμε ζητήσει και τη γνώμη των νομικών μα. Ένα πραγματικό κοινωνικό διάλογο είναι ότι και τα δύο μέρη μπορούν να ασκήσουν μία επιρροή στο αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή, στο κείμενο για τι συνθήκε εργασία είχαμε πολλέ συνεδριάσει, είναι αλήθεια. Όμω οι διερμηνεί δεν είχαν τη δυνατότητα να ακουστούν σε, καμία, σε κανένα από τα σημαντικά αιτήματά τους. Δεν ε, μιλάμε δηλαδή μόνο για απλή φυσική παρουσία σε μία αίθουσα, αλλά ζητάμε να ληφθούν ε, και υπόψη οι απαιτήσει του άλλου μέρους. Σε ό,τι αφορά τώρα τις επιτάξεις. είναι ξεκαθαρό ότι χρειάζεται μια ισορροπία μεταξύ του δικαιώματο ε, στην απεργία και τη απέτηση ε, των απαιτήσεων του θεσμού. Όμω ε, αυτή η απέτηση, δηλαδή να υπάρχει μια ελάχιστη υπηρεσία που να εγγυάται και το δικαίωμα στην απεργία. Οι επιτάξει όπω έγιναν την περασμένη αλλά και αυτή την εβδομάδα δεν εγγυούνται το δικαίωμα στην απεργία. Επομένω, ο πύχη ήταν πολύ κοντά στι απαιτήσει ε, του θεσμικού οργάνου και πολύ μακριά από το δικαίωμα τη απεργία και ε, αυτό φυσικά παραβιάζει και όλε τι διεθνεί συμβάσει που αναφέρατε. Και συγκεκριμένα χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια. Δεν έχουμε πρόσβαση σε ουσιαστικά δεδομένα που μας δείχνουν τι ακριβώ είναι απαραίτητο για αυτό το θεσμικό όργανο. Πάντοτε μας τα έχουν αρνηθεί. Η διοίκηση δεν ε, εκφράζεται εδώ, είναι αλήθεια σε αυτή τη συνεδρίαση, όμω έχει πολύ πιο εύκολη πρόσβαση στους βουλευτές. Ε, μάλιστα στους βουλευτές μοιράστηκε και μια παρουσίαση που όπως σα είπα παρουσιάζει μια ε, πολύ ανακριβή εικόνα της πραγματικότητα και πιστεύω λοιπόν ότι η διοίκηση είχε τη δυνατότητα να εκφραστεί επαρκώς. Είναι αλήθεια ότι οι δραστηριότητε μα είναι πολύ συγκεκριμένοι, πολύ ιδιαίτεροι, όπως είπε και η κυρία Κούνεβα, και γι' αυτό ε, οι ίδιες ώρες εργασίας έχουν διαφορετικό αντίκτυπο ανάλογα με τη δραστηριότητα. Στη διερμηνία ο αντίκτυπος είναι πολύ μεγαλύτερος σε ό,τι αφορά τις επόμενες διαπραγματεύσεις, ε, ρωτήθηκα αν θα συμμετέχουν οι διερμηνείς. Ε, η πρότυπη διαδικασία προβλέπει τη συμμετοχή διερμηνέων, όμως από πέρσι τον Νοέμβριο οι διερμηνείς έχουν αποκλειστεί από τις διαπραγματεύσεις. Εκπροσωπούνται από την Επιτροπή Προσωπικού, δεν είμαστε πλέον ε, άμεσα παρόντες στο τραπέζι τη διαπραγμάτευση. Ζητάμε να επιστρέψουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ζητάμε πολιτική παρέμβαση, πολιτική διαμεσολάβηση σε αυτό το σημείο, γιατί δεν κατορθώνουμε να, φέρνουμε, ε, να φέρουμε κοντά τι θέσει λόγω τη άκαμπτη ε, θέση τη διοίκηση. Ε, όπω σα είπα, υπάρχει μεγάλο αντίκτυπο, εμεί εργαζόμαστε άσχημα και ακόμη χειρότερα εσεί. Και όλοι όσοι σα ακούν και εκτό από εδώ, καταλαβαίνουν, δεν καταλαβαίνουν όπω πρέπει. Δεν μιλούν όλοι τόσε γλώσσε. Αν εμεί δεν μεταφράζουμε καλά, δεν θα καταλάβουν και αυτό ε, ουσιαστικά δεν εξυπηρετεί το να έρθει το θεσμικό όργανο κοντά στου πολίτε, ε, που πιστεύω είναι και δικό σα στόχο. Ε, και <laughs> με ε, αυτό που αναφέρατε, το σωματικό δεν βρίσκω κανένα λόγο προσβολή. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ελληνική και σας ευχαριστούμε και για τις πρωτοβουλίες σας. Να απευθυνθείτε απευθεία στον Πρόεδρο, στο Γενικό Γραμματέα και στις πολιτικές ομάδες. Γιατί, επαναλαμβάνω, αν υπάρχει πολιτική βούληση μπορεί να βρεθεί η λύση. Η δίκηση ήδη έχει αποκτήσει όλα αυτά που ήθελε. Εξοικονόμηση χρημάτων, μεγαλύτερη αποδοτικότητα των πόρων, μεγαλύτερη ευελιξία. Ήδη καλύπτουμε με τις νέες ανάγκες του Κοινοβουλίου. Δεν προσπαθούμε να αποκτήσουμε υπερβολικά. Λέγεται ότι το βέλτιστο είναι εχθρό του καλού. Αν προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε περισσότερα, μπορεί να καταστρέψουμε μια υπηρεσία που πάντοτε ε, ήταν υποδειγματική ε, σε αυτό το κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Je Ολοκληρώνουμε αυτή τη συνεδρίαση. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όσου συνεχίζουν να εργάζονται. Σα ευχαριστώ και για την παρουσία σα στην αίθουσα και να πω δύο λόγια. Δεν έχει περάσει και τόσο πολύ καιρό που διάφορε πολιτικέ ομάδε. Ε, είχαν ε, ε, οργανώσει μία συνάντηση με τον Αλεξάνδρ Κόζεφ. Ε, και αυτός ε, ο Ευρωπαίος φιλόσοφος και διαπραγματευτής που δυστυχώς απεβίωσε έλεγε ότι η διαπραγμάτευση είναι η συνάντηση των επιθυμιών. Έτσι λοιπόν, ας πράξουμε έτσι ώστε να συναντηθούν οι επιθυμίες.